Colleghi, per favore prendete posto, non possiamo aspettare l'arrivo di... Συνάδελφοι, παρακαλώ, καθίστε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε δυστυχώ την άφηξη όλων των συναδέλφων, διότι ο κύριο Σέρζ Μπραμέτ, εισαγγελέα στο διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο, ε, έφτασε εν Η μέρα μα είναι ιδιαίτερα φορτωμένη και παρακαλώ να ξεκινήσουμε ευθύ αμέσω τις εργασίες μας. Με τους λίγους παρόντε, τι να κάνουμε. Έχω την ιδιαίτερη ευχαρίστηση να καλωσορίσω τον κύριο Σέρζ Μπράμετ, εισαγγελέα στο διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Ιουκοσλαβία. Η επίσκεψή σας, δόκτωρα Μπράμετς, επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον μας, το ενδιαφέρον του Κοινοβουλίου, αλλά και της ε, Επιτροπής μας, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, για τις εξελίξεις στα Βαλκάνια. Μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι εξελίξεις ε, και η πρόοδος που επετεύχθη σε ζητήματα συνεργασίας ε, του, Ευρωπαϊ... του Διεθνούς Ποινικού δικαστηρίου με τις ε, τρεις ενδιαφέρουμενες χώρες, ε, Βία, Κροατία και Βοσνία Ριζεγοβίνη. Εξ ονόματος λοιπόν όλων των συναδέλφων θα ήθελα να επιβεβαιώσω πόσο ισχυρή είναι η υποστήριξή μας προς το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Δίχως δικαιοσύνη δεν μπορεί να υπάρξει συμφιλίωση ανάμεσα στους λαούς και τις εθνότητες που έζησαν αυτή την τραγική κατάσταση και αυτό τον αιματηρότατο πόλεμο, λοιπόν χωρίς συμφιλίωση, που είναι και το προήμιο για κάθε πρόοδο, δεν μπορούμε να θέσουμε σε ενέργεια το διαδικασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κοινότητές μας, η κοινότητά μας είναι μια κοινότητα ε, συμφερόντων αλλά και αρχών τις οποίες ε, συμμεριζόμεθα όλοι. Η συνεργασία με το δικαστήριο φυσικά αποτελεί μια βασική προϋπόθεση η οποία θα πρέπει να πληρωθεί. Είναι η προκατακτική προϋπόθεση για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις λόγω χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ε, αναφέραμε πάντα στο παρελθόν εξάλλου όταν εξετάσαμε αυτό το ζήτημα. Στις 13 ε, Δεκεμβρίου εσείς ε, κύριε Σαγγελέα παρουσιάσατε ενώπιον του Συμβουλίου ε, Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών την συνεργασία σας και την συνεργασία σας με τα λογοκράτη Και εσείς καταγράψατε μια σημαντική και σταθερή πρόοδο της κατάστασης στην Σερβία. Η συνεργασία ήταν απόλυτη και εξάλλου η σύλληψη του Ράντοβαν Βανεσάνσης χαιρετίστηκε από την διεθνή κοινότητα ως κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας. Παραμένουν ελεύθεροι ακόμα δύο όπως ο Γκόραν Ράντιτς και ο Ράνκο Μλάντιτς, δύο κατηγορούμενοι για εγκλήματα πολέμου. Αυτοί οι δύο φυγάδες λοιπόν θα πρέπει να συλληφθούν και αυτό αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την Σερβία. Και έχουμε εδώ τις μαρτυρίες ε, των σερβικών αρχών, εσείς ε, το σημειώσατε και αναφέρατε την δέσμευση που έχει αναλάβει η κυβέρνηση προς την κατεύθυνση αυτή. Η έκθεσή σας ήταν πολύ πιο, πολύ πιο αυστηρή σε ό,τι αφορά την Κροατία. Η συνεργασία θεωρήθηκε ότι δεν βρίσκεται στο ύψος των προσδοκιών, αλλά θα πρέπει να πούμε πως η δημοσιότητα η οποία δόθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο στις δηλώσεις αυτές τις δικές σας είχε θετικότατε συνέπειες διότι στην Κροατία αναπτύχθηκε ένα κίνημα και ιδιαίτερα σε κυβερνητικό επίπεδο αυτά τα λόγια σας αξιολογήθηκαν και είχαν θετικές επιπτώσεις τα όσα δηλώσατε στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Σε ό,τι αφορά το τη Βοσνία Ριζεγοβίνη, δεν είναι ικανοποιητική η κατάσταση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την συνεργασία, και δει σε ό,τι αφορά τους κινδύνους που αντιμετώπισαν οι μάρτυρες ε, πριν να μεταβούν στο δικαστήριο. βρίσκαν απειλές κλπ. Χρειάζεται λοιπόν ε, να μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι εμπλεκόμενες χώρες δεν έχουν δυνατότητα να κρίνουν και να δικάζουν ε, τις ε, εγκληματίες πολέμου. Αυτό τονίστηκε στην έκθεση ε, της οποίας η ήταν η κυρία Νέιτς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει αυτή τη στρατηγική και υπογραμμίζει την σημασία του να μπορέσει το δικαστήριο να ολοκληρώσει την εντολή του με την ε, δίκη, αφού συλληφθούν φυσικά, οι καταζητούμενοι του των λεχθέντων. Ε, να σας δώσω το λόγο κύριε Ισαγγελέα. Thank you very much, Mr. President. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Καλώς απόγευμα. Ευχαριστώ θερμά που με προσκαλέσατε σε αυτή την ε, συνεδρία σα. Με την αδειά σα θα ήθελα να σα δώσω μια σύντομη παρουσίαση τη κατάσταση στην οποία έχουμε σήμερα και βέβαια πάνω απ' όλα να ακούσω τι ερωτήσει σα. Θα ήθελα καταρχά για άλλη μια φορά να υπογραμμίσω την σημασία τη υποστήριξη που έχει προσφέρει ιδιαίτερω η διεθνή κοινότητα και τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω γνωρίζετε, έχουμε τακτικέ επαφέ και συζητήσει με το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με μεγάλη χαρά, βέβαια, είμαι εδώ παρόν σήμερα ενώπιον τη Επιτροπή των Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επί τη ευκαιρία και εκ μέρου ε, του Διεθνού Δικαστηρίου θα ήθελα να σα ευχαριστήσω και για το ψήφισμα του Μαρτίου που αποτέλεσε ε, σαφέστατο μήνυμα στήριξη προ το Διεθνέ Δικαστήριο σε αυτήν την τελική φάση τη ύπαρξή του. Σα είμαστε ευγνώμονε για τη στήριξη που μα προσφέρατε στο παρελθόν, αλλά θα θέλαμε να συνεχιστεί αυτή η στήριξη και στο μέλλον. Και είμαι βέβαιο ότι συμμερίζεστε όλοι τον ίδιο στόχο όπως και εμείς, δηλαδή την ε, απόδοση δικαιοσύνης για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στην, στην πρώην τα, ε, να στηρίξετε τους λαούς στην ε, πορεία τους προς το μέλλον και βεβαίως τη δικαιοσύνη των κρατών αυτών ώστε να είναι πιο αποδοτική και να επιτρέψετε όταν κλείσουν οι πόρτες του δικαστηρίου μας να δοθεί συνέχεια στις δίκες στα κράτη. Όπως γνωρίζετε, πριν από 16 χρόνια που ιδρύθηκε το δικαστήριο, στα πρώτα του βήματα ήταν δύσκολο το έργο των προκατόχων μου. Ήταν δύσκολο να χειριστούν τις υποθέσεις για λόγους επιμελητιακούς, οργανωτικού και βέβαια κύριο πρόβλημα ήταν όπως γνωρίζετε η σύλληψη των φυγάδων γιατί οι πολιτικές αρχές της εποχής δεν έσπευδαν να προσφέρουν χειραβοηθεία στο δικαστήριο. Με χαρά λοιπόν σημειώνουμε τις σημαντικές εκτοτεξελίξεις και Ιδιαίτερος σήμερα καλωσορίζουμε το γεγονός ότι οι πολιτικοί συνομιλητές μας έχουν διαφορετική στάση και ότι λαμβάνεται υπόψη η πολιτική σημασία και ως πολιτική σημασία στο έργο του δικαστηρίου. Έχει μεγάλο ρόλο διαδραματίσει και θα διαδραματίσει το δικαστήριο για την απόδοση της δικαιοσύνης και επίσης στην στήριξη της διαδικασίας ε, για απόδοση δικαιοσύνης σε διεθνές επίπεδο μαζί με άλλα δικαστήρια που ακολουθούν το παράδειγμα του δικού μας. Από την ε, ίδρυση του, του δικαστηρίου απευθύνθηκαν κατηγορίες κατά 161 ατόμων όπως γνωρίζετε, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ε, κατά 121, 86 υποθέσεις δηλαδή και τώρα μας μένουν ακόμα 10 τελευταίες ε, υποθέσεις με 25 κατηγορούμενους. Άλλες εκκρεμίε υποθέσεις δεν έχουμε και έχουμε ακόμη δύο μεγάλους, δύο φυγάδες ε, που ασφαλώς θα σας απασχολήσουν κατά την ώρα των ερωταποκρίσεων, αλλά πάντως η σύλληψη των φυγάδων αυτών, των δύο αυτών φυγάδων, είναι από τις κυρίες μας προτεραιότητες. Όχι μόνο για την περιοχή, για την ειρήνη στην περιοχή, όχι μόνο προτεραιότητα για το δικό μας το δικαστήριο, γιατί ασφαλώς με το που θα συλληφθούν αυτοί οι δύο φυγάδες μπορούμε να ολοκληρώσουμε το έργο και το καθήκον μας, αλλά ταυτόχρονα είναι ζήτημα αξιοπιστίας η σύλληψη των δύο αυτών φυγάδων και για τη διεθνή κοινότητα. γιατί για τη σύλληψη του Μλάντιτς και αντίστοιχων ε, ιδρύθηκε το δικαστήριο και στόχος μας είναι να συλληφθούν. Ξέρετε ότι έχουμε 10 υποθέσεις εκκρεμής όπως σας είπα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ένταση δικαστικού έργου που είχαμε ποτέ στην ιστορία μας και ταυτόχρονα παρακολουθούμε την ολοκλήρωση της στρατηγική, της στρατηγική ολοκλήρησης που ξέρετε ότι είχε αποφασιστεί ότι δεν θα υπάρξουν νέες ε, απαγγελίες κατηγοριών, νέες προσαγωγές στη δικαιοσύνη και έτσι είχαμε πει ότι τις ε, απαγγελίες κατηγοριών μέχρι το 2008 θα τις είχαμε ολοκληρώσει και το 2010 θα είχαμε κλείσει τις δίκες. Δυστυχώς οι προθεσμίες δεν μπόρεσαν να τηρηθούν. Γιατί, γιατί καταρχάς συνελήφθηκαν και ότι κάποιοι από τους φυγάδες και φυσικά έπρεπε να ε, συμπεριληφθούν στις διαδικασίες. Αυτή τη στιγμή με βάση τους υπολογισμούς μας σε πρώτο βαθμό ε, οι δίκε που έχουμε σε πρώτο βαθμό εκκρεμή θα, θα κλείσουν μέχρι το 2011 ίσω ίσως όπως του Κάρατζιτς να πάνε μία-δύο στο 2012 και σε δεύτερο βαθμό πάνε ίσω μέχρι το 2013 με μία ή δύο που θα πάνε μέχρι το 2014. Αυτό είναι το σχέδιο μέχρι στιγμή. Και από το προσεχές καλοκαίρι σκοπεύουμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία τη σταδιακή μείωση των πόρων μας, καταρχάς με τον προϋπολογισμό για τα επόμενα ένα-δύο έτη και επίσης ε, ως προς το προσωπικό για το 2010-2011 από το γραφείο μας θα δούμε από περίπου 60% του προσωπικού μας. Και ένα ζήτημα το οποίο σωστά πρέπει να συστήσουμε αργότερο είναι το θέμα της ε, παρακράτησης προσωπικού, γιατί έχουμε ακόμη ε, σημαντικό ποσοστό, σημαντικό αριθμό υποθέσεων που είναι εκρεμή, ενώ ταυτόχρονα ενημερώνουμε το προσωπικό μα ότι σε λίγο θα πρέπει να κινηθεί σε άλλε θέσει και έτσι αρχίζουν να αναζητούν θέσει εργασία στα ε, ε, Ηνωμένα Έθνη σε άλλε αντίστοιχε υπηρεσίες ε, και σιγά σιγά του βλέπουμε να αποχωρεί το προσωπικό ενώ ακόμα το χρειαζόμαστε γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί αυτέ οι υποθέσει και όπω γνωρίζετε ασφαλώ, πρόκειται για το πιο καλά κατερτισμένο προσωπικό σε τέτοιου είδου διεθνεί ποινικέ υποθέσει. μειώνεται λοιπόν το προσωπικό και οι πόροι μα και πολύ σημαντικό πρόβλημα, ζήτημα θα είναι για το εγγύς μέλλον η συνεργασία, το έχω ήδη υπογραμμίσει, ε, μια από τις κύριες διαφορές μεταξύ του να είναι κανείς εισαγγελέα μέσα σε ένα εθνικό σύστημα δικαίου, όπως ήμουν εγώ τελευταία, τα, τα, επί 15 έτη, και να είναι κανείς μέσα σε ένα διεθνές σύστημα δικαίου. Η κύρια διαφορά λοιπόν είναι ότι όταν είναι κανείς εισαγγελέα διεθνούς δικαστηρίου εξαρτάται απόλυτα από τη διεθνή υποστήριξη. Όποια υποστήριξη του προσφέρεται είναι απαραίτητη, όπως είναι απαραίτητη και σήμερα ακόμη η στήριξη της διεθνούς κοινότητας για τη σύλληψη των φυγάδων, όπως είναι απαραίτητη η στήριξη της διεθνούς κοινότητας για να επιβληθούν κυρώσεις εις βάρος αυτών που υποστηρίζουν ή υποθάλπουν τους ε, φυγάδες και επίσης Θέλουμε την ε, υποστήριξη εθνική κοινότητα και για την εξασφάλιση πρόσβαση σε έγγραφα και αρχεία. Και χρειαζόμαστε και την διεθνή υποστήριξη. για την πρόσβαση στα δεδομένα στις πηγές. Στα πρώτα χρόνια λοιπόν της ύπαρξης του δικαστηρίου μας, ε, οι συλλήψεις των φυγάδων ήταν ένα από τα κύρια μας προβλήματα. Τα τελευταία πέντε χρόνια ευτυχώς βλέπω σημαντική αλλαγή στη συμπεριφορά, στη στάση των κυβερνήσεων της περιοχής και καθιστάται απόλυτα σαφές ότι Εάν, εάν προέκυψε αλλαγή, η αλλαγή οφείλεται βέβαια στην αλλαγή κυβερνήσεων στι νέε κυβερνήσει που έχουν λάβει την εξουσία στην περιοχή, αλλά επίση και στι τάσει τη διεθνού κοινότητα των Ηνωμένων Εθνών, τη Ευρωπαϊκή Ένωση, των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ που έχουν εκφράσει την υποστήριξή του στο δικαστήριο και στην απέτηση για σύλληψη των φυγάδων. Όπω ε, άλλωστε το 2000 με τη διάσκεψη των χορηγών εκφράστηκε απερίφραστα η προπόθεση για τη χορήγηση τη χρηματοδοτική ε, στήριξη με τη σύλληψη των ε, φυγάδων. Και επίσης με την ε, προϋπόθεση που ορίστηκε από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης αμέσως μετά ε, για τη στήριξη στην Σερβία και, της, και, και την Κροατία, τη Βοσνία Σεκοβίνη για την προεταξιακή τους πορεία. Την, η προϋπόθεση αυτή τη συνεργασία με το Εθνικό Δικαστήριο που αποτέλεσε το κυριότερο εργαλείο, το κυριότερο όπλο στα χέρια μας. Μας βοήθησε πάρα πολύ λοιπόν αυτή η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις προποθέσει και τα κίνητρα βέβαια που δημιούργησε ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση στην, στα κράτη τη περιοχής αυτή. Δεν μπορώ να υπογραμμίσω, δεν έχω λόγια να εκφράσω την εγγνωμοσύνη μου για την ε, στήριξη που μα προσφέρατε και την αποτελεσματικότητά σα. Αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με τι ε, κυβερνήσει περιοχή. Ο Πρόεδρο ανέφερε τη συνεργασία με, την, ε, με τη Σερβία, με την Κροατία και με τη Βοσνία. Έχουμε συνεργασία. Ουσιαστικά καινούριο δεν έχω τίποτε να σας αναφέρω από την τελευταία μας έκθεση, τελευταία έκθεση προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του Δεκεμβρίου. Η γραμμή που αποκολουθήσαμε σε σχέση με τη Σερβία, όπως γνωρίζετε, ήταν ότι είμαστε ικανοποιημένοι με τις προσπάθειες από τις προσπάθειές της να μας βοηθήσει στο έργο μας. Έχουμε υπογραμμίσει ότι η συνεργασία είναι συνεργασία ρουτίνας, υποβάλλουμε το αίτημα για, υπο... για αρρωγή και γίνεται αυτή η ανταλλαγή σχεδόν καθημερινά, ανταλλαγή επικοινωνιών. Υπάρχει, ε, υπάρχει η πρόθεση για βοήθεια ως προς την αναζήτηση των φυγάδων ε, που είναι πολύ σημαντική δέσμευση, αλλά ακόμη δεν έχουμε καταλήξει και πρέπει να συνεχιστεί. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας και βέβαια παρακολουθούμε και εμείς και ε, συμβάλλουμε στο βαθμό που μπορούμε τις προσπάθειες της ε, σερβικής κυβερνήσεως, ελπίζοντας ότι στο εγγύς μέλλον θα μπορούμε να καταγράψουμε κάποια θετική εξέλιξη. Όσον αφορά την Κροατία, και πάλι δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες, πιστεύω ότι τις λεπτομέρειες πρέπει να τις συζητούμε στο δικαστήριο, μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Αλλά μια και πολλά πράγματα έχουν ήδη συστηθεί στο δημόσιο χώρο, στην κοινή γνώμη, έχουμε και ζητήματα σχετικά ε, με έγγραφα της επιχείρησης καταιγίδα. Με τις, με τις ε, υπηρεσίες του Ζάγκρεπ έχουμε ήδη αναπτύξει την επικοινωνία τη σχετική με την επιχείρηση αυτή. Εμείς ζητούμε να μας δοθεί δυνατότητα να διερευνήσουμε διεξοδικά τα έγγραφα αυτά. Δυστυχώς δεν έχουν ακόμη ε, ικανοποιηθεί αυτές οι επιθυμίες. Ακόμη περιμένουμε να δούμε τα έγγραφα και χαρακτηρίζουμε ως ευπρόσδεκτη την θέσπιση της ομάδα κρούσεως από τον Πρωθυπουργό Πρόσκο. Ωστόσο, σημειώνουμε ότι θα πρέπει οι εντατικέ τώρα προσπάθειες να διατηρηθούν έτσι ώστε να έχουμε θετικά αποτελέσματα από την Task Force το ταχύτερο δυνατό. Για τη Βοσνία. Όσον αφορά τη συνεργασία μα, την καθημερινή αν θέλετε συνεργασία με τη Βοσνία, δεν έχουν επισημάνω συγκεκριμένα ζητήματα, υποβάλλουμε αιτήματα, λαμβάνουμε τι απαντήσει Ε, διαρθρωτικής μάλλον φύση είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε σχέση με τη Βοσνία, φυσικά σε ένα νέο σε ένα θεσμό όπως ο δικός μας ε, πάντοτε είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε να μην ε, μπαίνουμε σε χωράφια πολιτικά, να μην παρεμβαίνουμε σε πολιτικά ζητήματα. Όταν όμως υπάρχουν ζητήματα ε, είτε άρσης ε, είτε ανανέωσης των θητιών των διεθνών δικαστών και του εισαγγελέα για τη Βοσνία, τελικά δόθηκε η παράταση της θητείας βέβαια των δικαστών και του εισαγγελέα, αλλά με μεγάλη καθυστέρηση είχαν ήδη αποχωρήσει από τη χώρα αρκετοί από αυτούς. Εν πάση όμως με ικανοποίηση σημειώνουμε τη λήψη της τελικής αυτής αποφάσεως και πιστεύουμε ότι η διεθνής παρουσία είναι ακόμα απαραίτητη. Εάν δεν είχαν ανανεωθεί αυτές οι εντολές αυτές οι θητείες θα είχαμε μεγάλα προβλήματα γιατί κάποιες από τις υποθέσεις θα έπρεπε να κλείσουν και να ανοίξουν από την αρχή. Οι διαδικασίες θα έπρεπε να ανοίξουν γιατί θα είχαν αποχωρήσει ή ε, επιφορτισμένοι με τους σχετικούς φακέλους δικαστές. Η δικαστική λοιπόν ε, διαδικασία, το δικαστικό διγύγναστε και εκεί χρειάζεται υποστήριξη, χρειάζεται υποστήριξη από την Εθνική Κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Ένωση ιδιαίτερως. Βρισκόμαστε σε καθημερινή συνεργασία επίσης με, τους, ε, με τις υπηρεσίες εισαγγελίων, εισαγγελέων που ασχολούνται με την πάταξη του εθνικού της, ε, των εγκλημάτων πολέμου. Η συνεργασία έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Πριν από 5-10 χρόνια θα λέγαμε ότι ήταν κατακόρυφη η σχέση δική μας με, την, ε, με τα τοπικά αυτά δικαστήρια, γιατί ήταν ε, η Χάγη εκείνη που έδινε κάποιες εντολές και ελάμβανε απάντηση, ενώ τώρα η κατάσταση είναι αμφίδρομη, η σχέση είναι αμφίδρομη, λαμβάνουμε και εμείς αιτήματα και δίνουμε απάντηση σε αιτήματα όπως και εκείνη ε, δέχονται τα δικά μας αιτήματα και ανταποκρίνονται σε αυτά. Τα τελευταία πέντε χρόνια και στο Ζάγκρεπ και στο Βελιγράδι και στο Σαράγεβο έχουμε αναπτύξει την αμφίδρομη αυτή συνεργασία με τους συναδέλφους στις σχετικές αρχές. Ύστερα από την απαόφαση για την θέση εφαρμογή της διαδικασίας ολοκλήρωσης ε, μετά το 2004 μεταφέρθηκαν 8 υποθέσεις στα εθνικά δικαστηρία για τις οποίες είχαν απεγγελθεί δικατηγορίες από το δικό μας δικαστήριο και έτσι αυτές οι υποθέσεις μεταφέρθηκαν στις ε, τρεις αυτές τις αγγελικές αρχές για τα εγκλήματα πολέμου που ήδη, και έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Έχουν φτάσει μάλιστα δύο από αυτές στην έφεση. Η μεταφορά ολοκληρώθηκε πριν από ένα μήνα με την αποστολή ε, ανακριτικού υλικού που είχαμε στη διάθεσή μας στη Χάγη και το αποστήλαμε στις, στις ε, για εγκλήματα πολέμου ε, στις αντίστοιχες χώρες. Για 43 υπόπτους τους είπαμε ότι δεν μπορούμε εμείς να, κάνουμε, να λάβουμε τη δίωξη από το δικαστήριό μας, αλλά ήμασταν βέβαιοι ότι μπορούσε να γίνει όπως έπρεπε η δίωξη στα τοπικά δικαστήρια. Και επίσης αναπτύσσαμε μια πραγματικά μια ουσιαστική εταιρική σχέση με τις υπηρεσίες αυτές, με μέγιστο επίτευγμα που θα ήθελα ρητά να αναφέρω, το γεγονός ότι από το περασμένο καλοκαίρι έχουμε μπορέσει να σωματώσουμε έναν ε, ε, ανακριτή δίωξη από την κάθε μία πρωτεύουσα, Βελιγράδη, Σαράγεβο και Ζάγκρεπ, που ασχολείται ε, με, με τις υποθέσεις που αφορούν τη χώρα του, λαμβάνει και αποστέλνει μηνύματα, αποτελεί λέει, το συνδετικό κρίκο, αλλά ταυτόχρονα διευκολύνει και το έργο των ε, δικών του, των εθνικών του δηλαδή ανακριτικών και εισαγγελικών αρχών, ε, διαβιβάζοντας τα μηνύματα και τα αιτήματα. Πράγμα το οποίο έχει υποστηρίξει βεβαίως και με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή ιδιαίτερως και την ευχαριστούμε, όπως έχει χρηματοδοτήσει και ε, σχέδια για την ενσωμάτωση 10 νέων ανακριτών στο, από τις από χώρες πρώην Από την ώρα που θα κλείσουν οι θύρες αυτού του Διεθνούς Δικαστηρίου σε μερικά χρόνια από τώρα, ξέρουμε ότι θα έχουν μπροστά τους δουλειά 10 με 20 χρόνια αυτοί οι ανακριτές και εισαγγελείς για ανακρίσεις και διερευνήσεις εγκλημάτων ε, πολέμου, εγκλημάτων γενοκτονίας και είμαστε ακράτατα πεπισμένοι ότι η τελική επιτυχία του, δικαστηρίου μας, του έργου του δικαστηρίου μας θα εξαρτηθεί από την ε, οργάνωση της μετάβασης ε, και μεταφορά των υποθέσεων αυτών από το δικαστήριό μας στα εθνικά δικαστήρια. Αυτή η σύνδεσμοι με την παρουσία τους μας προσφέρουν πολύ πρακτική βοήθεια, αλλά ταυτόχρονα έχουν και συμβολικό ρόλο να διαδραματίσουν, γιατί ε, αποδεικνύεται ότι τώρα ε, εργαζόμαστε σε ισότιμο επίπεδο για να διώξουμε τα ίδια εγκλήματα πολέμου, για να προσεγάγουμε τους ίδιους εγκληματίες πολέμου, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η αντιμετώπιση των προβλημάτων του παρελθόντος στην περιοχή. Δεν είναι πάντοτε βέβαια απρόσκοπτη συνεργασία. Ένα από τα προβλήματα που έχουμε είναι ότι η συνεργασία μεταξύ των χωρών της παραμένει δύσκολη. Και γιατί, διότι δεν υπάρχει νομική βάση παραδείγματι για έκδοση υπηκών από τη μία χώρα στην άλλη της πρώην Ιουκοσλαβίας. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαδικασίες μεταφοράς υποθέσεως από τη μία υπόθεση στην, στην άλλη. Ε, από, ε, υποθέσεως από τη μία χώρα στην άλλη. παράδοξο θα σας φανεί ίσως σε μια χώρα ενιαία στο παρελθόν όπου ήταν αυτονόητη μεταφορά μιας υποθέσεως εναγκλητικού υλικού. Τώρα όμως ε, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα και ελπίζουμε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να διαδραματίσουν ε, με την στήριξη που θα προσφέρουν στις χώρες οι οποίες τάσσονται υπέρ αυτής της, αλλαγή ε, αλλαγής αυτής της επικοδομητικό ρόλο. Θα σταματήσω εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν μόνο γενική η εισήγησή μου. Τρεις είναι οι βασικοί πυλώνες πάνω στους οποίου εργαζόμαστε, όπως ήθελα να σας εξηγήσω. Καταρχάς προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε το έργο που έχουμε σε εκκρεμότητα, τι εκκρεμίε δίκες. Έχουμε 25 κατηγορούμενους ε, σε Δίκε εκκρεμή ακόμη. Ξέρω ότι η ευρύτερη κοινή γνώμη μόνο την υπόθεση κάραζε και υπόθεση, αλλά υπάρχουν ακόμη 10 σημαντικέ δίκε με 25 κατηγορούμενους εκκρεμή, Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε και τον προπολογισμό και του λοιπούς ε, πόρου που μα χρειάζονται. Πρέπει επίση να εξασφαλίσουμε τη σύλληψη των λοιπών φυγάδων. Είμαστε ακράδαντα πεπισμένοι ότι η υποστήριξη Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ θα αποδειχθεί πολύτιμη και βεβαίω τρίτο πυλώνα η ενίσχυση της, ε, ε, του δικαστικού γίγνεσθε της, δικα, της δικαιοσύνης στις χώρες της περιοχής. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και είμαστε θέσεις σας για κάθε ερώτηση. <clears throat> Ε, σας ευχαριστώ κύριε Ισαγγελέφ θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας όλη φορά αυτό το ζήτημα στις 16.00 μέχρι 16.00. Ο συνάδελφο Πόστελ έχει το λόγο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπράμερτ. Δεν θέλω να πω ότι με αναφανδόν υπέρ του δικαστηρίου, ωστόσο έχω κάποιε επικριτικέ παρατηρήσει. Η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει με το ρόλο σα. Είσαστε γενικό Εισαγγελέα. Ομιλείτε εκ μέρου του δικαστηρίου αλλά το δικαστήριο δεν είστε μόνο εσείς. Έχει και δικαστές, έχει και κατηγόρους, έχει και συνηγόρους και άρα ίσως δοθεί εσφαλμένη εντύπωση ως προς την παρουσία σε εδώ και τον πολιτικό ρόλο του δικαστηρίου. Πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Σχετική με την ε, κατηγορία που απευθύνατε ως ελληπή συνεργασία με την ε, Κροατία. Εγώ θα ήμουν προσεκτικός εδώ γιατί η προκάτοχό σας μας είχε πει συγκεκριμένα εδώ ότι ξέρει πολύ καλά που βρίσκεται ο στρατηγός Κοτόβινα και μου είπε ότι βρίσκεται σε κάποιο μοναστήρι της ε, Βοσνίας Αρσεγοβίνης όταν τη ρώτησα και ότι ε, άλλοι λένε ότι είναι στο Βατικανό ενώ στην πραγματικότητα είναι στην Ισπανία. Ε, μάλλον αποδείχθηκε μετά ότι ήταν στην Ισπανία υπό την προστασία του Βατικανού και όταν τη στήσαμε να ζητήσει συγγνώμη για το λάθο αυτό και για τι κατηγορίε που απευθύνει, αρνήθηκε. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να προσέχουμε πάρα πολύ ω προ τι πληροφορίε που διαδίδουμε γιατί οδηγούν μερικέ φορέ σε παρεξηγήσει και παρερμηνίες. Πώ γνωρίζετε λοιπόν εσεί από τα έγγραφα στα οποία ε, τα οποία επικαλείστε ότι όντω υπάρχουν αυτοί οι φυγάδε ή για το πού βρίσκονται αυτοί οι φυγάδε. Και τελευταία ερώτηση ω προ το ζήτημα της συμφωνίας ε, έκδοσης, δεν υπάρχουν συμφωνίε έκδοση, μα είπατε, μα, ε, ναι, μπορεί να ήταν ένα κράτο, όπω είπατε η Ιουγκοσλαβία αλλά υποκομμουνιστική δικτατορία, υπό πόλεμο, υπό διώξεων και δεν είναι παράδοξο το ότι δεν υπάρχει εντωμεταξύ συμφωνία εκδόσεω. Εγώ ασφαλώ θα ήμουν υπέρ του να μην υπάρχει τέτοιου συμφωνία, διότι τέτοιο υλικό τόσο ευαίσθητο, τόσο ε, σοβαρό, θα έπρεπε με πολύ μεγάλη προσοχή να το χειριζόμαστε. Ευχαριστώ το λόγο η κυρία Ντεκάιζερ για τρία λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Μπραμέρτς. Γνωρίζετε πως ανέκαθεν στηρίζαμε τον αγώνα σας υπέρ της δικαιοσύνης και των ανθρωπινών δικαιωμάτων σχετικά με την συνεργασία του δικαστηρίου με την Κροατία. Ο κύριος Πόσελτ αναφέρθηκε σε αυτό το ζήτημα. Η, η Κροατία μετά από επανελειμμένα αιτήματα για τον πόλεμο που είχε γίνει για το 93-95 μετά από σύσταση ομάδας εργασίας ε, κάλεσε να συμμετάσχουν και τρίτη. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ερωτήσω εάν πιστεύετε πως η εργασία αυτής της, εργασία αυτής ε, ή καθαρά εργασίες πραγματογνωμοσύνης και θεωρείτε ότι θα πρέπει να συμμετέχουν και τρίτοι. Ποια είναι η καθαρα εργασιες πραγματογνωμοσυνης και θεωρειτε οτι θα πρεπει να συμμετεχουν και τριτη ποια ειναι η αποψη σας σχετικά. Έχετε κάποια γνώμη. Να δώσετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ντεκάιζερ. Η συνάδελφος Νέιτς έχει το λόγο που ήταν και η συγγήτρια για το δικαστήριο της Χάγης ε, στην προηγούμενη θητεία του Κοινοβουλίου. Τρία λεπτά. Κύριε Πρόεδρε και Μπράμερτς, αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω Πρόεδρε που αναφερθήκατε στην έκθεση μου που εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου. Με μεγάλη χαρά έκανα αυτή τη δουλειά και νομίζω ότι τα σχόλια των δύο συναδέλφων καταδεικνύουν πόσο, πόσα εμπόδια έχετε μπροστά σας και στον δρόμο που ακολουθείτε, διότι ο καθένας προσπαθεί να σας ε, πάρει με το μέρος του και να σας ε, φέρει στο πεδίο δράσης του. Πιστεύω λοιπόν ε, πως ε, η στάση σας πραγματι είναι αντίθετη με την στάση του προκατόχου σας. Το λέω αυτό με θετική έννοια. Ε, θεωρώ πως δεν θα πρέπει να υπάρξει ατιμορρησία, διότι αυτό είναι απαράδεκτο οποιαδήποτε και αν είναι η εθνικότητα, η εθνότητα, η θρησκεία κλπ. Νομίζω ότι το κατηγορτήριο είναι πάρα πολύ σοβαρό για τους εν λόγω, εν λόγω τώρα. Στην ε, Δημοκρατία της Σερβίας υπήρξαν ε, κάποιες ε, δραπετεύσεις ε, και οι καταδικασμένοι απέδρασαν η μας συνεργασία με τις διάφορες αρχές της Βοσνίας Ερζεγοβίνης ε, βελτιώθηκαν. Ίσως θα μπορούσατε να μας πείτε κάτι παραπάνω πάνω στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ, συνάδελφο Σβόμποντα. Έχει το λόγο πρόεδρο τη Ομάδα Εργασία για τα Δυτικά Βαλκάνια. Τρία λεπτά. Uh, Ευχαριστώ. Έχω δύο θέματα. Σε ό,τι αφορά τι ε, εκδόσει, συμφωνώ απόλυτα μαζί σα. Νομίζω ότι θα πρέπει να ασκήσετε πολύ πιο πολύ πίεση στι κυβερνήσει τη περιοχή γιατί ήταν ουσιαστικά ένας εμφύλιος πόλεμος που έλαβε χώρα και δεν μπορεί να αποδεκτώ, για παράδειγμα, να φεύγει κάποιο από την Κροατία να πηγαίνει στην Βοσνία Ζεγοβίνη και να μην υπάρχει δυνατότητα έκδοσης και νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό να τεθεί το θέμα αυτό, να σκεφτεί πίεση στις χώρες. Για το άλλο θέμα τώρα. Δεν έχετε ακόμη απαντήσει στη συνάδελφο Βερονίκ Τικάιζερ. Αλλά διαπιστώνουμε το εξή. Είσαστε πολιτική προσωπικότητα και η πολιτική είπαν ότι είναι σημαντικό. Υπάρχουν κάποια σημαντικά κριτήρια για τη συμπερίληψη, για την προσχώρηση των χωρών αυτών στην Ένωση. Νομίζω ότι και η ομάδα κρούσης έχει το έργο της και θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο η χώρα εκτελεί και ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της. Και τώρα το ερώτημά μου. Είπατε, και αν δεν είμαι και δικηγόρο, έχω σπουδάσει νομικά. Είπατε ότι δεν έχουμε πετύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την Κροατία και στη συνέχεια αναφέρατε ότι θα πρέπει να καταβληθούν και να συνεχιστούν οι προσπάθειε. Να συνεχιστούν οι προσπάθειες ή να γίνουν πιο Έντονε προσπάθειε γιατί στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επανέλθουμε σε αυτό που είπε ο κύριος Πόσελτ. Η Κροατία δεν συνεργάζεται πλήρως. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να, κάνουμε, να κάνει μεγαλύτερες προσπάθειες ή συνεργάζεται και πρέπει να συνεχίσει να καταβάλει τις ίδιε προσπάθειες. Ξέρετε, είναι δύο λέξει, αλλά περιέχουν μεγάλη πολιτική πολιτικό αντικτύπο για τη χώρα. Υπάρχει συνεργασία και πρέπει να διατηρηθεί το ίδιο επίπεδο συνεργασίας ή μήπως δεν γίνονται ακόμα επαρκείς προσπάθειες. Το οποίο δηλαδή θα, θα σήμαινε ότι η Κροατία ξέρει που βρίσκονται τα στοιχεία που λείπουν, αλλά δεν τα αναζητά. Αλλά αν αυτή είναι η αλήθεια, να το πούμε τουλάχιστον. Ε, Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον ε, εισαγγελέα Μπράμετς. Ε, αν θα μπορούσατε να μείνετε μέσα σε 5-10 λεπτά θα μας ε, εξυπηρετούσε το θέμα. Να ξεκινήσω με τα πρώτα δύο-τρία σχόλια. Θέσατε την ερώτηση κατά πόσο το έργο μας δεν είναι πολύ πολιτικά χρωματισμένο. Και το μοναδικό χρονικό σημείο στο οποίο είπα ότι εξ ονόματος του δικαστηρίου μιλάω ήταν όταν ανέφερα το ψήφισμα, γιατί νομίζω ότι πολιτικά δεν κάποιο θέμα, γιατί φυσικά το ψήφισμα υποστηρίζει όλο το δικαστήριο. Κατά τα άλλα, προσέχω πάντα ιδιαίτερα να μιλώ πάντα εξ ονόματος της Αγγλικής Αρχής και ξέρω ότι σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν διαφορές, όπως και σε εθνικό επίπεδο. Εγώ ίδιος θεωρώ ότι είμαι τεχνικός εμπειρογνώμονας, ο οποίος προσπαθεί στο βαθμό του δυνατού να συντάξει μία τεχνική έκθεση αναφορά για τα θετικά και αρνητικά στοιχεία και άλλοι θα κρίνουν το πολιτικό αποτέλεσμα. Προσπαθώ λοιπόν πάντα να μένω πάντα στα δικά μου χωράφια. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό και τακτικά με ρωτάνε και οι δημοσιογράφοι κατά πόσο θεωρώ ότι έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου να προσχωρήσει η Κροατία, η Σερβία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε καμία περίπτωση δεν απαντώ τέτοιε ερωτήσει. Δικό μου καθήκον είναι το όσο πιο αντικειμενικά γίνεται να παρουσιάσω τα στοιχεία, τα θετικά και τα αρνητικά. Και είναι, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα να κρίνω πολιτικά το αποτέλεσμα. Μιλήσατε για την προκάτοχό μου. Ε, δεν φαντάζομαι να περιμένετε σχόλια εκ μέρου μου προ αυτή την κατεύθυνση, αλλά είναι γεγονό ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε και με τι μυστικέ υπηρεσίε. Τα άτομα που αναζητούμε δεν είναι συνηθισμένοι εγκληματίε, είναι άτομα με πολιτικέ επαφέ, οι οποίοι, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον ε, στρατηγό Μλάντιτ, έχουν ιστορικέ σχέσει με τι μυστικέ υπηρεσίε, αλλά δεν θα προβώσω δηλώσει σε καμία περίπτωση και ποτέ δεν είπα ότι εκεί κρύβεται ο Μλάντης και παραδίπλα ο Χάτζιτ. σε καμία περίπτωση. Πάντα αυτό που έλεγα είναι ότι βάσει των στοιχείων που μας διαβιβάζουν οι Σέρβοι δεν έχουμε λόγο να θεωρήσουμε ότι, δεν βρίσκεται, ότι βρίσκεται στη Σερβία. Και πρόκειται για το ίδιο ερώτημα που έθεσε και τελευταίο ομιλητή σε ό,τι αφορά τι διαδικασίε έκδοση. Φυσικά πρόκειται για μια περιφέρεια, για μια περιοχή που μαστίστηκε, που μαστίζεται από πόλεμο. Και φυσικά υπάρχουν προβλήματα σε ό,τι αφορά τη διαδικασία συμφιλίωσης. Αλλά το θετικό είναι ότι τακτικά συναντιόμαστε με τους γενικού εισαγγελίε των τριών χωρών και ότι ε, καταρτίζουμε μια κοινή τράπεζα δεδομένων υπάρχει συντονισμός των εργασιών και νομίζω ότι η πρακτική συνεργασία έχει προχωρήσει περαιτέρω και από ότι θα διευκόλυνε και θα επέτρεπε ε, το νομικό πλαίσιο. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να το διευκρινίσουμε. Κυρία Ντεκάιζερ, μιλήσατε για θέματα συνεργασίας με την Κροατία. Είναι πολύ λεπτό το ζήτημα και δεν είναι εύκολο να απαντήσω το κατά πόσον οι εργασίες ε, της Επιτροπής ε, της Εξεταστικής Επιτροπής ε, είναι πιο πολιτικού ή τεχνικού χαρακτήρα. Δεν είναι προφανές για μας, διότι υποχρέωση συνεργασίας με το δικαστήριο, αυτή η υποχρέωση είναι υποχρέωση της κυβέρνησης, η οποία αποφάσισε να συστήσει αυτήν την Διοικητική Επιτροπή προκειμένου να οργανώσει τον όλα έγραφα, το, φάκελο κλπ. Ξέρετε, στο παρελθόν είχαν υπάρξει διάφορες διοικητικέ ε, επιτροπές για την αναζήτηση φακέλων. Η κυβέρνηση έλαβε ε, απόφαση να συστήσει αυτήν την task force. Εγώ δεν ε, θα ήθελα να κρίνω κατά πόσον πρόκειται για 90% πολιτικό, 10% τεχνικό, τεχνικής φύσης ή το αντίστροφο. Είναι δύσκολο να κάνουμε την διάκριση συχνά ανάμεσα στα δύο αυτά ζητήματα. Και ε, φτάνω τώρα στην ερώτηση που θέσατε στο τέλος, ότι δηλαδή <clears throat> τι επιθυμούμε από πλευράς Κροατίας. Με ρωτήσατε αν ε, ήμασταν υπέρ μιας ε, υποστήριξης από τρίτους και ή όχι. Και εδώ είναι πολύ λεπτή η θέση μου η Κροατία. Είναι μια, ένα κυρίαρχο κράτο που έχει την υποχρέωση να συνεργαστεί με το δικαστήριό μα. Αν η Κροατία κρίνει πω μια εξωτερική στήριξη και βοήθεια θα ήταν επωφελή, γιατί όχι. Εγώ προσωπικά δεν βλέπω ότι θα μπορούσαν να πράξουν τα λόγω άτομα επιπλέον. Αλλά, εν θα σα λέω ότι είναι δική του η απόφαση. Κυρία Νέιτς, με ρωτήσατε για το τι συμβαίνει στο Σεράγεβο στη Βοσνία. Όπως είπα, είχαμε αρκετές συνεδριάσεις με τους συναδέλφους ε, της υπηρεσίας ε, εγκλημάτων πολέμου. Ε, οι τελευταίες εξελίξεις φυσικά αποδυνάμωσαν αυτή την υπηρεσία και η Βοσνία φυσικά έχει τον μεγαλύτερο αριθμό φακέλων. Έχει χιλιάδες φακέλους οι οποίοι θα πρέπει να εξεταστούν, να γίνουν ανακρίσεις κλπ. Οι πόροι είναι περιορισμένοι, φυσικά αυτό αποτελεί τεράστια πρόκληση για τα προσεχή και κάθε πρωτοβουλία που μπορούσε να βοηθήσει τους αδέρφους εκεί επιτόπου είναι ευπρόσδεκτη. Τέλος, τελευταία ερώτηση αφορούσε στην παρουσίασή μου ότι αφενός είπε ότι όλα θα πρέπει να διατηρηθούν, αφετέρου χρειάζονται περισσότερες ε, προσπάθειες. Θα προσπαθούμε ως δικαστήριο να είμαστε ρεαλιστές ε, και κατά δύναμη αντικειμενικοί και ορθοί. Εάν στο τέλος ε, και φυσικά δεν γνωρίζω κατά πόσον τα λόγω έγγραφα καταστράφησαν ή όχι. Αυτό το οποίο γνωρίζω όμως είναι ότι αυτά τα έγγραφα υπήρξαν και οι Κροάτες συνεργάτες μας συμφωνούν. Εμείς ε, διαφωνούμε σε ό,τι φορά τον αριθμό των εγγράφων, αλλά για κάποιες επιχειρήσεις όπως ποιες καταιγίδα χρειάζονται τις στρατιωτικές χάρτες και άλλα έγγραφα. Επίσης υπήρξαν πολλοί ε, που συμμετείχαν στην αφαίρεση αυτών των εγγράφων. Αυτό το οποίο δεν γνωρίζουμε κατά πόσο τα εν λόγω έγγραφα, κατεστραμμένα ή μη, εάν και κάποια αντίγραφα τα οποία κάπου ε, βρίσκονται. Αυτό το οποίο μου ζητάτε είναι ε, σωστό και πρέπει θέλουμε να ε, είμαστε συνεκτικοί, δηλαδή να κάνουμε μια σειρά συστάσει στις ακροατικές αρχές, διότι θεωρούμε ότι ορισμένες οδοί δεν ακολουθήθηκαν σωστά και να είμαστε και αξιόπιστοι σχετικά με την παρουσίαση των εγγράφων από πλευρά του. Εμεί δεν ε, περιμένουμε κάτι το αδύνατο από πλευρά του ή το, το ακατόρθωτα. Είπαμε ότι αναγνωρίζουμε την ε, σημασία της σύστασης αυτής της ταξης για την κυβέρνηση μας είπε ότι τώρα αυτή είναι μια ε, απασχόληση μια πλήρη απασχόληση full time. Θα προτιμούσα αυτό να είχε συμβεί πριν από δύο έτη, όταν είχαμε κάνει το αρχικό αίτημα, αλλά όχι τώρα, αλλά θεωρούμε ότι είναι ένα θεωρητικό στοιχείο. Γνωρίζουμε επίση ότι αυτή η task force εργάζεται και παροτρύνουμε τις αρχές να συνεχίζουν να δουλεύουν προκειμένου να ευρεθούν αυτά τα έγγραφα. Αυτά, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Ε, επόμενες παρεμβάσεις, δύο λεπτά. Η κυρία Κόπα, δύο λεπτά. Ε, κύριε Μπράμερτ, ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω στο... Ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να σας ευχαριστήσω για τις προσπάθειες που καταβάλλετε για την απόδοση δικαιοσύνης στα εγκλήματα που έλαβαν χώρα στην πρώην Ιουγκοσλαβική Ομοσπονδία. Ε, θα ήθελα παράλληλα να καλωσορίσω και την πρόσφατη έκθεσή σας για τη Σερβία προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ η οποία επέτρεψε την απεμπλοκή της ενδιάμεσης εμπορικής συμφωνίας, φέρνοντάς την ένα βήμα πιο κοντά ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις ε, σχετικές σας δηλώσεις αναγνωρίσατε ότι η Σερβία σημείωσε συνεχή πρόοδο στη συνεργασία για τη σύλληψη του Ράτκο Μλάντιτς και του Γκόραν Χάτζιτς και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου αποφάσισε ότι θα επανεξετάσει το ζήτημα της κύρωσης της Συμφωνίας Σύνδεσης και Σταθεροποίησης τους επόμενους έξι μήνες. Αυτό μας δείχνει ότι το συνδέει απόλυτα με την επόμενη εξάμηνη έκθεση που θα παρουσιάσετε τον Ιούνιο. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω και νομίζω είναι σημαντικό για την Επιτροπή αυτή να ξέρει τι ακριβώς ζητάτε ακόμα από τη Σερβία μέσα στους επόμενους μήνες, εκτός προφανώς από την ίδια σύλληψη των εγκληματιών. Τι νόημα δίνεται στον όρο που και εμείς χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά σε όλα τα κείμενα, πλήρη συνεργασία. Τι υπάρχει ακόμα που μπορούσε να έχει κάνει η Σερβία και δεν έχει κάνει ε, ώστε να οδηγηθούμε στη σύλληψη των δύο αυτών εγκληματιών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριο Κάτσιν, δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κυρία Μπράμερτς να σας συγχαρώ για το έργο σας ως εισαγγελέα. Πέρα από το ότι πολλοί δεν ικανοποιούνται με τα απορίσματα του Δικαστηρίου της Χάκης, νομίζω ότι είναι σημαντικό, πραγματικά κρίσιμη σημασία να διώκονται οι εγκληματίε πολέμου. Είναι πραγματικά κρίσιμο το έργο σας και θεωρώ ότι όχι μόνο δημιουργείτε τους σωστούς όρους για να κινηθούμε από τη συλλογική ευθύνη η οποία επικρατεί στην περιοχή, γιατί κατηγορούνται ολόκληρα έθνη για εγκλήματα, να περάσουμε λοιπόν στην ατομική ευθύνη, στην ευθύνη συγκεκριμένων ατόμων α, της ε, περιοχής. Και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να προσεχθούν το συντομότερο δυνατόν τα άτομα αυτά. Αυτό θα ευνοήσει και την πολιτική ατμόσφαιρα και την συμφιλίωση στην περιοχή. Και είναι σημαντικός και πολιτικός αντίκτυπος, γιατί εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορέσουμε στην περίπτωση αυτή να ξεκινήσουμε την επικύρωση τη Συμφωνία Σταθεροποίηση και συνεργασία. Αλλά η πρόοδος της συνεργασίας ε, με τη Σερβία καταδεικνύει ότι η εφαρμογή της ενδιάμεσης ε, εμπορικής ε, συμφωνίας θα τεθεί σύντομα σε εφαρμογή. Αλλά αυτό που προέχει, θεωρώ, είναι κάτι άλλο. Τα εγκλήματα αυτά να ενταχθούν και να βρουν τη θέση τους στη συλλογική ευρωπαϊκή μας μνήμη σε ό,τι αφορά δηλαδή και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Δυτικά Βαλκάνια. Γιατί γίνεται στο Βαλιγράδι σήμερα μια πολύ αμφιλεγόμενη συζήτηση για το κατά πόσο θα πρέπει να τοποθετηθεί η Σερβία σε ό,τι αφορά τα εγκλήματα τη Ρεμπρένιτσα. Αν ήταν γενοκτονία ή όχι, αν χρειάζεται ένα ενιαίο ψήφισμα ή πολλά ψηφίσματα σχετικά. Θα ήθελα να ακούσω τη δική σα άποψη, αν θα θέλατε να μα ε, την παρουσιάσετε. Νομίζω ότι η Σερβία θα χρειαστεί μια φάση ομφαλοσκόπησης και στοχασμού για να ταινίσει το μέλλον. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό και θα είναι και πολύ απλή η εξατομίκευση, αν θέλετε, της ευθύνης, γιατί ε, πρέπει να προσαχθούν πιο πολλά άτομα πέρα από τον Λάντιτς και τον Κάρτζιτς και τον ε, Ο συνάδελφος Αγκουράκης για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, έχω τη γνώμη ότι και από την παρουσίαση που ακούσαμε σήμερα και από τις εξελίξεις ότι έχει φτάσει ο καιρός πια αυτό το δικαστήριο να σταματήσει τη δράση του. Ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό δημιουργήθηκε ω αποτέλεσμα του Νατοϊκού πολέμου στη Ιουκοσλαβία και είναι προφανέ, δέκα χρόνια έχουν περάσει από τότε, ότι αντικατοπτρίζει τη δίκη, την ε, δικαιοσύνη των νικητών στον πόλεμο. Προ υπεβεβαίωση των όσων λέω, θα ισχυριστώ ότι η ύπαρξη αυτού του δικαστηρίου και εμπολής η άδικη δράση του ε, είναι παράγοντας ε, αστάθειας στα Βαλκάνια και σε όσους θα αντιτείνουν ότι δήθεν αυτό το δικαστήριο είναι αναγκαίο για να τιμωρηθούν τα εγκλήματα πολέμου τα οποία προφανώς και υπήρχαν αλλά δεν είναι έργο ε, των νικητών να τα κρίνουν θα τους πω ότι παρά την ύπαρξη αυτού του δικαστηρίου έγινε η γενοκτονία στη Γάζα και δεν είδα το, στο δικαστήριο να, να πηγαίνουν οι υπεύθυνοι του Ισραήλ και δεν είδα επίσης Παρά το γεγονό ότι ο κύριο Τόνι Μπλερ αναγνώρισε ότι είπε ψέματα στην κοινή γνώμη τη Βρετανία και του κόσμου για τον πόλεμο στο Ιράκ, δεν είδα κανέναν να θέλει να παραπέμψει τον κύριο Μπλερ στο δικαστήριο αυτό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε κύριε Μπράμερτς. Είναι μεγάλο το ηθικό βάρος που έχετε. Σας έχουν αναθέσει την, ε, το έργο τη συμβολή στην κάθαρση για όσα έχουν γίνει στην περιοχή και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεχίσετε το έργο σας. Επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια θετικά και για την ε, προκάτοχό σας η οποία κατέβαλε τεράστιες προσπάθειες για να βγάλει νόημα, για να πετύχει αποτελέσματα, για να μην περάσουν τα εγκλήματα ατιμόρυτα. Και ίσως κάποιοι ξεκίνησαν να γράφουν τα απομνημονεύματα τους λίγο ε, πρόωρα. Ελπίζω να χρησιμοποιήσετε το χρόνο που θα χρειαστείτε για να αναλογιστείτε πρωτού ξεκινήσετε κι εσείς κάποιο τέτοιο έργο. Για την Κροατία τώρα, την οποία, από την οποία, για την οποία όλοι θέλουμε να προσχωρήσει σύντομα στην Ένωση. Αν συνεχίσει τις εργασίες όπως προβλέπετε. Και είμαι σίγουρος ότι το Κοινοβούλιο θα το θα συνεχίσει την ε, παρακολούθηση των εργασιών αυτών. Νομίζω ότι έγινε ένα μεγάλο λάθος όταν δόθηκε άφεση σε ένα άτομο που δολοφόνησε ένα παιδί. Και αυτό καταδεικνύει πόσο σημαντικό είναι να επέλθει αυτή η κάθαρση που ανέφερα προηγουμένως. Και μάλιστα να επέλθει με τρόπο ε, το σε όλη την περιοχή. Σα ευχαριστώ. Ολοκληρώνει ο κ. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε και όπω και οι υπόλοιποι καλωσορίζω την, ε, τον κύριο Μπρέμετς, και είμαι βέβαιος ότι η υποστήριξή μας είναι σημαντική προς το στήριο σας και είναι σημαντικό να συνεργαζόμαστε και με τις χώρες της περιοχής για να πετύχουμε τα ευκταία αποτελέσματα. Να ρωτήσω αν θέλετε να σχολιάσετε σε ό,τι αφορά τις ε, περιπτώσεις εγκλημάτων, ε, εγκλημάτων πολέμου εντός της δικαιοδοσίας της Κροατίας. Όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, θα σας αναπευθούν ε, τέτοιες υποθέσεις δεδομένων των, της απόδοσης του δικαστικού συστήματος στην Κροατία. Πιστεύετε ότι οι υποθέσεις που θα αναπευθούν στο δικαστικό σύστημα της Κροατίας θα τύχουν τη σωστή εξέταση και αν μπορείτε να σχολιάσετε επίσης κατά πόσο δεν υπάρχουν διακριτικές μεταχειρήσεις βάσει εθνότητας σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των εγκλημάτων πολέμου εντός του δικαστικού συστήματος της Κροατίας. Υπάρχει ακόμα μια παρέμβαση ενός λεπτού του Πρόεδρου της Πολιτικής Ασφάλειας ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ακούσαμε 10-12 παρεμβάσει σήμερα. Μιλήσαμε για την Κροατία, την υποβολή εγγράφων κλπ. Έχουμε όμω τον Μπλάντιτ, ο οποίο συνεχίζει να παραμένει ελεύθερο. Εδώ και 15 χρόνια μετά τη Στρεμπέντσα. Μιλάνε για πρόοδο, διερωτώ μας επίσης κατά πόσον είναι πλήρης ε, συνεργασία των σερβικών ε, αρχών εγώ χαίρομαι για την πρόοδο που έχει υπάρξει, αλλά μπορείτε να μας πείτε κάτι παραπάνω, διότι υπάρχει ένας φυγάς ε, και πρόσφατα έλαβε χρήματα από τις ε, σερβικές αρχές, ε, την σύνταξή του κλπ. Αυτό και αυτό συνέβη μέχρι πριν από μερικούς μήνες. Εντάξει, μιλάμε για πρόοδο, αλλά τι είδους είναι αυτή η πρόοδο. Μπορούμε, πιστεύετε, να έχουμε κάποια από τα αποτελέσματα σύντομα και να μην μιλάμε με γενικόλαγα, χωρίς να έχουμε αποτελέσματα αυτά. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Ντόνζο. Ο κύριος Αγγελές έχει το λόγο. Παρακαλώ, μπορείτε να παραμείνετε μέσα στο χρονικό πλαίσιο των τεσσάρων. Παρακαλώ. Πρώτη ερώτηση σε ό,τι αφορά το τι περιμένουμε από τη Σερβία και φυσικά είναι η πρώτη και τελευταία ερώτηση αυτή που ακούσαμε. Απαντά ταυτόχρονα. Τον Μάιο θα καταρτήσουμε μία ειδική έκθεση όπου θα αναφέρουμε τι έχει επιτευχθεί από την τελευταία έκθεση του Δεκεμβρίου. Πέρα από το θέμα των φυγάδων, τα πράγματα είναι business as usual. Έχουμε το Συμβούλιο της Συνεργασίας με τον κύριο Λάιτ. Υπάρχει καλή συνεργασία, λαμβάνουμε όλα τα έγγραφα που ζητάμε. Επίσης υπάρχει το θέμα των φυγάδων πέραν αυτού. Και δεν θέλω να δώσω την ε, εντύπωση, κάθε άλλο, ότι όλα είναι τέλεια και ότι δεν χρειαζόμαστε τίποτα παραπάνω, δεν χρειάζονται περαιτέρω κίνητρα σε καμία περίπτωση. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό ως εισαγγελέα για μένα να είμαι αξιόπιστος. Συνεργαζόμενος λοιπόν με τις, με τις υπηρεσίες αυτές σε εβδομαδιαία βάση. Έως τώρα εμπιστεύδομαι την δέσμευσή τους να πετύχουν το ευκταίο αποτέλεσμα και λαμβάνω τεχνικές ε, ενημερώσεις για τα θέματα αυτά. Δεν μπορώ να επισέλθω σε λεπτομέρειες, το καταλαβαίνετε, αλλά παρακολουθώ στενά τις λειτουργικές αυτές δραστηριότητες αν στεφτούν με επιτυχία, και κάποιες έχουν ήδη στεφτεί με επιτυχία, θα έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα μέχρι τον Ιούνιο. Αν όμως κάποιες από αυτές δεν στεφτούν με επιτυχία και αν η ποιότητα κάποιων ενεργειών δεν είναι αυτή που επιθυμούμε, θα αναφερθεί αυτό στην έκθεση. Το επαναλαμβάνω ότι η σύλληψη των φυγάδων αποτελεί την υπαριθμό ένα προτεραιότητα. Στην πραγματικότητα είναι πολύ περιορισμένο ο αριθμό των ατόμων που είναι, έχουν εντολή, ε, τους έχει ανατεθεί η αναζήτηση των φυγάδων. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητο το εγχείρημα αυτό και στην τελευταία έκθεση τα θετικά στοιχεία που αναφέρθηκαν σε ό,τι αφορά τις λειτουργικές αυτέ ομάδε από θετική πλευρά, ήθελα να τους ενισχύσω, να τους ενθαρρύνω, να συνεχίσουν το έργο τους. Θα δούμε όμως τι θα έχουμε πετύχει σε ορισμένους μήνες. Για το δικαστήριο εξορισμού δεν ε, κάνει δίωξη χωρών, γίνεται δίωξη ατόμων. Αυτό είναι σαφές στην περιοχή. Δεν έχουμε πρόβλημα με τη Σερβία, με το σερβικό λαό. Αναζητούμε συγκεκριμένα άτομα τα οποία έχουν ατομική ευθύνη για κάποια από τα πιο φρικτά εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί στην Ευρώπη. Είναι σαφές ότι διώκονται άτομα και η συνεργασία με τις υπηρεσίες επιτόπου κινούνται, κινείται προς την ίδια κατεύθυνση. Τώρα για ε, τα ψηφίσματα δεν θα σας προκαλέξει έκπληξη ότι αυτό, ότι θα σας πω ότι είναι ιστορικό το ζήτημα αυτό της Σερβίας. Τώρα, σε ένα πιο ευρύ πλαίσιο, επειδή και έργο μας είναι να διευκολύνουμε τη συμφιλίωση και αυτό θα μπορούσαμε να το ζητήσουμε επί ώρες και καταλαβαίνω ποιοι είναι οι περιορισμοί που αντιμετωπίζουμε. Η συμφιλίωση αποτελεί ένα πολύ πιο ευρύ θέμα και πιστεύω ότι οι τοπικές πολιτικές αρχές θα πρέπει να διδραματίσουν πολύ πιο σημαντικό ρόλο. Θα έχετε δει στον τύπο, κατά πάσα πιθανότητα, ε, το Δεκέμβριο αναφέρθηκε ότι το 65% του πληθυσμού στη Σερβία είναι κατά της έκδοσης του στρατηγού Μλάντιτς. Όλοι νομίζω ως δικαστήριο, ως πολιτική, ως διεθνής κοινότητα θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αν δεν καταφέρουμε να εξηγήσουμε σε εκατομμύρια ανθρώπους ενός μελλοντικού ενδεχομένως ε, κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το τι πιστεύουμε για τον στρατηγό Μλάντιτς δεν θα έλεγα ακριβώ ότι πρόκειται για γενική αποτυχία, αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό θα αποτελούσε μία ένδειξη ότι θα πρέπει να γίνουν πολλά παραπάνω. Θα πρέπει λοιπόν οι πολιτικοί, οι τοπικοί, να διαδραματίσουν πιο έντονο ρόλο και να υποστηρίξουν το έργο τη διεθνού δικαιοσύνη. Τελευταία ερώτηση. Για το πόσοι εμπιστοσύνη έχουμε στο δικαστικό σύστημα της Κροατίας. Ξέρετε ότι ο Γενικός εισαγγελέα της Κροατίας είναι ο Γενικός Εισαγγελέα Βάιτς, ο οποίος είναι συνάδελφος με τον οποίο συνεργάζομαι επί α, κάποιο καιρό τώρα και πραγματικά εμπιστεύομαι την ηγεσία του. Ποτέ δεν μας έχει δώσει λόγο να αμφισβητούμε τη δέσμευσή του για την εξέταση των υποθέσεων αυτών. Φυσικά, σε ό,τι αφορά τους πόρους, τα πράγματα δεν είναι τέλεια και ιδανικά. Ιδιαίτερα εν ώψη του αριθμού και του όγκου των διώξεων που, α, με τους οποίους έχουν επιφορτιστεί. Το βασικό πρόβλημα είναι ουσιαστικά η Βοσνία, γιατί ο αριθμός των υποθέσεων σε σχέση και σε σύγκριση με τους πόρους που διατίθενται, είναι σαφές ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να εξεταστούν όλες αυτές οι υποθέσεις, ούτε καν ένας μικρός αριθμός εξ αυτών. Δεν ξέρω αν απάντησα έτσι όλες τις ερωτήσεις σας. Το ελπίζω. possiamo concludere a questo punto. Μάλιστα. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε στο σημείο αυτό αφού προηγούμε να ευχαριστήσουμε τον εισαγγελέα κύριο Μπράμερτς για την παρουσία του και για την ευγένεια που είχε να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις αλλά και να ανταποκριθεί στο αίτημα της ε, Επιτροπής μας να τον ευχαριστήσουμε για την σημαντικότατη εργασία του και του υποσχόμεθα ότι θα είμαστε στο πλευρό του. Ευχαριστώ να κάνουμε μια διακοπή μερικών λεπτών τεχνικής φύσης και θα ξεκινήσουμε με το επόμενο σημείο, δηλαδή με την ακρόαση του κυρίου Φουερέ, ειδικό εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, καθώς επίσης και το ψήφισμα σχετικά με την έκθεση προόδου της πρώην Ιουκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας για το 2009 του συναδέλφου Τάλερ.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 Συνάδελφοι, πέρασαν τα δύο λεπτά, επαναλαμβάνουμε τις εργασίες μας, έχουμε ανάμεσά μας ε, τον προσεκλημένο μας, ε, τον δόκτωρ Ερουάν Φουερέ, ειδικό εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Είναι η τέταρτη φορά, κύριε Φουερέ, όπου εσείς ως ειδικό εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, παρίσταστε σε ακρόαση στην Επιτροπή μας και αυτό καταδεικνύει το ενδιαφέρον του Κοινοβουλίου για τις εξελίξεις ε, στην περιοχή που εσείς ελέγχετε. Α, και τι εξελίξεις έχουν υπάρξει. Η Επιτροπή μας σήμερα, μάλιστα, θα εξετάσει παράλληλα με την ακρόασή σας τις τροπολογίες ε, επί ε, ψηφίσματος ε, για την έκθεση πρόοδο της πρώην Δημοκρατίας της Μακεδονίας του κ. Τάλερ θα ψηφίσουμε από το πρωί. Έχει υπάρξει μια πολύ σημαντική διαδικασία προσέγγισης και οι αρχές της Ιουκλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας κατέδειξαν πως έχουν την ικανότητα και τη δυνατότητα να ε, μαθαίνουν από τα σφάλματά τους προκειμένου να εφαρμόσουν τα όσα τους έχουν ζητηθεί προκειμένου να υπάρξει μια προσέγγιση περαιτέρω με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από την τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία εξετίμησε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και συνέστησε στην εκκίνηση των διαπραγματεύσεων για την ένταξη. Μολόντως λοιπόν υπάρχουν αυτές οι σημαντικές θετικές πρόοδοι, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Υποθέσεων του 6 Δεκεμβρίου αποφάσισε να ε, καθυστερήσει τη λήψη απόφαση για την έκθεση διαπραγματεύσεων στο Συμβούλιο του Μαρτίου. 10 Μαρτίου και να ξεβρεθεί μια συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση αναφορικά με την ονομασία αυτού του ε, νομικού μορφώματος που θα δώσει επιτέλους ε, τέλος ε, σε αυτή τη διαμάχη. Η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία θα πρέπει να αντιμετωπίσει φυσικά και οι προορέ προκλήσει. Η μεταρρύθμιση τη δικαιοσύνη, η περαιτέρω ενίσχυση ανεξαρτησία τη, η καταπολέμηση τη διαφθορά, η βελτίωση τη ε, διοίκηση και πρόοδο στο ανθρώπινα δικαιώματα, βελτίωση εφαρμογή της συμφωνία του όριτ ε, και σχέσεις με την αλβανική μειονότητα. Θα πρέπει να πούμε ότι από, από τον 19 Δεκεμβρίου οι πολίτες της ε, πρώην ε, Ιγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας έχουν, απολαμβάνουν μια ελευθερία σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία και διακίνηση στο πλαίσιο της, ε, του χώρου Σέγγεν, διότι έχουν καταργηθεί οι προξενικές θεωρήσεις. Όλα αυτά λοιπόν ε, είναι πολύ ενδιαφέροντα, αλλά φαντάζομαι ότι αυτά που θα έχετε να μας πείτε θα είναι ακόμα πιο ενδιαφέροντα. Αγαπητέ κύριε Φούερε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εξέτοιμα μέλη της Επιτροπής των Εξωτερικών. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να πάρω στο ενώπιον σας και έτσι να συνεχίσουμε και σήμερα την ε, παράδοσή μας της ετήσιας συνάντησης ε, που έχουμε διατηρήσει από τον Νοέμβριο του 2005 τον οριστικά ειδικό πρόσωπο για την πρώην Δημοκρατία της Μακεδονίας. Και δεν θέλω να αναφερθώ ιδιαίτερα και στον ε, ρόλο που διαδραματίσετε εσεί για τη συμφωνία για την απελευθέρωση καθεστώ θεώρηση Βατηρίων. Ήταν καθοριστικό χώρο αυτό, όχι μόνο για την ε, παγίωση του κύρου σα, αλλά και διότι δείξατε στου πολίτε τη χώρα αυτή, όπω και άλλων γειτονικών χωρών, ότι οι σκληροί κόποι του και οι προσπάθειέ του για τη μεταρρύθμιση βρίσκουν ανταπόδοση και ανταμοιβή και όσοι ήσασταν παρόντες για, την, για τους εορτισμούς στις 18 Δεκεμβρίου στη Μεγάλη Πλατεία των Σκοπίων θα είδατε με πόση χαρά δέχτηκαν την ανακοίνωση, υποδέχτηκαν την ανακοίνωση αυτής της αποφάσεως οι πολίτες της χώρας. Επίσης θέλω ευχαριστήσω τον κύριο Ταλόρ για την, ε, Τάλερ για την ε, δουλειά που έχει κάνει και προετοιμάζοντα την έκθεση για τον κύριο Χατζημαρκάκη για τη συνδρομή συμβολή του ω Προέδρου τη Επιτροπή. Και περιμένουμε βεβαίω και την έκθεση Επιτροπή των Εξωτερικών και τη Μικρή Κοινοβουλευτική Επιτροπή που του αναμένουμε με τι αντιπροσωπείε του στα Σκόπια ε, το Φεβρουάριο. Έχει μεγάλη σημασία η Μεκτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή με το ρόλο τη, ενισχύει τι σχέσει μεταξύ των δύο κοινοβουλίων και ενθαρρύνει τι μεταρρυθμίσει στην χώρα. Ελπίζω δε αυτό να συνεχιστεί. Κύριε Πρόεδρε, όπως επισημάνατε το 2009 ήταν όντω έτος με θετικές εξελίξεις για τη χώρα. Ήταν ένα καλό έτος. Είχαμε και προεδρικές και τοπικές εκλογές που σε μεγάλο βαθμό ε, ενίσχυσαν την δημοκρατική αξιοπιστία της χώρας και τις επέτρεψαν να φτάσει σε προδιαγραφές διεθνούς επίπεδος προς την διεξαγωγή των εκλογών με τις ε, αποστολέ των παρατηρητών. Αρχές ε, του Θέρους και του Φθινοπόρου είχαμε επίσης μια ενισχυμένη διαδικασία εκδημοκρατισμού με την ορμή που είχε πάρει αυτή η διαδικασία της αλλαγής και βεβαίως την, θέση, την ανάλυση μάλλον των καθηκόντων του νέου, ε, του νέου Κοινοβουλίου που ε, οφείλουμε στο σύνολο αυτή τη διαδικασία στην συνεργασία των συντονιστών και τα ορόσημα που όρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που συχνά ορίζονται συνενετικά. Η Επιτροπή επίσης αναγνωρίζει από πλευρά της τις προσπάθειες αυτές με την ε, πρόταση της για την ημερομηνία εκείνης των διαπραγματεύσεων. Επίσης ε, έκλεισε και το ζήτημα του προσδιορισμού των συνόρων με το Κοσμοπέδιο πέρυσι ακόμη. Έτσι λοιπόν η πρώην Οικοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας είναι η πρώτη χώρα στην περιοχή που έχει επιλύσει όλα αυτά τα προβλήματα και είναι με τον τρόπο αυτό η χώρα η οποία συμβάλλει ε, στη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή. Αυτό χάρη και στην συμμετοχή της στην ε, αποστολή άντρια της του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμβάλλει δηλαδή και με τα στρατιωτικά μέσα στην σταθερότητα στην περιοχή. Υπήρξαν βέβαια κάποια προβλήματα όπως ε, η δημοσίευση της ε, αμφιλεγόμενης εγκυκλοπαίδειας, η οποία προκάλεσε πολλές ανησυχίες και φόβους ε, στην περιοχή, στις κοινότητες της περιοχής και που τελικά αποσύρθηκε. Επίσης θα ήθελα να σημειώσω ότι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου έγιναν δεκτά με απογοήτευση μάλλον. Έχουμε υπογραμμίσει και πολλές φορές υπογραμμίσει στην κυβέρνηση της χώρας αυτής ε, τη σημασία της ε, επίλυση του ζητήματο του σχετικού με το όνομα. Έχουν λάβει χώρα κάποιε θετικέ εξελίξει με τι συναντήσει μεταξύ των δύο πρωθυπουργών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη εμπιστοσύνη, πάνω στην οποία θα πρέπει τώρα να οικοδομήσουμε και πιστεύουμε ότι έχει έρθει πλέον η στιγμή ηγετική παρησία και θάρρος να προσδιορίσουν το νέο πεδίο για την εξέβριση μια λύσης. Αναμφίβολα, οι έξι προσεχείς μήνες είναι απαραίτητο να αξιοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Κάθε περαιτέρω καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές δυσκολίες μεταξύ των διαφορών εθνοτικών ομάδων και κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε ενδεχόμενη αστάθεια. Ποιε είναι οι μεγάλε προκλήσει που έχει η χώρα ενώπιον τη, πέραν της επίλυσης του, προβλήματος, ε, του ζητήματος του ονόματος, έχουμε την ενίσχυση του δημοκρατικού πολιτικού διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών. Το προηγούμενο Δεκέμβριο είχα την ευκαιρία να προσκαλέσω σε, μια, σε ένα δείπνο ε, επί τη ευκαιρία του νέου έτους με τους ε, πολιτικούς ηγέτες. Ήταν η πρώτη φορά, πρέπει να σας πω, που συναντιόντουσαν από τον Ιούλιο που είχε προηγηθεί. Μεγάλες προσπάθειες λοιπόν χρειάζονται από όλους και από κάθε πλευρά ε, για την επίλυση των προβλημάτων. Και βέβαια και η κυβέρνηση πρέπει να δώσει πρώτη το παράδειγμα. Η κυβέρνηση φύμβλεται, ελέγχει και το κοινοβούλιο και την Προεδρία και τα δύο τρίτα των ε, τοπικών αρχών δημών και κοινοτήτων. Άρα έχει μεγάλη ευθύνη, πρέπει να την χειρά βοηθείας και κάθε ένας από τους πολιτικές ηγέτες πρέπει να εξαντλήσει τις ε, προσπάθειές του σε επικοδομητική στάση και όχι σε ανταλλαγή προσβολών όπως είδαμε δυστυχώς τις τελευταίες εβδομάδες αλλά σε επικοδομητικές προσπάθειες, σε μεταρρυθμίσεις αποτελεσματικές και σε κοινέ προσπάθειες για την επίλυση του προβλήματος του ονόματος γιατί αυτό μόνο με κοινή προσπάθεια μπορεί να αντιμετωπιστεί. Και έτσι με τη συνενετική αυτή προσπάθεια θα μπορέσουμε ελπίζω να έχουμε εξελίξεις. Ε, στην προσπάθεια αυτή έχουμε το Εθνικό Συμβούλιο για την ε, ένταξη που μετέχουν η κοινωνία των πολιτών, οι πολιτικές αρχές, η εκκλησία, η θρησκευτική ηγεσία και ε, χρειάζεται υποστήριξη και από την κυβέρνηση για να αναπτύξει έναν ευρύτερο διάλογο μεταξύ όλων των παραγόντων της χώρας. Άλλο η σημαντική πρόκληση είναι η συμφωνία πλαίσιο της Οχρίδας που αποτελεί το μόνο πλαίσιο για την εξασφάλιση της στοιχιζόμενης πολιτικής σταθερότητας και την αντιμετώπιση των διαφυλετικών συγκρούσεων. Σημαντική είναι η πρόοδο που έχει σημειωθεί αναμφίβολα μεν, αλλά χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια και περισσότερη πρόοδο. Δεν ε, λείπει η νομοθεσία ή η εφαρμογή τη νομοθεσία, όσο περισσότερο η ευαισθητοποίηση ω προ την ε, υλοποίηση του πνεύματο τη συμφωνία αυτή τη Οχρίδα αυτό είναι το έλλειμμα που σημειώνουμε και το σημειώνουμε ιδιαίτερα στο χώρο της παιδείας, όπου τα τελευταία χρόνια παρουσιάστηκε μια επικίνδυνη τάση για ε, διαφορετικές ή χωριστές τάξεις, γλωσσικά διαχωρισμένες τάξεις, ένα είδος διαχωρισμού που ευτυχώς ε, ανετράπει ως τάση τώρα, χάρη και στις ε, συστάσεις του είπα του εκπροσώπου για τις μειονότητες του ΩΣΑ, αλλά άλλη μια σύσταση του είπα του εκπροσώπου που μιλούσε για την διδασκαλία της επίσημης γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στα αλβανόφωνα σχολεία οδήγησε σε πολλές αντιδράσεις, ακόμη και σε αποκλεισμό ή αποχή από, τις, ε, από τα μαθήματα των ε, μαθητών. Δηλαδή βλέπουμε ότι δεν υπάρχει επαρκής προσπάθεια για προετοιμασία του πεδίου που θα χρειαζόταν. Είναι πολλέ οι προσπάθειε και καλέ, αλλά χρειάζονται ακόμη περισσότερε προσπάθειε από την κυβέρνηση ώστε να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα εθνοτικά ζητήματα ε, με μεγαλύτερη ευαισθησία. Η αποκέντρωση επίση. Έχουν σημειωθεί πολλέ προόδοι, αλλά χρειάζονται ακόμη περισσότερε προσπάθειε για να ε, χτίσουμε πάνω στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί και τι τοπικέ αρχέ να εξασφαλίσουν του πόρου που χρειάζονται για να διαχειριστούν και τι νέε του αρμοδιότητε. Και άλλο ένα σημαντικό ε, πεδίο της ε, Συμφωνίας Πλαισίου της ε, Οχρίδας είναι η ισότιμη εκπροσώπηση, όπου σημειώνεται καλή εξέλιξη, καλή προόδος προς την εκπροσώπηση και των αλβανόφωνων στους κρατικούς θεσμούς, στα κρατικά θεσμικά όργανα, αλλά πολύ περιορισμένη πρόοδος ως προς την εκπροσώπηση των τουρκόφωνων και των Ρωμά. Πρόοδο υπάρχει, χρειάζεται ακόμη περισσότερη προσπάθεια. Δυστυχώ είχαμε κάποιο οπισθοδρόμηση του τελευταίους μήνες και παρακαλούμε την κυβέρνηση να φροντίσει ώστε να μην συνεχιστεί αυτή η οπισθοδρόμηση, αυτή η διολίστηση. Σημαντική νομοθεσία ε, και ευρωπαϊκή που είχε να κάνει με τα ύδατα έχει καθυστερήσει επί τέσσερα χρόνια, πρέπει να έχει τεθεί σε εφαρμογή εφέτος, όμως ε, ως αποτέλεσμα αυτής δεν μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή ε, μια σειρά προγραμμάτων για διαχείριση αποβλήτων ε, και άλλα προγράμματα που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης περιμένουμε να εκδοθεί η νομοθεσία για την κατάληψη των διακρίσεων, την απαγόρευση των διακρίσεων και άλλη σχετική νομοθεσία. Μεγάλο πρόβλημα παραμένει η ουσιαστική υλοποίηση, εφαρμογή της νομοθεσίας και για να επιτύχει αυτή χρειάζονται ακόμη περισσότερες προσπάθειε και ως προς την αποκέντρωση της δημόσιας διοίκησης, γιατί ακριβώς εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα ε, στην δημόσια διοίκηση, η οποία καθοδηγεί τη διαδικασία της εφαρμογής νομοθεσίας. Επίσης μεταρρύθμιση στην αστυνομία έχει μεγάλη σημασία, έχει μεγάλη, μεγάλο πρόβλημα αξιοπιστία στην αστυνομία. Σχετική με αυτή είναι η μεταρρύθμιση του σοφρονιστικού συστήματος που ελπίζουμε ότι θα προχωρήσει με βάση και τα, ε, τις συστάσεις ε, της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την απαγορεύση των βασανιστήριων. Ε, χρειάζονται επιπλέον εντατικέ ε, προσπάθειε για την καταπολέμηση τη διαφθορά, έτσι ώστε να βελτιωθεί το επιχειρησιακό περιβάλλον, το επιχειρηματικό περιβάλλον και να ε, μπορέσουν να έρθουν στη χώρα περισσότεροι επενδυτέ και επενδύσει. Και επιπλέον θα ήθελα, Πρόεδρε, να σημειώσω ότι χρειάζονται σημαντικέ προσπάθειε από την κυβέρνηση στη χώρα Ω προ τη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, προ το συμφέρον τη χώρα, και πρέπει να το αντιληφθούν αυτό, ότι θα πρέπει να επιτραπεί η συνεργασία τη κοινωνία των πολιτών σε δικασία λήψεων αποφάσεων σε κάθε επίπεδο και εν τέλει θα πρέπει να αναφερθώ και στην ελευθεροτυπία, στην ανεξαρτησία των μέσων μαζική ενημέρωση, γιατί υπήρχε σαφή προσπάθεια και σαφή δυνατότητα παρέμβαση στα μέσα μαζική ενημέρωση, ενώ θα πρέπει να επιδιώξουμε πιστόρια διαφάνεια μεταξύ της ε, ε, ως προς τη σχέση της κυβέρνησης και των ΜΜΕ, να μην υπάρχει δηλαδή διαπλοκή και να εξασφαλιστεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης ε, αμφωτέρωθεν. Μεγάλε προκλήσεις προκλήσει λοιπόν για τη χώρα, Πρόεδρε. Θα πρέπει να σταθεί και να χτίσει πάνω στι επιτυχίε του 2009, να διατηρήσει την ορμή των μεταρρυθμίσεων και βεβαίω η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο πλευρό του για να του στηρίξει με όλα αυτά τα προγράμματα που έχει, αναπτύξει. Ε, εν τέλει όμω, ε, όσε προσπάθειε και να κάνουμε εμείς τελική επιτυχία θα εξαρτηθεί από την ίδια την κυβέρνηση. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ. Να δώσω τον λόγο τώρα στον συνάδελφο Τάλερ που είναι η σου. το ψήφισμα του Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην πρώην Ιουκλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Παρακαλώ να παραμείνετε εντό των τριών-τεσσάρων λεπτών κατά νότα τον όριο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε εκπρόσωπε, για την εκπαιδευτική εργασία σας και για το έργο που κάνετε στην ε, πρώην ε, Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Νομίζω ότι όλοι βρισκόμαστε στο ίδιο σκάφος. Πού στοχεύουμε. Στοχεύουμε σε κάποιες θετικές ε, εξελίξεις και βελτιώσεις στην περιοχή. Αργότερα θα έχω τη δυνατότητα να πω κάποια πράγματα αναφορικά με το ψήφισμα, το οποίο βρίσκεται προς συζήτηση σήμερα στην Επιτροπή μας. Θα επικεντρωθώ τώρα σε κάποιες ερωτήσεις προς εσάς. Πού βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει δυνατότητα για περαιτέρω εξελίξεις μεταξύ, στους, μεταξύ των διηγητών, δηλαδή της Ελλάδας και της ε, πρώην ε, Ιουγκραβική Δημοκρατία Μακεδονίας. Η Ελλάδα είναι μέλος ε, και η ουκρανική Δημοκρατία είναι υποψήφιο μέλος. Τον φθινόπωρο είχαμε νέες εκλογές ε, στην Ελλάδα, εξελέγησε η κυβέρνηση και υπήρξαν κάποιες θετικέ εξελίξεις. Ε, προηγούμενα δεν είχαν υπάρξει άμεσες επαφές, ε, είχαν διακοπεί. Νομίζω ότι η σχέση τώρα ανάμεσα στους δύο πρωθυπουργούς είναι πολύ καλύτερη. Πώς βλέπετε λοιπόν αυτό το θέμα των σχέσεων μεταξύ μιας υποψήφιας χώρας και μιας χώρας μέλους. Γίνεται τίποτα σε επίπεδο οικονομικής συνεργασίας, πολιτικής συνεργασίας, διαστορικής συνεργασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τάλερ. Ο συνάδελφος Πόστελτ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι ο συνάδελφος Τάλερ έχει καταρτήσει μια πολύ καλή και ισορροπημένη έκθεση και ήταν πολύ ενδιαφέρουσε οι δηλώσει του κυρίου Φουέρε. Αλλά θα ήθελα να του θέσω και μία ερώτηση. Είπε ότι η συνθήκη για τα βασανιστήρια δεν έχει εφαρμοστεί πλήρω. Θα ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει κάποια συγκεκριμένη παραβίαση, μπορεί να μα αναφέρει κάποια συγκεκριμένη παραβίαση και επίση να συνηγορήσω υπέρ της δικαιοσύνης. Είπατε ότι εξαρτάται από την κυβέρνηση της Μακεδονίας λέει ο να αναρρυθμίσει το θέμα αυτό. Όμως το θέμα του ονόματος εξαρτάται από δύο πλευρές και έχει υποβάλει πολλές προτάσεις η Μακεδονία, οι οποίες έχουν, δεν έχουν γίνει αποδεκτές. Χρειάζονται λοιπόν να συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές. Και θα ήθελα να πω με σαφήνεια ότι υπάρχει μια ενδιάμεση συμφωνία βάσει των διμερών μάλλον που δεν επιτρέπονται να εφαρμοστεί βάσει των ε, διαφωνιών. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτή η ενδιάμεση συμφωνία και να μην βρεθούμε όμοιροι ενός διμερούς ε, ζητήματος και σε ό,τι αφορά τις μειονότητες. Όλες οι μειονότητες εκπροσωπούνται στην κυβέρνηση. Ξέρω πολύ καλά τη χώρα. Μίλησα με όλες τις ε, μειονότητες που εκπροσωπούνται και αν όλε. Ε, οι... Θα ήμασταν πολύ ευτυχεί αν όλε οι κυβερνήσει είχαν την ίδια εκπροσώπηση μειονοτήτων στην κυβέρνηση όπω η Μακεδονία. Η κυρία Κοπά έχει το λόγο δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Φουερέ για την παρουσίασή του, αλλά και τον εισηγητή τον κύριο Τάλερ για το αρχικό του κείμενο που είναι αρκετά ισορροπημένο. Ε, θα ήθελα να κάνω απλώ κάποιε παρατηρήσει πάνω στι συμβιβαστικέ τροπολογίε. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση, με το που ανέλαβε πριν από 100 περίπου μέρες, πήρε πρωτοβουλίες για να ξαναρχίσει ο διάλογος στα Ηνωμένα Έθνη και οι απευθείες επαφές των δύο πρωθυπουργών, πάλι με ελληνική πρωτοβουλία, που ήρθαν να υποστηρίξουν τη διαδικασία αυτή στα Ηνωμένα Έθνη, έδειξαν ότι μπορούσε να υπάρχει ένα breakthrough. Αυτό δεν επιβεβαιώθηκε πριν τη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου. Ε, η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να εργάζεται για εξέβρεση λύσης, όπως έκανε από τη στιγμή που ανέλαβε η κυβέρνηση αυτή την εξουσία. Για όλους μας πάντως το πλαίσιο παραμένει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Γι' αυτό και μόλις χθε ο αναπληρωτής Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας ζήτησε από το διαμεσολαβητή κ. Νίμιτς να επισκεφτεί τις επόμενες μέρες στην Αθήνα για να ξαναρχίσει εντατικά ο διάλογος. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι για το λόγο αυτό θα ήταν επιθυμητό το μόνο συμφωνημένο πλαίσιο που είναι ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών να αναφέρεται στις συμβιβαστικές τροπολογίες 4 και 5. Είναι παράλληλα άδικο να γίνεται σύσταση σε γειτονικέ χώρες όπως στη συμβιβαστική 5, ε, σύσταση να αποφεύγουν πράξεις και δηλώσεις που αρνητικά επηρεάζουν την καλή γειτονία. Κύριε Πρόεδρε, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και από όσο γνωρίζω και τη Βουλγαρία, ούτε η μία ούτε η άλλη χώρα δεν έχουν δώσει δείγματα γραφής ε, ρητορικής μίσους, ε, ρητορικής αναφοράς στην αρχαιότητα, τουλάχιστον το πρόσφατο παρελθόν, που να δικαιολογούν μια τέτοια αναφορά στην έκθεση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Κάτσιν, δύο λεπτά. Ε, ευχαριστώ πρόεδρε και καλώς ορίσατε κύριε Φουέρε και σας συγχαίρω για το έργο σας ε, στα Δυτικά Βαλκάνια. Δεν έχω υπόψη μου μόνο τη Μακεδονία μιλώντα ε, για το έργο σας, αλλά και το προηγούμενο έργο σας για τη Σλοβενία. Εμπιστεύομαι λοιπόν τι ικανότητε σα. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν συναισθηματικά προβλήματα, τα οποία επί σειρά ετών αποτελούσαν και την πηγή του θέματος, του μπλοκαρίσματος αν θέλετε, που επικρατούσε για το θέμα της ονομασίας. Η Μακεδονία είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία, αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε ότι πολλά βρίσκονται ακόμα στα χέρια του κ. Γκρουέτσκι, του Πρωθυπουργού. Ερωτώ λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε στο σημείο αυτό για να ενισχύσουμε το ρόλο της Ρομπράνια, του Κοινοβουλίου της Μακεδονίας. Πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε τους ε, βουλευτές να επιτύξουν μεγαλύτερη ευελιξία για τη συντελική ανάλυση. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε κάποια, κάποιο συμβιβασμό. Θα ήθελα να πω ότι τακτικά οι βουλευτές της Μακεδονίας επισκέπτονται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά σε τελική ανάλυση θα είναι μεγάλη η απόφαση που θα, ληφθούν, που θα κληθούν να πάρουν και θα χρειαστούν την υποστήριξή μας. Το δεύτερο θέμα που ανακύπτει είναι ότι το Κοινοβούλιο της ε, Μακεδονίας και του Μαυροβουνίου έχουν εγκρίνει το ψήφισμα του Κοινοβουλίου του Ευρωπαϊκού για τη Σρεμπρενίτσα. Αλλά αυτό δεν συνέβη στο Κοινοβούλιο της ε, Μακεδονίας, μόνο της Κροατίας και του Μαυροβουνίου. Και όταν μίλησα με τους βουλευτές, ε, μου είπαν ότι μου δόθηκε εντύπωση ότι φοβόντουσαν τις ε, Αντιδράσει του Βελεγραδίου. Πώ μπορούμε λοιπόν να ενισχύσουμε του συναδέλφου μα στο Μακεδονικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Το λόγο για δύο λεπτά έχει ο κ. Σαλαβράκος. Κύριε Πρόεδρε, ε, άκουσα τον κύριο Φουαρέ με μεγάλη προσοχή και συμφωνώ σε πολλά από αυτά τα οποία λέει, όπως συμφωνώ βεβαίως και με την έκθεση του κ. Τάλλα σε πολλά σημεία. Βεβαίως δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι πληρούνται τα κριτήρια της Κομεχάγης για την ένταξη αυτής της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως συμπαθώς βλέποντας αυτή τη χώρα δεν θα μπορούσαμε και να αρνηθούμε ότι θα πρέπει να την υποβοηθήσουμε να γίνει μέλος της Ενωσεώ μας. Να την υποβοηθήσουμε όμως με τα δεδομένα εκείνα τα οποία εξασφαλίζει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών με την κουβέντα την οποία γίνεται και τη διαπραγμάτευση που γίνεται μέσα σε αυτόν με τη διαμεσολάβηση του κ. Νίμιτς σε σχέση με το όνομα ε, της υποψήφιας αυτής χώρας. Ο κύριος Φουαρέ ανέφερε ότι υπήρξε το πρόβλημα μιας αμφιλεγόμενης εγκυκλοπαίδειας. Η αμφιλεγόμενη αυτή εγκυκλοπαίδεια λοιπόν, την οποία πρέπει και τον παρακαλώ να αναλύσει, για να λάβουν ε, υπόψη τους όλα τα μέλη της Επιτροπής το τι λέει, λέει ότι πέραν του ονόματος υπάρχει αλυτρωτισμός ε, για τη χώρα αυτή και επεκτατικές βλέψεις στην Ελλάδα και ότι η πρωτεύουσα της χώρας αυτής πρέπει να είναι η Θεσσαλονίκη, η οποία είναι η δεύτερη σε πληθυσμό χώρα της Ελλάδος. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πυροδοτείται από αυτή την αμφιλεγόμενη, όπως είπε ο κ. Σουαρή, ένα κλίμα κακής γειτονία το οποίο προέρχεται από την πλευρά της ε, υποένταξη αυτής της χώρας, της Φύρου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τα προβλήματα τα οποία έχει αυτή η χώρα και κατά πόσον θα πρέπει να βάλει λίγο νερό στο κρασί τη ως προς την πραγματικότητα. Ερωτάτε λοιπόν, ε, παρακαλώ ε, κύριε Φουάρε, αναλύσατε το τι λέει αυτή η εγκυκλοπαίδεια, πείτε μας σας παρακαλώ εάν έχετε πληροφορίες για τυχόν θετική εξέλιξη για την, από την διαμεσολάβηση του κ. Νίμης, ε, και θα παρακαλούσα επίσης να μου πείτε εάν υπήρξε ενημέρωση της κοινή γνώμης σε σχέση με την καλή θέση των Ελλήνων Ευρωβουλευτών ε, για την ελευθεροκίνηση των ε, κατοίκων της Φύρου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σαλαβράκο Να δώσω το λόγο στον ειδικό εκπρόσωπο για 5-6 λεπτά. Παρακαλώ. Ε, Σας ευχαριστώ πρόεδρε και σας ευχαριστώ και για τις ερωτήσεις που μου θέσατε. Θα απαντήσω με τη σειρά που τις θέσατε. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τον κύριο Τάλερ, θεωρώ ότι υπάρχει ανάγκη να ενισχυθούν οι διμερείς σχέσεις εμπιστοσύνη σε δύο επίπεδα. Σε πολιτικό επίπεδο που έγιναν οι δύο συναντήσεις μεταξύ πρωθυπουργών, οι οποίες συνέβαλαν στο να σπάσει ο πάγος, αν θέλετε, και να δημιουργηθεί ένα πιο θετικό κλίμα και θεωρούμε ότι περισσότερες συναντήσεις τέτοιου τύπου θα βοηθήσουν. Σε τοπικό επίπεδο τώρα υπάρχει πραγματικά ανάγκη να βελτιωθεί η συνεργασία. Και έχουμε κάποια εξαιρετικά παραδείγματα επαφών μεταξύ των λαών, μεταξύ ελληνικής πλευράς και από πλευρά τη πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία. Έχω επισκεφτεί πολλά τέτοια προγράμματα, project που αφορούν πολιτισμικά ζητήματα, που έχουν ως στόχο να προσεγγίσουν οι τοπικές κοινωνίες και έχουμε πλέον νέα προγράμματα. Θα υποβληθούν νέες προτάσεις Είχαμε κάποιε καθυστερήσει, πρέπει να παραδεχτώ από ελληνική πλευρά και καλούμε την κυβέρνηση, καλέσαμε την κυβέρνηση να επιταχύνει τι διαδικασίε αυτέ. Και νομίζω ότι πραγματικά αυτό είναι σημαντικό γιατί μιλάμε και για χρήματα και θα ήταν πραγματικά σημαντικό να αναπτυχθούν τέτοιε πρωτοβουλίε. Τέτοιε πρωτοβουλίε ε, αναπτύσσονται και με τη Βουλγαρία και την Αλβανία. Αυτέ οι επαφέ μεταξύ των λαών επηρεάζουν ιδιαίτερα την οικοδόμηση εμπιστοσύνη σε τοπικό επίπεδο. Τώρα, να απαντήσω στον κύριο Πόσελτ δεν υπάρχουν ε, αν θέλετε, παραβιάσει συγκεκριμένε της ε, Συμφωνίας πλαισίου της Οχρίδας. Πρόκειται, μιλά πιο πολύ για μια ανατροπία που δεν συνάδει ίσως με την ε, συμφωνία πλαίσιο της Οχρίδας. Ερώτηση εκτό μικροφώνου. I spoke ο κύριος Πόσελτ μίλησα για την ε, συνθήκη για τα βασανιστήρια του Συμβουλίου της Ευρώπης και ρώτησα αν γνωρίζετε κάποια συγκεκριμένη περίπτωση παραβίασης της συνθήκης. Όχι, ναι, συγγνώμη. Σε ό,τι αφορά τα βασανιστήρια έγιναν πολλές συστάσεις σε ό,τι αφορά την πρόληψη βασανιστήριων από το 2007, οι οποίες δυστυχώς δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμη. Έχω επισκεφτεί φυλακές και έχω δει ποιες είναι οι φρικτέ συνθήκε που επικρατούν. πώς ζουν οι φυλακισμένοι και υπάρχει δέσμευση ε, από πλευρά της κυβέρνησης, αλλά έχουν καθυστερήσει σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των συστάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Για να απαντήσω στην κυρία Κοπά. Ερώτηση εκτός μικροφώνου. Δεν μπορώ να απαντήσω καταφατικά στο, στην ερώτηση αυτή. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ερώτηση της κυρίας Κοπά. Φυσικά, η διαδικασία Νίμιτς αποτελεί την επίσημη διαδικασία η οποία έχει δημιουργηθεί, ιδρυθεί από την συμφωνία, από την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για το θέμα της ονομασίας. Και αυτό εξακολουθεί να ισχύσει. Θεωρούμε όμως ότι οι δημερείς επαφές θα συνδράμουν, θα συμβάλλουν αν θέλετε, θα αποτελέσουν έναν επιπρόσθετο παράγοντα για να δοθεί περαιτέρω όθεση και ελπίζουμε οι διμερείς ε, επαφές που ξεκίνησαν το φθινόπωρο θα συνεχιστούν. Και όταν ο κύριος Νίμιτς ε, μεταβεί στην περιοχή θα τον βοηθήσουν. Γιατί πραγματικά αυτό που χρειάζεται είναι μια σαφής συνεχιζόμενη προσπάθεια από αμφότερες τις πλευρές για την εξέβρεση λύσης και φυσικά και ο Νίμιτς θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην όλη διαδικασία. Για να απαντήσω τώρα στον κύριο Κατσίν. Χαιρόμαστε που υπάρχει σύμφωνη για την ε, δημιουργία κοινοβουλευτικών θεσμών με την βοήθεια των Τσέχων ε, και με τη βοήθεια των εθνικών θεσμών και αυτό προφανώς θα δώσει μεγαλύτερο ρόλο στο Κοινοβούλιο για τη Σρεμπρένιτσα. Σύμφωνο απόλυτα μαζί σας, θα πρέπει να υπάρξει και να καταβληθεί τεράστια προσπάθεια από όλες τις χώρες για τη συμφιλίωση. και δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να ανησυχούμε από πλευράς ε, του Κοινοβουλίου των Σκοπίων σε ό,τι αφορά ενδεχόμενη αντίδραση της Σερβίας, γιατί μιλάμε για τη συμφιλίωση όλης της περιοχής και δυστυχώς η κυκλοπαίδη αυτή αποτέλεσε ένα θέμα, γιατί έθεσε σε αμφισβήτηση πολλά θέματα της Συμφωνίας Πλαισίου της Οχρίδας και δημιούργησε, αν θέλετε, ένα κλίμα προκατάληψης. Προκατάληψης που εξακολουθεί να επικρατεί και η κυβέρνηση α, διατήρασε αποστάσεις από την εγκυκλοπαίδεια, αλλά αυτό καταδεικνύει ότι υπάρχουν ακόμα τεράστιος όγκος ε, δουλειάς που πρέπει να γίνει προκειμένου η περιοχή να πετύχει τη συμφιλίωση. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια προς την κατεύθυνση της συμφιλίωση. και να αναφέρω πάρα πολύ να επιβεβαιώσετε τι λέει η εγκυκλοπαίδη αυτή για να καταλάβουν. Ε, παρακαλώ, παρακαλώ. Συγγνώμη, αλλά εδώ δεν κάνουμε διάλογο. Ας αφήσουμε να ολοκληρώσει την απάντησή του και δεχόμενα ζητάτε το λόγο εκ των υστέρων. Ναι. Να διευκρινίσω ότι είμαι βέβαιο ότι εσεί γνωρίζετε καλύτερα ότι παρά το γεγονό ότι υπάρχουν πλαίσια για τη συνεργασία, για την προώθηση των ε, πολυεθνικών ε, συνεργασιών, ποτέ κανεί δεν μπορεί να πάρει δεδομένα μερικά πράγματα στα Βαλκάνια. Προφανώ θα πρέπει να ενισχυθεί το κλίμα εμπιστοσύνη και να αναπτυχθεί το ο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Το λόγο έχει ο κ. Κούκαν, πρόεδρος αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με την Ανατολική Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και για την παρουσία εδώ του κύριου Φουερέ και το έργο του και την αφοσίωση του στο έργο του. Όσον αφορά το ψήφισμα προ την έκθεση πρόοδου για τη ΦΥΡΟΜΑ. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Τάλερ για το σχέδιό του και να εκφράσω την εκτίμησή μου για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την επεξεργασία του εγγράφου. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα στους συναδέλφους που ε, ενεργοποιήθηκαν και ε, υπέβαλαν, δραστηριοποιήθηκαν μάλλον και υπέβαλαν τροπολογίες. Είναι μια καλά ισορροπημένη έκθεση αυτή και προτείνω να την υποστηρίξουμε. Οι δικές μου τροπολογίε είναι σε ευθεία γραμμή με τις προτάσεις του εισηγητού στο μέγιστο βαθμό. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. ω προς τα θετικά, καταρχάς όντως είδαμε πρόοδο σημαντική από την ΦΥΡΟΜ ε, πέρυσι και προχωρεί στην τήρηση των κριτηρίων για την συνέχιση των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. πρόκειται για την οικονομική ε, ανοικοδόμηση, τις προϋποθέσεις για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω επίση να υπογραμμίσω την επιτυχία τη χώρα ω προ την επίτευξη των οροσίμων για την απελευθέρωση του συστήματο των θεωρήσεων διαβατηρίων. Η εκείνη των διαπραγματεύσεων για την ένταξη, όπω αποφασίστηκε, είναι μια θετική εξέλιξη, πιστεύω, και θα πρέπει να ξεκινήσει στο, εγγυσμένο. Ως προς τα αρνητικά στοιχεία, υπάρχουν ακόμη κάποια σημεία στα οποία περιμένουμε περισσότερες προσπάθειες και πρόοδο ειδικότερα στον τομέα της δικαστικής ε, εξουσίας της δημόσιας διοίκησης, μεταρρύθμιση δηλαδή της δικαιοσύνη και της δημόσιας ε, διοίκησης, την αντιμετώπιση της διαφθοράς, ε, τη συμπερίληψη όλων των μειονοτήτων στο δημόσιο βίο, την απαλλαγή από τη διαπλοκή των ΜΜΕ, ανεξάρτητα ΜΜΕ και θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τη χώρα να συνεχίσει σε αυτέ τι τάσει που ήδη είναι θετικέ. Θα ήθελα να υπογραμμίσω λοιπόν την ανάγκη να υποστηρικτούν όλε αυτέ οι τροπολογίε που πηγαίνουν προ το στόχο αυτό και τι συμβαστικέ τροπολογίε που έχουμε συντάξει σε συνεργασία με τον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Κούκαν. Ο κύριο Κυρίλοφ έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πρέσβη. Ξέρετε ότι ήταν πολύ σοβαρό το πρόβλημα εκείνο το οποίο οδήγησε σε πολλές αντιδράσεις ε, στην Βουλγαρία, την γειτονική Βουλγαρία. Μια μητέρα με, το, με μωρό που θύλαζε τριών μηνών μπήκε στη φυλακή γιατί υποτίθεται αρνήθηκε να επιτρέψει στον διαστάσει σύζυγό της να μείνει στο ίδιο σπίτι μαζί της. Υποτίθεται ότι δεν τον άφηνε να δει το παιδί. Ωστόσο, αυτό ήταν η πρόφαση, αυτό που προβλήθηκε στα μέσα μαζική ενημέρωση. Ε, το πρόβλημα ήταν άλλο όμω ότι η γυναίκα αυτή είχε αποκτήσει ε, μερικούς μήνες πριν τη βουλγαρική υπηκότητα και αισθανόταν ω υπήκο τη Βουλγαρία. Αυτό δεν είναι μόνο μονομένη περίπτωση. Είχαμε πολλά προβλήματα. Είπε το καθεστώς ε, του Τίτο είχαν πολύ χειρότερη μεταχείριση οι άνθρωποι αυτοί. του έστελναν στα στρατόπεδα συγκεντρώσεω. Γιατί λοιπόν ε, αναφέρομαι στην περίπτωση αυτή. Γιατί όλοι οι ενδιαφερόμενοι από τη Βουλγαρία απέστειλαν επιστολή στον κύριο Όλι Ρεν και ε, τρεις μήνες πριν εκπνεύσει η προθεσμία των τριών μηνών ε, απελευθερώθηκε η γυναίκα αυτή από τη φυλακή, αποφυλακίστηκε, που όμως δεν της έχει ακόμη επιτραπεί να δει το μωρό της. Μιλάτε λοιπόν για τη σχέση μεταξύ Βουλγαρίας και Μακεδονίας. Από πότε κύριε πρέσβη τέτοιου είδους παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι ζήτημα μόνο διμερών σχέσεων. Εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τέτοιου είδους παραβιάσεις δεν τις αντιμετωπίζουμε με τέτοιο τρόπο. Από πού σας ήρθε σας αυτό και πώς είναι δυνατόν. Ναι, θέλετε να παρέμβετε, εντάξει, δεν θέλετε να κάνετε δήλωση, πολύ καλά. Αλλά τουλάχιστον δείτε το ως ένα σοβαρό πρόβλημα των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Αυτή η γυναίκα ακόμη δεν έχει δει το κοριτσάκι της. Ο κύριος Κορνέλησεν, δύο λεπτά. Η κυρία Κορνέλισεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ξεκινήσουμε με το ζήτημα της ονομασίας. Νομίζω όλους μας απασχολεί. Φυσικά πρέπει να βρεθεί λύση. Η εθνικιστική ορολογία που χρησιμοποιείται και από τις δύο πλευρές θα πρέπει να σταματήσει και πρέπει να κοιτάμε το μέλλον και όχι το πολύ απότερο παρελθόν. Ωστόσο, δεν μπορεί αυτό να αποτελέσει προϋπόθεση για την ένταξη. Η εξέβρεση λύση στο όνομα δεν μπορεί να αποτελέσει προπόθεση για την ένταξη, όπως φαίνεται ότι νομίζουν ορισμένοι τώρα. Και δεν μιλάμε μόνο για αυτή την υπόθεση, δεν ισχύει μόνο αυτή την υπόθεση, ισχύει και για την Ελλάδα βέβαια ω προς τη Μακεδονία, αλλά και για τη δική μου τη χώρα, την Ολλανδία, ω προ τι κατοχώρε ω προ την Ισλανδία, αλλά και τη Σερβία ή την Κύπρο σε σχέση με την Τουρκία. Ελπίζω όλες αυτές οι χώρες να ακολουθήσουν το αξιέπαινο, αξιέπαινο παράδειγμα της Σλοβακίας, η οποία εξομάλυνε τις σχέσεις με την Κροατία και έως εκ τούτου δεν υπάρχει πλέον ε, εμπόδιο προς τη Σλοβακία για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Κροατίας. Θα παρακαλέσω λοιπόν τους πάντες να κάνουν δεκτή τροπολογία παριθμών 57 που έχουμε υποβάλει, η οποία ορίζει ότι διμερεί ζητήματα θα πρέπει αυτά καθεαυτά να αποτελούν πρόσκομα στην πρόοδο προς την ένταξη. Τούτων λεχθέντων θα ήθελα να προχωρήσω σε άλλα θέματα, πολύ σημαντικά. Κατά την άποψή μου, η επιτυχία μιας χώρας, η οριμό μιας χώρας προσμετράται από τον τρόπο με τον οποίο μεταχειρίζεται τους πιο ευάλωτους πολίτες της. Τους Ρωμά, παραδείγμα. Τις γυναίκες πέφτουν θύματα της βίας, παραδείγματι. Πρόοδος, ναι, έχει επιτευχθεί. Θα ήθελα όμως περαιτέρω εφαρμογή των σχεδίων που έχουν διατυπωθεί και θα ήθελα η νομοθεσία που αφορά την κατάρριξη των διακρίσεων να εγκριθεί και να προσφερθεί υποστήριξη κυρίως με τη μορφή των ένδικων μέσων ή βοηθμάτων σε όποιους έχουν υποστεί τέτοιου είδους διακρίσεις. Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια. Έχει λήξει ο χρόνος σας, κύριε Κορνέλ, κύριε έχει το λόγο. Πρόεδρε, και ευχαριστώ τον κύριο Φουέρα για τις αναφορές του. Ήθελα να σημειώσω τα εξής ως προς τις συμβιβαστικές τροπολογίες καταρχήν. Ε, οι συμβιβαστικές τροπολογίες 4 και 5 δεν αντανακλούν στις τροπολογίες ε, από τις οποίες υποτίθεται ότι προέρχονται. Ιδιαίτερα στην 4, όπου αναφέρεται η επαφή μεταξύ των δύο πρωθυπουργών, δεν αναφέρεται ότι η συνεννόηση αυτή τη στιγμή γίνεται υπό την ε, αιγίδα και την ευθύνη των Ηνωμένων Εθνών και του ειδικού διαμεσολαβητή του κυρίου Νίμιτ. Πρέπει να αναφερθεί. Στην ε, τροπολογία 3 συμβιβαστική, ο ποταμός Βαρντάρ λέγεται αξιός από την πλευρά της Ελλάδος και πρέπει να αναφερθεί. Στη δε τροπολογία 5 ουδέμια σχέση έχει η συμβιβαστική με τις τροπολογίες από τις οποίες προέρχεται. Οι τροπολογίες από τις οποίες προέρχεται λένε τελείως διαφορετικά πράγματα από τη συμβιβαστική. Τούτα αυτό συμβαίνει με τις τροπολογίες του εισηγητού 67 ε, και 58. Δηλαδή άλλα πράγματα έλεγε η βασική έκθεση, σχολίαζε την επιθετικότητα που υπάρχει ε, και τις ε, διάφορες προπαγανδιστικές ρίσεις από πλευράς της ΦΥΡΟΜ και εδώ έχουμε φτάσει να καθιστούμε υπεύθυνε τις χώρες οι οποίες είναι γειτονικέ για ό,τι συμβαίνει στη ΦΥΡΟΜ. Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση αυτή δεν αντανακλά την πραγματικότητα η οποία υπάρχει και εγώ καλώ τον ίδιο τον εισηγητή να επανέλθει στην αρχική του εισήγηση. Δεν αντιλαμβάνομαι πώς έχει διαστραφεί η αρχική εισήγηση του εισηγητού και εμφανίζεται να λέει ότι οι χώρες που είναι γειτονικέ είναι υπεύθυνε αν δεν εισέλθει ταχύτατα η φύρομ στην Ευρωπαϊκή Ένωση διότι διαφορετικά θα δημιουργηθούν συγκρούσει μεταξύ εθνοτικών ομάδων. Από πότε κύριε Πρόεδρε τα προβλήματα τα εσωτερικά μιας χώρας και οι συγκρούσεις εθνοτικών ομάδων καθιστούν υπεύθυνε άλλες χώρες αν δεν κάνουν το χατήρι της χώρας αυτής η οποία έχει αναλάβει δέσμευση ως προς το όνομα Θέλω να τονίσω ότι το όνομα σαφέστατα είναι προϋπόθεση ένταξης, διότι δεν πρόκειται να γίνει δεκτό από την ελληνική κυβέρνηση η χώρα αυτή να γίνει μέλος χωρίς να διευθετηθεί η υπόθεση του ονόματος. Για δύο λεπτά Αγκουράκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και από την ε, τοποθέτηση του κυρίου Φουερέ αλλά και από, την, από το σχέδιο ψηφίσματος και από τις συζητήσεις που έχουμε κάνει σε αυτή την αίθουσα, ε, φαίνονται πραγματικά ότι γίνονται προσπάθειες στη γειτονική χώρα, δεν χωράει καμία αμφιβολία, για βελτίωση της κατάστασης και των σχέσεων ε, με γειτονικές χώρες. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Αυτό μας που με ανησυχεί, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν, είναι προφανές ότι υπάρχουν και αν ε, το πρόβλημα του ονόματος είναι ένα πρόβλημα που πρέπει, χρειάζεται να γίνουν προσπάθειες και από τις δύο πλευρές και εδώ υπάρχουν ε, ε, υπάρχει ανάγκη και ε, να συνεχιστούν οι προσπάθειες ε, γιατί είναι δυνατή να βρεθεί μια λύση. Εγώ άλλο ήθελα όμως να σημειώσω. Το είπε και ο κύριος Φουερέ για το ότι διαπίστωσε μια ένταση των διεθνωτικών αντιθέσεων, τριβών και στο θέμα του σχολείου το είχε πει και σε θέματα που έχουν σχέση με κάποιες μειονότητες κτλ. Η ερώτηση μου είναι εξής. Μήπω, κύριε ε, εκπρόσωπε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το ζήτημα αυτό έχει να κάνει με τα πραγματικά μεγάλα εσωτερικά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή η χώρα προβλήματα τα οποία αντανακλούνται και στο, σε αυτό που σημειώνεται στην έκθεση και εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω ότι αυτή πρέπει να είναι η προοπτική της χώρας ένα μεγάλο ποσοστό ανεργίας όπως λέει και επίσης σε μια παράδεκτη κατάσταση κατά τη γνώμη μου αν είναι έτσι όπως το σημειώνει η έκθεση όσον αφορά τα εργατικά συνδικαλιστικά δικαιώματα και τις διαδηλώσεις που έχουν γίνει στη γειτονική χώρα από γυναίκες εργαζόμενες ειδικά στην κλωστοϊφαντουργία που πραγματικά ε, νομίζω ότι υπογραμμίζουν την κατάσταση αυτή. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν δεν υπάρχει μια άλλη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη χώρα αυτή και αν δεν υπάρχουν απτυξιακές πολιτικές τότε είναι σίγουρο τα εθνοτικά προβλήματα θα εντάθουν. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Νέιτς για δύο λεπτά έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εξ ονόματος της αντιπροσωπείας μου θα ήθελα να υποβάλω μια προφορική τροπολογία σε αντικατάσταση του συναδέλφου, ε, των πρασίνων είναι κάτι το οποίο είχα παρουσιάσει στην Επιτροπή μας όταν συζητήσαμε το ζήτημα της διεύρυνσης. Δεν είναι κάτι το εντελώς καινούριο, απλά είναι επανάληψη κάτι ε, επί του οποίου έχουμε ήδη συμφωνήσει. Θα, θα το διαβάσω λοιπόν. Θέλουμε στο τέλος τροπολογίας 19 να πούμε τα εξής τονίζει πως ε, παρόμοιες ε, διμερείς ε, διαφωνίες θα πρέπει να επιλύονται από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Αν τυχόν δεν το καταφέρουν οι ενδιαφερόμενοι, τότε η Ένωση θα πρέπει να καταβάλει προσπάθειες προκειμένου να εξευρεθεί λύση. εάν παρόμοιες διαφωνίες από μόνες δεν αποτελούν πρόοδο στην ένταξη, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μην αναμειχθεί με παρόμοιες διενέξεις, αλλά αυτές να επιληθούν ε, εγκαίρως. Είναι εύκολο να πούμε ότι παρόμοιες ε, διαφορές δεν αποτελούν εμπόδιο στην ε, ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν πιστεύω θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου να αρθούν παρόμοια εμπόδια. Ευχαριστώ. Bene, questa nostra riunione prevede η συνεδρία αυτή προβλέπει έναν συνομιλητή, τον κύριο Φουαρέ. Τώρα, εάν εσείς ε, κύριε Τάλερ θέλετε να απαντήσετε σε δύο-τρεις ε, ερωτήσεις που αφορούν τροπολογίες, θα σας δώσω δύο λεπτά χρόνο για να απαντήσετε και παρακαλώ είστε σύντομος. Ευχαριστώ. Πιστεύω πως ε, το ψήφισμα έχει σημαντικά βελτιωθεί. Έχουμε εδώ δημιουργήσα ένα επικοδομητικό κλίμα ανάμεσα σε όλες τις πολιτικές ομάδες πάνω στο ζήτημα και χαίρομαι γι' αυτό. Σε τι στοχεύουμε. Στοχεύουμε πρωτίστως να ενθαρρύνουμε την Μακεδονία να συμμορφωθεί με τις ε, ευρωπαϊκές αρχές. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να επιτευχθεί πρόοδος και τους ενθαρρύνουμε να αναλάβουν πιο φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις ε, σε όλους τους τομείς και επίσης να εξευρεθεί μια λύση στο ζήτημα της ονομασίας. Αυτό αναφέρεται ρητά στο ψήφισμα και στις τροπολογίες. Επίσης, στοχεύουμε να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας πως είμαστε υπεύθυνοι για τις θετικές αλλαγές στην περιοχή, για την ειρήνη, την οικονομική και κοινωνική πρόοδο, την σταθερότητα. Θα πρέπει λοιπόν να απογνωρίσουμε ότι το θέση όπως το διατήρηση status quo κλπ. δεν είναι ε, θέση ουδέτερη. Η διατήρηση του status quo είναι κάτι το αρνητικό, διότι τα Δυτικά Βαλκάνια είναι σαν το ποδήλατο. Όσο προχωρούν, εντάξει προς την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει πρόοδο Κρατάνε ισορροπία. Εάν όμως σταματήσει την πορεία του, τότε το ποδήλατο πέφτει. Έτσι και τα Δυτικά Βαλκάνια. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να φροντίσουμε να, διατηρήσουμε, να διατηρηθεί η πορεία του ποδηλάτου προς την ευρωπαϊκή πλευρά. Τώρα, όπου κατέστη δυνατόν, εγώ υποστήριξα κάποιες τροπολογίες εφόσον πηγαίνουν προς ε, αυτή την προς αυτή την ε, πορεία. Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες ε, που θα μπορούσαν νομίζω να βελτιωθούν, αλλά εν αυτό είναι θέμα της αυριανής συνεδρίασης όπου και θα ψηφίσουμε. Προσβλέπω λοιπόν ότι όλοι μαζί κάναμε μια εξαιρετική εργασία όλα τα κόμματα. Ας τη συνεχίσουμε λοιπόν. Κύριε Σιγητά, επειδή ε, θίγησαν κάποια ζητήματα περί του θέματος αυτού, το ζήτημα της, ε, των διμερών διαφωνιών και της παρεμπόδισης ε, κλπ. Θα ήθελα να μας διευκνήσετε ποια είναι η άποψή σας περί αυτού. Κοιτάξτε, αναφέρεται ρητά και στο κείμενο ότι υποστηρίζουμε την εξέβρεση αμοιβαίας αποδεκτής λύσης. Διμερός δηλαδή, να εξευρεθεί μια λύση στο ζήτημα του ονόματος. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κείμενο ότι τέτοιου είδους, το θέμα του ότι τέτοιου είδους διαφορές δεν θα πρέπει να παρεμποδίζουν την ένταξη, την προσφόρηση μια χώρας, δεν συμφωνώ απόλυτα με το προτινόμενο κείμενο, αλλά εν θα ψηφίσουμε περί αυτού. Και κάτι ακόμα. Αυτό μπορεί να αποτελέσει και μια δικαιολογία προκειμένου να μην επενδύσουμε περισσότερες προσπάθειες για την επίλυση αυτών των διμερών προβλημάτων που αναφίβολα παρεμποδίζουν κάποιες διαδικασίες εδώ και χρόνια. Ευχαριστώ για την διευκρίνηση που μας κάνατε, κύριε Σιγητά. Σας καλώ λοιπόν να βρείτε ένα συνενετικό κείμενο. Σας αφαιρέσαμε χρόνο, κύριε Φουερέ, αλλά έπρεπε να μοιράσουμε την ώρα αυτή μεταξύ ημών και του εισηγητή. Έχετε το λόγο λοιπόν για να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Να απαντήσω καταρχάς ε, στον ε, κύριο Κυρίλοφ. Λάβαμε πολλές αιτήσει για προβλήματα που αντιμετωπίζουν ε, οι πολίτες της χώρας, των γειτονικών χωρών και του καθεξής. Πολλές τέτοιες αναφορές λάβαμε. Αν ε, έπρεπε να απαντήσω σε όλες, θα έπρεπε να μετατρέψω το γραφείο μου σε γραφείο αναφορών. Δεν είναι αυτή η εντολή μου. Αυτό όμως που κάνω είναι σε όλες μου τις επαφές με την κυβέρνηση να υπενθυμίσω πάντα τις ευθύνε που έχουν σε ό,τι αφορά τις δικαστικές μεταρρυθμίσεις, τον σεβασμό του δικαστικού σώματος και ούτω καθεξής. Και παρακολουθούμε όλα τα θέματα αυτά. Δεν μπορούμε όμως και δεν είναι και άλλωστε τμήμα της εντολής μας να παρεμβαίνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Σε ό,τι αφορά το θέμα των Ρωμά και την βία κατά των γυναικών ασφαλώς και πρόκειται για ε, σοβαρά και απτά ζητήματα και νομίζω ότι η κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο αντιλαμβάνονται τα προβλήματα και έχουμε αρκετά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να συνδράμουμε την μειονότητα των ε, Ρωμά και για να αντιμετωπιστεί το θέμα της βίας κατά των γυναικών που αποτελεί απτό πρόβλημα, καθώ και όλα τα άλλα θέματα διακριτική μεταχείρισης και στο σημείο αυτό θα είναι πολύ σημαντικό ο νόμος κατά των διακρίσεων και ενθαρρύνουμε την κυβέρνηση να επιτρέψει τη συμμετοχή όλων των επιπέδων της κοινωνίας προκειμένου τελικά να εγκριθεί το καλύτερο δυνατό νομοσχέδιο από το Κοινοβούλιο το οποίο θα αντικατοπτρίζει και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοψίζει και όλα τα προβλήματα. Και τώρα, σε ό,τι αφορά την οικονομική διάσταση, σε ό,τι αφορά τις ε, μειονότητες. Οι κοινότητες ε, ασφαλώς αποτελούν ένα θέμα που διαχωρίζει τι εθνικέ κοινότητε, αλλά η οικονομική πραγματικότητα τη χώρα είναι πραγματικά δύσκολη. Άνω του 30% ανεργία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους νέους και σε πολλά μέρη της χώρας βλέπει κανείς ε, ανέργους στον δρόμο. Ωστόσο, έχουν ληφθεί μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης και ελπίζουμε ότι θα χρηματοδοτηθούν όλα εκείνα τα προγράμματα που χρειάζονται για να διασφαλιστεί ότι τα μέλη της περιθωριοποιημένης αν θέλετε κοινωνίας θα προστατευτούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τις δράσεις της κυβέρνησης και από την χρηματοδοτική ενίσχυση. Και έτσι κλείνω πρόεδρε τα σχόλιά μου. Σας ευχαριστώ εκ νέου για την πρόσκλησή σας. Μπορεί να μην απάντησα ικανοποιητικά όλες σας τις ερωτήσεις, αλλά πιστεύω ότι κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να συνεχίσουμε τις επιτυχίες των τελευταίων ετών και ελπίζουμε να υπάρξει λύση σε ό,τι αφορά το θέμα της ε, ονομασίας τους επόμενους μήνες. Αυτό αποτελεί την ειλικρινή μας ε, επιθυμία. Ευχαριστώ κύριε ειδικέ εκπρόσωπε. Ήταν πολύ η ανταλλαγή απόψεων. Τώρα σε ό,τι φορά τι τροπολογίε ε, που δεν εξετάστηκαν για λόγους ε, χρονικού περιορισμού. Παρακαλώ τους ε, συντάκτες και τους ηγητέ να έχουν μια διμερή συνάντηση ώστε να εξεύρουν τρόπο και να τα συζητήσουν με του συναδέλφου. που δεν μπόρεσαν να εκφράσουν την απόψή του και να απαντήσουν. Ευχαριστώ τον ειδικό εκπρόσωπο. Και περνάμε στο επόμενο σημείο της μεσαίας διατάξεως, ο πρώτος ψηφίσματος σχετικά με την έκθεση προόδου της Κροατίας. Ε, συγητής ο κύριος Βόμποντα, παρακαλώ. Ο κύριος Βόμποντα, ευχαριστώ. Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Είχαμε συνομιλίες και με τους χειώδεις ε, εισηγητές και πετύχαμε σε μεγάλο βαθμό συμφωνία. Υπάρχουν κάποια ανοιχτά ζητήματα τα οποία όμως θα επιληθούν αύριο στην ψηφοφορία. Θα ήθελα καταρχάς να έρθω στο θέμα του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Ακούσαμε και τον ε, κύριο Μπράμετς και διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μία μικρή διαφορά μεταξύ των όσων θεωρεί ο κύριος Μπράμετς απαραίτητα και των όσων πράττει η κροατική κυβέρνηση. Συγγνώμη κυρία Βυσβόποντα. Σας ε, παρακαλώ συνάδελφοι όσοι εγκαταλείπετε την αίθουσα παρακαλώ να αποχωρείτε ησύχως. Άρα δεν έχω τη δυνατότητα να πω ότι υπάρχει ήδη πλήρη συνεργασία και νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να παραμείνουμε στο τύπο το συμβιβαστικό που υπάρχει. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ της κατάστασης που επικρατεί και της πλήρους συνεργασία, αλλά θα πρέπει να αποστείλουμε μήνυμα προς την Κροατία ότι θα πρέπει να καταβληθεί ακόμη μια προσπάθεια για να καλυφθεί αυτό το μικρό χάσμα. Κατά δεύτερον, σε ό,τι αφορά την δικαστική μεταρρύθμιση και την καταπολέμηση της διαφθοράς, η Κροατία έχει πραγματικά πετύχει πάρα πολλά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Φυσικά θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες, αλλά θεωρώ ότι η κυβέρνηση με την καινούργια Πρωθυπουργό θα πρέπει να καταδείξει ότι κανείς, κανείς όσο υψηλή και είναι η θέση του, δεν εξαιρείται από θέματα έρευνας για διαφθορά. Και φυσικά επίσης η σχέση με την Κροατία έχει βελτιωθεί πολύ μεταξύ και της Σλοβενίας, συγγνώμη, έχει βελτιωθεί πολύ. Χαίρομαι που έχει ήδη επικυρωθεί η συμφωνία στο Συμβούλιο και Ελπίζουμε και η Σλοβενία σύντομα να επικυρώσει την συμφωνία αυτή. Τελευταίο θέμα είναι η ημερομηνία. Γίνονται συζητήσεις για το θέμα της ημερομηνίας προσχώρησης της. Είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Πρόκειται για μια ημερομηνία στόχο υπό τον όρο ότι η Κροατία θα συνεχίσει τις ε, προσπάθειές της ε, κατά το έτος 2010. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει την έκβαση, αλλά θεωρούμε ότι μπορεί, μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή εάν η Κροατία συνεχίσει την επίλυση των προβλημάτων. Υπάρχουν κάποιες μικρές διαφορές, όπως είπα, εδώ και εκεί, αλλά νομίζω ότι εν γέννη μπορούμε να ψηφίσουμε αύριο και να αποστέλουμε και τα σχετικά μηνύματα ιδιαίτερα προς την Κροατία, για να τονίσουμε ότι αυτές οι μικρές διαφορές, αυτά τα μικρά χάσματα που παραμένουν, θα πρέπει να γεφυρωθούν, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή το 2010 και φυσικά θα πρέπει να καταβληθούν αναλογικές προσπάθειες και από το Συμβούλιο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε ό,τι αφορά τις καλές ε, γειτονικέ σχέσεις μεταξύ και Κροατίας. Να ζητήσουμε η συμφωνία όντως να κυρωθεί πλήρως, προκειμένου η όλη διαδικασία να τεθεί σε εφαρμογή και σε... να επιληθεί τελικά και το διμερές θέμα, το οποίο αφορά φυσικά και διμερείς σχέσεις μεταξύ Κροατίας και άλλων γειτονικών χωρών. Γενικά είναι θετική η έκθεση και ελπίζω να είναι και η τελευταία έκθεση πρόοδου. Αυτό θα εξαρτηθεί και από το διαπραγματευτικό αποτέλεσμα το οποίο εξαρτάται με τη σειρά του από τις συνεχιζόμενες προσπάθειες α, της Κροατίας. Ευχαριστούμε τον ισίδη και ο Σπόσελ. Δύο λεπτά. Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σβόποντα για το εξαιρετικό κείμενό του και να τον ευχαριστήσω όπως και τους λοιπούς ε, σκιώδες ηγητές, όπως και τους σκιώδες για την πολύ καλή συνεργασία. Συμφωνούμε σε πολλά σημεία στην έκθεση, ίσως κάποια επιμονωμένα σημεία να μας βρίσκουν σύμφωνους. Θα ήθελα να αναφερθώ λοιπόν στα σημεία εκείνα στα οποία έχουμε τις συμβαστικές τροπολογίες και πιστεύω ότι ο κύριος Σφόποντα, ε, σε σχέση με τα όσα είπε ο κύριος ε, Μπράμαλς θα πρέπει να ε, ξανααναλογιστεί το κατά πόσον θα μπορούσε στα δύο, στο δεύτερο τμήμα, στα, από τα τέσσερα που έχουμε χωριστές ψηφοφορίες, να διαγράψει το δεύτερο κομμάτι, γιατί ο κύριος Μπράμαρτς μας είπε ότι δεν γνωρίζει εάν υπάρχουν τέτοιου είδους έγγραφα. Ήταν απόλυτα σαφής η τοποθέτηση του κύριου Μπράμαρτς. και είδαμε ότι ήταν πολύ προσεκτικός πάντοτε στις διατυπώσεις του. Παρακαλώ λοιπόν το κομμάτι αυτό να το διαγράψει ή να αναλογιστεί μια διαφορετική ε, λύση διατύπωση για την πρώτη συμβαστική τροπολογία. Για τη δεύτερη θα καταψηφίσουμε, στη δεύτερη συμβαστική. Η ομάδα μας καταψηφίζει γιατί είπαμε ότι πρόκειται για την έκθεση ε, πλαίσιο που δεν μπορεί να είναι διαφορετικά διατυπωμένη από ότι ε, για τις λοιπές χώρες ενώ βλέπουμε και βλέπουμε ότι για τη Μακεδονία έκθεση είναι διαφορετική από αυτήν ε, που έχουμε στην Κροατία. Δεν μπορούμε να το δεχθούμε λοιπόν. Στη συμβαστική τροπολογία είμαστε σύμφωνοι όπως επίσης και για τις τρεις προφορικές τροπολογίες οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές. Και θα ήθελα να σημειώσω ότι ίσως να υπήρξε κάποια παρεξήγηση παιδογραμματίας. Πολύ γρήγορα να αναφερθώ στην υπαριθμόν δύο προφορική τροπολογία. Κατά την έποψή μου, ως σκιώδου εισηγητού, ε, είχα καταλάβει ότι είχαμε συμφωνήσει να μην υπάρξει η αναφορά στις επερχόμενες τροποποίησεις, upcoming changes στο ε, σύνταγμα της χώρας και να περιμένουμε ότι μόνο πράγματι θα υλοποιηθούν αυτές οι αλλαγές. Τώρα βλέπω όμως ότι έχει συμπεριληφθεί στο κείμενο. Παρακαλώ να το επαληθεύσουμε. Κατά τα άλλα είναι πολύ καλή αυτή η προφορική τροπολογία. Ε, Ο κύριος Βάικελ για δύο λεπτά. Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με τους δύο προηγούμενους ομιλητές για να σημειώσω ότι είναι πολύ θετικό το ψήφισμα μια πολύ καλή εξέλιξη και βέβαια είναι και καρπός πολύ καλής συνεργασίας μεταξύ των πολιτικών μας ομάδων εδώ στο Κοινοβούλιο και κυρίως όσων εξημών ενεργά συμμετέσχουν στην διατύπωση του σχεδίου ψηφίσματος. Θα ήθελα να πω ότι είναι θετικό το κείμενο, είναι πηγή ε, ελπίδας, ενθαρρυντική. Κάποια προβλήματα παραμένουν, ωστόσο θα πρέπει οι αρχές Κροατίας να αντιμετωπίσουν και πιστεύω ότι η ανάληψη των ε, καθηκόντων της νέας κυβέρνησης αποτελεί ήδη ένα πολύ καλό μήνυμα. Δείχνει ότι η νέα αυτή κυβέρνηση θα έχει διαφορετική στάση απέναντι στη διαφθορά, το οργανωμένο έγκλημα και λοιπά προβλήματα που έχουμε επανελειμμένως επισημάνει σε σχέση με την Κροατία. Ο πόλεμος είχε πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην Κροατία και μαζικές ε, μαζική μετανάστευση από πολιτών και οι καλύτερα προσφυγικές ροές και τώρα πολλές περιπτώσεις, πολλούς Σέρβους περιμένουν να επανέλθουν στις αιστείες τους. Ε, είναι η στιγμή πιστεύω να υπενθυμίσουμε στην Κροατία το χρέος που έχει απέναντι στους πολίτες της και βέβαια την νομοθετική της υποχρέωση να διευκολύνει τον επαναπατρισμό των προσφύγων αυτών. και να διορθώσει τα δεινά του παρελθόντος. Επίσης, ε, ε, εκφράζονται εδώ προσδοκίες η Κροατία, όπως και η Σερβία και άλλες χώρες που μεταφούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να αρχίσουν να χρησιμοποιούν κοινή γλώσσα. Γλώσσα δεν υπάρχει γιουγκοσλαβική γλώσσα. Πρέπει να δείχνουμε ανοχή και ε, αποδοχή των διαφορετικών γλωσσών που υπάρχουν τόσο στην πρώην Ιουγκοσλαβία όσο και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Κύριος Μπράντερ για δύο λεπτά. Κυρία. Πρόεδρε ευχαριστώ. Η έκθεση και οι συμβαστικέ τροπολογίε είναι πολύ καλέ, πολύ καλό πνεύμα διατυπώθηκαν. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ σημαντική είναι η, πρόοδο που έχει σημειώσει η Κροατία στην ενταξιακή τη πορεία. Βεβαίω και παραμένουν ε, τα έγγραφα αυτά, κύρια έγγραφα και επιβεβαιώνεται από τα όσα ακούσαμε και σήμερα σχέση με το Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωση και ότι θα πρέπει να επιβίνουμε ώστε να προχωρήσουμε στην υπόθεση αυτή, να επιτευχθεί πρόοδο. Ένα άλλο θέμα στο οποίο θα θέλω να φερθώ είναι το ζήτημα τη δικαιοσύνη και η εφαρμογή τη νομοθεσία προ τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των μειονοτήτων, όπου υπάρχουν κάποιε πρόοδε προ την νομοθετική πτυχή, αλλά δεν υπάρχει επαρκή πρόοδο στην υλοποίηση και θα θέλαμε να ζητήσουμε επιπλέον, άλλωστε το έχουν υπογραμμίσει μέσα από το κείμενο και οι τροπολογίε μα, αυτή την πτυχή. Για το 2010 βλέπω ότι δεν ορίζεται πλέον ως προθεσμία καταληκτική το μέσο, τα μέσα του 2010. Εμείς ως ομάδα θεωρούμε ότι έχουμε μια γενική υποχρέωση, ευθύνη καλύτερα για την ενταξιακή διαδικασία ολόκληρη τη πρώην και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και με την Κροατία. Εάν κάνουμε το σφάλμα που διαπράξαμε με την ε, Βουλγαρία και τη Ρουμανία, προσδιορίζοντα συγκεκριμένη ημερομηνία προσχώρηση, για να διαπιστώσουμε στη συνέχεια ότι δεν ήταν αρκετά έτοιμε οι χώρε και χρειαζόταν να ετεθούν υπό επιτήρηση, ε, θα έχουμε αποστείλει πολύ λάθο μηνύματα, θα έχουμε κάνει μεγάλο σφάλμα και νομίζω ότι είναι, το χειρότερο αυτό παρά, ε, είναι χειρότερο αυτό παρά να πούμε στι χώρε και στου πληθυσμού ότι θα πρέπει να κάνουν περισσότερες προσπάθειε για να προσαρμοστούν στο κοινωτικό κεκτημένο. Είναι ε, σφάλμα λοιπόν να μιλάμε για 2010 και ταχύρυθμη διαδικασία ε, ένταξης με επιτήρηση. Θα ήταν το χειρότερο αποτέλεσμα αυτό. Α είμαστε τίμοι λοιπόν με τη χώρα αυτή και α του πούμε ότι τώρα θα κρυθούν μόνο όταν θα είναι απολύτως έτοιμοι χωρίς επιπλέον επιτήρηση. Ας μην τους δίνουμε κάποια αυθαίρετα κριτήρια ή ε, προθεσμίες οι οποίες συνεπάγονται ότι θα παραμείνουν ε, για καιρό μετά υπό καθεστώς επιτήρησης. Να είναι έτοιμη η Κροατία και μετα απο καθεστως επιτηρησης να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς επιτήρηση. Ο κύριος Πέτερ λέγε δύο λεπτά. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάθε φορά που είχαμε να εξετάσουμε έκθεση και σημειώναμε την πρόοδο της, ε, ιδιαίτερα τη Κροατία που είναι και γειτονική τη ε, πατρίδα μου Σλοβενία, αισθανόμουν ιδιαίτερη χαρά και γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερω για τι προσπάθειε του κύριου Σλόμποντα, ε, προσπάθειες ε, που στοχεύουν στην όσο δυνατόν πιστή παρουσία της κατάστασης ε, στην Κροατία. Τον ευχαριστώ λοιπόν πολύ φυσικά και εμείς τον ε, συνδράμαμε στις προσπάθειες αυτές. Ε, καθήκον μας είναι, πιστεύω, να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη μιας ατμόσφαιρας, ενός κλίματος καλύτερα, που θα ενθαρρύνει την ε, πρόοδο, ενός κλίματος το οποίο μάλλον θα τίνει προς μια ισορροπημένη λύση για κάθε εκρεμές πρόβλημα που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν. Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να σημειώσω επίσης ότι η έκθεση είναι ισορροπημένη, έχει καλές ισορροπίες και δεν δείχνει κάτι που βλέπαμε στο παρελθόν ε, σε άλλες εκθέσεις ως υπέτεια για την έλλειψη προόδου την Σλοβενία. Βεβαίω θα μπορούσαμε να βρούμε καλύτερε ισορροπίε στο παρελθόν, ε, σε ορισμένα σημεία. Αλλά οι ε, αντιρρήσει που είχε στο παρελθόν διατυπώσει η Σλοβενία δεν είναι παρά μόνο ένα μέρο ε, επιφυλάξεων ή αντιρρήσεων που έχουν διατυπώσει και άλλε χώρε. Και γι' αυτό θέλουμε να υπάρχουν τροπολογίε που να αντικατοπτρίζουν στην πραγματικ την πραγματική κατάσταση. Εμεί θέλουμε πράγματι να αριθμιστεί η κατάσταση το χειτερό δυνατό και να προχωρήσει η ένταξη της ε, Κροατίας στο χειρότερο δυνατό υπό τους κατάλληλους όρους και προϋποθέσεις, έτσι ώστε να κερδίζουμε όχι μόνο και οι δύο πλευρές αλλά και οι τρεις πλευρές, και η Κροατία και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η Σλοβανία. Η Σλοβενία. Για τα μεταξύ μας προβλήματα διαιτητής, ε, επιδιαιτητής νομίζω δεν χρειάζεται, πρέπει να είμαστε σε θέση μεταξύ μας να τα επιλύσουμε. Και επίσης θα ήθελα να σημειώσω ότι η διαδικασία της επιδιαιτησίας έχει γεννήσει πολλές ελπίδες βλέπω ότι δυστυχώς ε, η τοποθέτηση του Επιτρόπου Ρεν, ε, η φιλοσοφική αν θέλετε θεώρηση του Επιτρόπου Ρεν, έχει εγκαταληφθεί μάλλον και, ότι θα, και λέγεται ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε ταυτόχρονα να πιέσουμε προς την ένταξη και την επίλυση των διμερών ε, διαφορών με την επιδιαιτησία. Τώρα βλέπουμε ότι η επιδιαιτησία θα ξεκινήσει μόνο μετά από την Συμφωνία Σύνδεση της Κροατίας, πράγμα το οποίο είναι μάλλον αρνητική εξέλιξη και θα έχει σοβαρέ επιπτώσει. Γι' αυτό ελπίζω οι δύο χώρε με τη βοήθεια και την αρρωγή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσουν να βρουν τρόπο να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά εν ευθέτω χρόνο. Ευχαριστώ. Έχουμε πρόσωπο της Κομισιόν που επιθυμεί να παρέμβει. Όχι. Κύριε Σβόμποντα, αν θέλετε να σχολιάσετε τα όσα ακούστηκαν. Με ενδιαφέρον θα σας ακούσουμε. Για τα θέματα τα οποία ανέφερε ο συνάδελφος Πέτερλε μόλις, θα πρέπει να διευκρινίσω ότι αντικείμενο της συμφωνίας είναι η διαδικασία διαπραγματεύσεων να γίνει μετά τις διαπραγματεύσεις. Δεν μπορούμε να αντιστρέψουμε αυτό. Αυτά που έχουν συμφωνηθεί ε, θα πρέπει να ακολουθηθούν. Έτσι έχει συμφωνηθεί για το θέμα της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας και το σχετικό επιχείρημα υπάρχει μια διαφορά γιατί τότε είχε αναφερθεί συγκεκριμένη ημερομηνία ένταξης προς την οποία κινηθήκαμε. Τώρα μιλάμε μόνο για μια δυνατότητα, δυνατότητα να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις με όλες τις διαδικασίες επικύρωσης που θα πρέπει να ακολουθήσουν. Κατά τρίτον, προς τον κύριο Πόσελτ να απαντήσω. Μπορώ να φανταστώ μια τέτοια αλλαγή, αλλά αυτό ασφαλώς εξαρτάται από το κατά πόσο θα συμφωνήσουμε, γιατί μπορεί να θέλετε να αποδυναμώσετε την ε, τροπολογία. Θα μπορούσε να είναι μια συμβαστική τροπολογία που θα διατυπώνει το εξή το πρώτο τμήμα προς το τέλος, ότι επαναλαμβάνει ότι μία ανησυχία δεν έχει αντιμετωπιστεί και έχετε δίκο, δίκιο. Μίλησε για το ένα αυτό θέμα ο κύριος Μπράμερτς, μία ανησυχία. Η πρόοδος για την εξέβρεση των ε, απολεσθέντων στρατιωτικών εγγράφων και μετά να πούμε ότι καλούμε εκ νέου την κυβέρνηση της Κροατίας να εντατικοποιήσει τις προσπάθειές της σε ό,τι αφορά την πλήρη συνεργασία με το ΙΚΤΙ. Ε, έτσι θα παρακάμψουμε το θέμα της, ε, των στρατιωτικών εγγράφων. Θα έχουμε κάνει μια γενικότερη διατύπωση. Μπορούμε να το συζητήσουμε με τον συνάδελφο Πόσελτ να γίνει μια τέτοια αλλαγή. Αν θεωρεί ότι και αυτό είναι υπερβολικά επικριτικό, θα πρέπει να ψηφίσουμε τι να γίνει. Αυτά κύριε Πρόεδρε. Και όπως σας είπα, ο... τις μικρές αυτές διαφορές μπορούμε να τις ψηφίσουμε σε δημοκρατικό πλαίσιο. Δεν θεωρώ όμως ότι κατά τα άλλα υπάρχουν σημαντικά προβλήματα. Να αναφέρω ένα στοιχείο ακόμα. Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας της Κροατίας κατέδειξε και την οριμότητα της χώρας γιατί μεταξύ του πολύ λαϊκιστικά ενεργούντα υποψηφίου αφενός και ενός υποψηφίου που τελικά εκλέχθηκε, φάνηκε ποιος εκλέχθηκε. Ο σοβαρός υποψήφιος, ο οποίος τάχθηκε κατά της ε, διαφθοράς. Νομίζω ότι ήταν πολύ θετικό το σημείο αυτό, το μήνυμα αυτό που έστειλε η Κροατία. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Θα πρέπει να διακόψουμε για τρία λεπτά. Για τεχνικούς λόγους δεν υπάρχει κανένας αντιπρόεδρος που να μπορέσει να με αντικαταστήσει. Συγγνώμη. Επανέρχομαι δρυμύτερος. Προτού να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια κυρία Όμεν Ρόιτεν για την πρόταση ψηφίσματος ε, σχετικά με την έκθεση προόδου της Τουρκίας, θα ήθελα να καλωσορίσω την αντιπροσωπεία της Επιτροπής ε, του Κοινοβουλίου της ε, Τουρκίας τις εξωτερικές υποθέσεις και την πρόεδρό του. Η ε, αντιπροσωπεία αποτελείται από μέλη της ε, Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Εναρμόνιση των Ευρωπαϊκών Προτύπων και τον συμπρόεδρο της Μικτής ε, Επιτροπής Τουρκίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν η συνέλφος ο Μανρό ήταν είναι έτοιμη, τη βλέπω πανέτοιμη στο έδρανό της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 Παρακαλώ, εξέλθετε τις αιθούσεις. Πρέπει να ακούσουμε την κυρία Όμεν Ρόιτεν ηρέμος. Ευχαριστώ πρωί, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την σημαντική συνεισφορά τους στην ε, σύνταξη της ε, εκθέσεώς μου. Υπήρξε πολύ καλή συνεννόηση και διαβούλευση με τους σκιώδεις ηγητές και για τον λόγο αυτό μπορέσαμε να εναρμονίσουμε τις θέσεις μας επί πολλών σημείων. Θα ήθελα, Πρόεδρε, το Κοινοβούλιο μας να λάβει μια σαφή θέση, ισόρροπη αλλά και συνεπή. Και ψάχνω λοιπόν, ε, αναζητώ μια ευρεία πλειοψηφία. Πρωτού περάσω στις ε, τροπολογίες, θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρίες οι οποίες ε, θεωρώ ότι είναι σχετικές και για μένα και για τους συναδέλφους. Παρατηρήσεις για πρόσφατες εξελίξεις. Καταρχάς, να πω το εξής, ότι την προηγούμενη εβδομάδα έγινε μια συζήτηση στο Στρασβούργο για την απαγόρευση του DTP. Μετά την απόφαση του δικαστηρίου το Δεκέμβριο έγιναν κάποιες ε, τρομοκρατικές επιθέσεις και έγιναν συλλήψεις από το DTP και ακόμα επαπειλούνται περαιτέρω συλλήψεις η πολύ θετικά αξιολογούμενη συζήτηση που είχε ξεκινήσει το καλοκαίρι φαίνεται να έλαβε τέρμα, τέλος. Και εγώ ως εκπρόσωπος ε, του Κοινοβουλίου θα πρέπει να λάβω αποστάσεις από τις αποφάσεις του δικαστηρίου, αλλά από ό,τι κατάλαβα, ακόμα και το δικαστήριο ζήτησε την εφαρμογή των συστάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Επιτροπής της Βενετίας. Και γι' αυτό λοιπόν στη συμβαστική υπαριθμών 4 προσπαθώ να αποτυπώσω με τον σαφέστερο δυνατό τρόπο την στάση μας. Πρόεδρε, μιλάω λίγο πιο αργά για την προηγούμενη φορά ε, ήταν λάθος η διερμηνία προς τα αγγλικά. Έγινε κάποιο λάθος, γι' αυτό λοιπόν θα μιλάω τώρα πάρα πολύ αργά. Την προηγούμενη πέμπτη, Πρόεδρε, το Συνταγματικό Δικαστήριο εξέδωσε μία απόφαση για την δικαιοδοσία των στρατιωτικών δικαστηρίων και τον νόμο που θα περιόριζε την δικαιοδοσία αυτή την οποία αξιολογώ θετικά στην έκθεση μαζί με τους συναδέλφους. Το Συνταγματικό Δικαστήριο α, πάρα ακύρωσε την απόφαση αυτή. Και αυτό με ανησυχεί ιδιαίτερα. Και επίσης ανησυχώ η υπόθεση βαριά, sledgehammer, στην Τουρκία και ποιος θα είναι ο αντίκτυπός της. Νομίζω, Πρόεδρε, ότι όλα αυτά που αναφέρω, η απόφαση του δικαστηρίου α, λαμβάνεται υπόψη βάση νομοθεσίας. Αν λοιπόν λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις βάση νομοθεσίας, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι σαφές ότι χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση, γιατί μόνο αυτό θα λύσει τα προβλήματα. Γιατί οι πρόσφατες αποφάσεις ενισχύουν την έκκλησή μας προς την κυβέρνηση αλλά και προς την αντιπολίτευση, Πρόεδρε, να συνεργαστούν προκειμένου να επιληθεί το πρόβλημα αυτό το συνταγματικό και να γίνουν όλες οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες είναι απαραίτητες. Ένα τρίτο σημείο, Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έκανε ένα πρώτο έλεγχο για τις ε, ε, επιχορηγήσεις που έγιναν το 2002 έως 2006. Το 2002 έως 2004 ε, είχε αναφερθεί ότι δεν ήταν επαρκής ο ρυθμός απορρόφησης στην Τουρκία. Από το 2004 στο 2006, Πρόεδρε, υπήρξε αυτή η ικανότητα απορρόφησης των πόρων. Έγινε καλή διοργάνωση από πλευράς της Τουρκίας και νομίζω ότι θα πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό, αλλά ε, το θέμα είναι ότι τέθηκαν υπερβολικά πολλέ προτεραιότητε και τελικά δεν υπήρχε καμία προτεραιότητα. Και θα ήθελα να ζητήσω λοιπόν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τον αντίκτυπο του μέσου ΕΠΑ, το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί με καλύτερο τρόπο. Πρόεδρε, να κοιτάξουμε τώρα τις τροπολογίες. Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες και τους συμβιβασμούς, να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτη παρατήρηση. Προσπάθησα να ε, χωρέσουν όλα στις συμβιβαστικές τροπολογίες. Υπήρχαν ε, κάποιες τροπολογίες οι οποίες δεν είχαν ε, να κάνουν απαραίτητα με την πρόοδο το 2009. Γι' αυτό και δεν τις συμπεριέλαβα. Στα υπόλοιπα θέματα ακολουθώ τις συστάσεις των συναδέλφων σε ό,τι αφορά την ε, τροπολογία 70 του κ. Ντιλάμστορφ, του κ. Μάουρο 116, του Λάμστορφ 167, του κ. Χατζηγεωργίου 137, 173, Χάουιτ και ούτω καθεξής. Πρόεδρε, λοιπόν, στα υπόλοιπα παραμένουμε κατά. Το θέμα της Κύπρου που έπαιξε μεγάλο θέμα σε ό,τι αφορά το EPC. Μαζί με τους κοιότητες εισηγητές αναζήτησα μια σαφή αλλά και ευρεία συμφωνία. Γιατί υπήρχαν πολλές αντικρουόμενες απόψεις και θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους τώρα να σεβαστούν αυτή την ισορροπία που επικράτησε, γιατί αυτός είναι ο σκοπός, να καταλήξουμε στην συμβαστική υπαριθμό 10 και ζήτησα να αποσυρθούν όλες οι τροπολογίες σε ό,τι αφορά την παράγραφα 28, 29, 30 και η ιατρολογική σκέψη 1. Πολλοί δεν το έχουν κάνει και πολλοί μπορούν να το κάνουν ακόμη. Και να επαναλάβω, Πρόεδρε, και έξω ονόματος των σοσιαλιστών συναδέλφων, ότι η αίσθησή μου για την αναζήτηση και την εξέβρεση συμβιβασμών είναι να μείνει έτσι ο συμβιβασμό. Ένα τρίτο σημείο, Πρόεδρε, το οποίο μου προκαλεί ειλικρινά ανησυχία. Τις τροπολογίες οι οποίες ε, υπευλήθησαν για την ιδεολογική σκέψη Α, είπα ότι δεν μπορώ να τις υποστηρίξω. Και γιατί, γιατί Πρόεδρε, γιατί Έχω εμπειρία στο Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά την έκθεση αυτή και γνωρίζω επίσης ότι, για παράδειγμα, η τροπολογία 28 έχει μεγάλες πιθανότητες να μην υποστηριχθεί από την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου. Επιπλέον, η τροπολογία υπαρθμών 28 δεν προσθέτει κάτι στην αιτιολογική σκέψη Α, γιατί η αιτιολογική σκέψη Α αποτελεί ένα συμβιβασμό, την οποία τότε είχα συμφωνήσει και με τον συνάδελφο Σβόμποτα και με άλλους συναδέλφους. Και τι αναφέρει η τελογική σκέψη α, ότι η προσχώρηση αποτελεί και πολύ προσεκτικά έχουμε διατυπώσει το κείμενο που δεν προκαλεί απογοήτευση σε άλλους για να αναφέρουν και άλλες δυνατότητες οι οποίες δεν αποτελούν όμως το στόχο των δράσεών μας η έναρξη διαπραγματεύσεων σύμφωνα με το πρωτόκολλο προσχώρησης. Πρόεδρε, τέλος να επαναλάβω ότι και φέτος στόχος μου θα είναι να θέσω ένα σαφές μήνυμα με την έκθεση αυτή και να επαναλάβω άλλη μια φορά ότι η έκθεση αυτή τώρα πλέον βρίσκεται στα χέρια τα δικά σας, στα χέρια των βουλευτών. Η έκθεση αυτή θεωρώ αποτυπώνει την ισχυρή πεποίθηση σε ό,τι αφορά την ένταξη της Τουρκίας και θα πρέπει να αποστείλουμε ένα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία. Ένα σαφές μήνυμα το οποίο θα περιλαμβάνει όλους τους βουλευτές του Κοινοβουλίου. Το μήνυμα αυτό μπορεί να είναι ισχυρό μόνο αν συνειδητοποιήσουμε ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλες τις θέσεις και επειδή αυτό φροντίζω να γίνει. Αυτό φρόντισα να γίνει. Ζητώ από τα μέλη, από τους βουλευτές που δεν απέσυραν α, τις τροπολογίες τους, τους ζητώ για μία φορά ακόμη να τις αποσύρουν. Γιατί μόνο έτσι θα αποστείλουμε το ισχυρό μήνυμα που θέλουμε να αποστείλουμε εξ ονόματος όλων. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Έχω έναν ε, σημαντικό αριθμό συναδέλφων που ζήτησαν το λόγο. Παρακαλώ, λακωνικοί. Καταρχήν θα δώσω το λόγο στους ε, συντονιστές ε, και οδησηγητές που στην περίπτωση αυτή είναι η αυτοί. Ο κ. Χάουιτ έχει το λόγο για δύο λεπτά. Αν πρόκειται για δύο λεπτά, πρόεδρε, θα πρέπει να συμπιέσω πολύ αυτά που θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει, ξεκινώ ευχαριστώντα την κυρία Όμεν Ρόιτσεν. Δεν μπορέσαμε να καταλήξουμε σε πλήρη συμφωνία, αλλά πάντω κάναμε απεγνωσμένε προσπάθειε να το καταφέρουμε. Υπάρχουν κάποιοι τομεί διαφωνία, αλλά είναι πολύ λίγοι πλέον. Η φιλοσοφία που χαρακτηρίζει τις ε, τροπολογίες μας, τροπολογίες τη οριστικής ομάδας για το δεύτερο τμήμα, το βεβαίω βεβαίως ε, περίοδο, είναι επικριτικές για να αντιμετωπιστούν κάποια δύσκολα προβλήματα σχετικά με την Κύπρο και ιδιαίτερα των επικιστών από την Τουρκία στο Ινένο ε, νήσο στο βόρειο κομμάτι του νησιού δηλαδή, τα προβλήματα της αντιμετώπισης των μειονοτήτων και θέλουμε να εξορροπήσουμε το κείμενο. Όπως είπε και η κυρία Όμεν Ρόιτεν, υπάρχουν διαφορετικέ επιλογές, δύσκολες επιλογές και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι με την έκθεση αυτή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει την υποστήριξή του, την υποστήριξη για τη μεταρρύθμιση στην Τουρκία. Συμφωνούμε, μπορούμε να συμφωνήσουμε για τις συμβαστικές τροπολογίες. Δύο μόνο πτυχέ θα ήθελα να επισημάνω στη συζήτηση εδώ, ότι καταρχάς ήθελε η συγγήτρια να αποσύρουμε την υπαριθμόν 28 ε, ε, την υπαριθμόν 1 τροπολογία στην 28 παράγραφο όπου ε, σημειώνουμε ότι έχει ξαναρχίσει η μεταρρύθμιση, η διαδικασία των μεταρρυθμίσεων, αλλά χρειάζεται περισσότερη ε, αποφασιστικότητα στην πορεία αυτή και να σημειώσουμε τα, τα συμπεράσματα τη ε, εκθέσεω πρόοδου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέγοντα όμω, ότι, κύριο, ότι αποτέλεσμα, επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και κατάληξη αυτή τη διαδικασία πρέπει να είναι η πλήρη ένταξη και επίση λέμε ότι θα πρέπει πλέον ω Κοινοβούλιο να ε, εκθέσουμε τη διατύπωση αυτή της ε, πλήρου συμμετοχής σε μια δοκιμασία για να ζητήσουμε να τοποθετηθούν οι μεν και οι δε. Δηλαδή να πούμε με την τροπολογία αυτή, κοιτάξτε τι λέμε εμείς στην Τουρκία, κοιτάξτε τι λέει η Τουρκία σε εμά και εμείς να απαντούμε ναι, παρακαλούμε συνεχίστε αυτή τη διαδικασία για την ένταξη και εμείς θα σα υποστηρίξουμε μέχρι το τέλο. Αυτό λοιπόν για να ε, απευθυνθώ τώρα προ τον Πρόεδρο και τη Γραμματεία. Ο κατάλογο των, των ε, ψηφοφοριών για, την, για τη συμβαστική τροπολογία παριθμών 10 συμπεριλαμβάνει και τι τροπολογίε για την παράγραφο 28 αλλά και για την αδειολογική σκέψη Α. Θα δείτε λοιπόν από τι σημειώσει τη προηγούμενη εβδομάδα από τη συνεδρίασή μα ότι δεν είχαμε συμφωνήσει στην συνεδρίαση ότι συμφωνήσαμε στη συνεδρίαση 152 τροπολογίε τη σοσιαλιστικής ομάδας και 22 και 23 των σοσιαλιστών μεμονωμένων μελών ε, για την, ε, θα πήγαιναν στη συμβαστική τροπολογία υπεριθμών 10 και θα, γινόταν, ε, θα ενσωματώνονταν εκεί. Παρακαλώ λοιπόν αυτό να αντικατοπτριστεί, διότι θα θέλαμε να έχουμε τη δυνατότητα τη τροπολογία μα, στην υπέρ 152, 22 και 23, να τι υποβάλουμε προ ψηφοφορία, παρακαλώ. Κύριε Χόβιτ, ξεπεράσατε κατά πολύ τον χρόνο που σας είχαμε δώσει. Επειδή μιλήσατε για ένα τεχνικό ζήτημα, σας άφησα να συνεχίσετε. Αλλά παρακαλώ, συνάδελφοι, φροντίζετε οι παρεμβάσεις σας ε, να μην υπερβαίνουν τα δύο λεπτά. Ο κύριος Ντάσντορφ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και εγώ την ε, Ρία και τους άλλους συναδέλφους για την πολύ καλή συνεργασία. Ε, είχαμε πολύ καλή συνεργασία όντως με αποτέλεσμα μια ισορροπημένη έκθεση στην οποία εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούμε να εκφράσουμε την υποστήριξή μας για τη μεταρρυθμιστική ατζέντα της Τουρκίας. Ε, ρητά το ανέφερε και ο κύριο Χάουιτ και τον υποστηρίζω. Ε, πρέπει να στηρίξουμε τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στην Τουρκία. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς πιστεύω, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πιστεύω ε, ότι δεν πρέπει να ψηφίσουμε την τροπολογία υπαριθμών 28, στην ε, παράγραφη υπαριθμών 28, γιατί έχουμε βρει συμβαστικές λύσεις που μιλούν για τις πραγματικές προενταξιακές και δεν υπάρχει λόγος τώρα να επαναλαμβάνουμε ποιοι είναι οι στόχοι, ε, ότι είναι ανοιχτή διαδικασία, ότι μπορεί να υπάρξει πλήρη ένταξη εφόσον εκπληρωθούν όλα τα κριτήρια, αλλά ότι δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι η κατάληξη διαδικασία. Γι' αυτό είναι πολύ καλά ισορροπημένη τωρινή διατύπωση της ε, τυρολογικής σκέψης παριθμών α και γι' αυτό θα ήθελα να απορριφθούν οι όποιες τροπολογίες έχουν υποβληθεί σε αυτήν. Απευθύνουμε με την έκθεση αυτή τώρα ένα πολύ σαφέ μήνυμα που έχει να κάνει και με την ομολογία του Σταγματικού Δικαστηρίου και ευχαριστώ την κυρία Όμεν Ρόιτεν για την προφορική τροπολογία στην υπαριθμόν 9 ε, παράγραφο, γιατί βεβαίω και θέλουμε να υπάρχει ο έλεγχο τη πολιτική δικαιοσύνη, τη πολιτική πάνω στην ε, στρατιωτική εξουσία και γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι ήταν σφάλμα, ότι ήταν ατυχής η, εν λόγω δικαστική απόφαση. Επίσης θέλουμε να υποστηρίξουμε την ελευθερία του λόγου και της έκφρασης ε, για τα δικαιώματα του τύπου και την ανεξαρτησία του τύπου την παράγραφο, στην παράγραφο 23 συμφωνούμε με την τροπολογία που στοχεύει στην, ε, ε, στο στόχο αυτόν Θεωρούμε όμω ότι θα πρέπει να υπάρχει το κατάλληλο νομικό πλαίσιο που να εξασφαλίζει την ελευθεροτυπία και την ανεξαρτησία των μέσων μαζική ενημέρωση, πράγμα το οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Η κυρία Φλότο, πρόεδρο τη Επιτροπή τη Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Και εγώ να συμφωνήσω με τις ευχαριστίες που ακούστηκαν διότι αυτό από αυτό το έργο που έχουμε μπροστά μας αποτελεί τον καρπό μια ευρύτατη συνενέσεως. Τώρα το ότι οι συζητήσεις μας ε, εξαφάνισαν κάθε ενδιαφέρον για την αυριανή ψηφοφορία κλπ. Όχι. Δεν έχει συμβεί αυτό, αλλά βρισκόμαστε πολύ κοντά στις θέσεις μας, συμμεριζόμαστε τις απόψεις που περιέχονται και το τι θα πρέπει να πούμε σήμερα για την κατάσταση που επικρατεί στην Τουρκία. Θα ήθελα να καταστώ πιο σαφής σε ό,τι φορά τις τροπολογίες και τις συμβαστικέ προτάσεις που έχουν καταπιστεί. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ την κυρία Μενρόιτε ε, που προσέθεσε μια προφορική τροπολογία που επιτρέπει να εκφράσουμε την απογοήτευση που ε, προκύπτει από την απόφαση του Δικαστηρίου. Θεωρώ ότι έχουμε απόλυτο δίκιο αλλά χρειάζεται να συνοδέψουμε αυτήν την λύπη μας ε, μια αίτηση αναζήτησης από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση μιας συνένεσης και αυτό είναι κάτι το οποίο πονάει διότι υπήρξε η απομάκρυνση η αυτού του κόμματος θα μπορούσαμε πούμε από την ε, Λοιπόν, θα πρέπει να υπάρξει μια ευρύτερη συνένεση στην ε, τουρκική εθνοσυνέλευση πάνω στο ζήτημα. <clears throat> Αποσύρω τροπολογία με παρθμό 16, αλλά νομίζω πως η κυρία Ομινρόιτον το έχει καταγράψει, αφορούσε το θέμα της ε, προστασίας και φύλαξης κάποιων χωριών. Τώρα για την τροπολογία 132 που δεν είναι αντικείμενο συμβασμού να επιστρέψει την προσοχή των συναδέλφων σχετικά με την κατάσταση των αντιρρησιών συνείδηση, που είναι μια, ένα καθεστώ μη αναγνωρισμένο και αυτό παραβαίνοντα ε, την απόφαση του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτό είναι ένα θέμα που αφορά πολλά πρόσωπα στην Τουρκία και εμεί εδώ ω κοινοβουλευτικοί θα πρέπει να κάνουμε μια ρητή αναφορά στο πρόβλημα και καταλήγω στην, ε, στον συμβασμό 10 που αντιθέτως από ό,τι αναφέρεται στην κατάλογο των ψηφοφοριών η τροπολογία 156 δεν αποτελεί μέρος αυτού του συμβασμού στο μέτρο που θα υπάρξει χωριστή ψηφοφορία πάνω σε κάτι το ιδιαίτερα απλό το οποίο λέει ότι επιθυμούμε η Τουρκία να καταβάλει κάθε προσπάθεια όπως επίσης και τα εμπλεκόμενα μέρη, δηλαδή εμείς, το Ηνωμένο Έθνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. για την εξέβρεση μιας ε, διαρκούς ε, λύσης του προβλήματος της Κύπρου και αναφέρω την τροπολογία 28 που επιβεβαιώνει τον στόχο της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρώ ότι είναι σωστή και θα τύχει της υποστήριξης μας. Ευχαριστώ συνάδελφε. ευχαριστώ κυρία Ρόιτον. Το λόγο έχει ο κύριος Βαν Όρντεν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν έπρεπε να εξαντλήσω το δίλεπτό μου, γιατί καταρχάς θέλω να πω ότι όντως συμφωνώ που θα πρέπει να απευθύνουμε ένα σαφές μήνυμα στην Τουρκία ως προς την ανάγκη να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να είμαστε και δίκαιοι και ακριβοδίκαιοι και ακριβείς και να μην καταχρώμεθα της ιδέας των συμβαστικών ή της λύσεως των συμβαστικών τροπολογιών, διότι κατά με συμβαστική τροπολογία είναι μια τροπολογία η οποία αντικατοπτρίζει όλα τα στοιχεία του συμβασμού. Η υπαριθμόν 10 όμως, σαφώς, ενώ ισχυρίζεται ότι έχει συμπεριλάβει την 140, την 169 και την 175 δικές μου τροπολογίες, σαφώς δεν τις αντικατοπτρίζει. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν οι συμβαστικές τροπολογίες να χρησιμοποιούνται ως ε, μέθοδος ε, απαλυφής από τον κατάλογο των ψηφοφοριών των τροπολογιών των βουλευτών. Γιατί αυτό βλέπω να συμβαίνει και παρακαλώ να διορθωθεί ο κατάλογος των ψηφοφοριών ώστε να αντικατοπτρίζονται και οι δικές μου τροπολογίες. Και αυτό που ζητώ είναι μια ισορροπημένη προσέγγιση. Φερρυπίν. Στην 169 τροπολογία μου δεν απευθύνω απλώς έκκληση προς τουρκική κυβέρνηση να υποστηρίξει ενεργά τις ε, συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις ε, που γίνονται στην Κύπρο, αλλά απευθύνω έκκληση και προς τις λοιπές κυβερνήσεις, όπως σε παραδείγμα την ελληνική. Πρέπει και προς την ελληνική κυβέρνηση να απευθύνουμε έκκληση για να συμβάλλει σε θελική θετική των διαπραγματεύσεων. 175 έχει να κάνει με τις ε, δραστηριότητες εξόρυξης πετρελαίου στην Ανατολική Μεσόγειο, σε αμφιλεγόμενες, διαφυσμητούμενες ζώνες πράγμα το οποίο θα έχει και επιπτώσει ως προς τις προσπάθειες για επίλυση του κυπριακού ζητήματος. Πρέπει να συμπεριληφθεί το κείμενο αυτό, Πρόεδρε. Και όταν επιπλέον λέμε ότι δεν εφαρμόζει το πρόσθετο πρωτόκολλο, ή το συμπληρωματικό πρωτόκολλο η Τουρκία, θα πρέπει ταυτόχρονα και να σημειώνουμε ότι ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει τη δική της απόφαση περί άρσης της απομόνωσης της Βόρειας Κύπρου, που είναι, αν μπορώ να το πω έτσι, η άλλη όψη το αντάλλαγμα για αυτή τη συμφωνία και δέσμευση. Με ανησυχεί ιδιαίτερο το γεγονός ότι γίνεται κατάχρηση των συμβαστικών τροπολογιών. Ευχαριστώ κύριος Χατζηγεωργίου για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θέλω πρώτα απ' όλα να συγχαρώ για την κυρία Νόουμε για τον κόπο τη, τη μεγάλη δουλειά που έχει καταθέσει και όλους τους συναδέλφους που εργάστηκαν Κύριε Πρόεδρε, εμεί είμαστε υπέρ τη ένταξη τη Τουρκία. Ξεκινώ πάντα την αναφορά μου όταν συζητούμε θέμα Τουρκία με αυτή την φράση. Γιατί θέλω να γίνει κοινή πεποίθηση ότι καταλαβαίνουμε καθαρά και σταθερά ότι το συμφέρον και της Κύπρου είναι η εκδημοκρατικοποίηση της Τουρκίας, η λύση του Κυπριακού και η συνακόλουθη ένταξή της. Είμαστε στο μέσο συνομιλιών, κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι στην Κύπρο και νομίζω ότι οι τροπολογίες μας καλόν είναι να υποβοηθήσουν την τελευταία ίσως μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλεται σήμερα να λυθεί το Κυπριακό. Γιατί στέκομαι πάνω στη φράση ότι οι τροπολογίες πρέπει να βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Η τροπολογία που υπάρχει που ζητά όλα τα μέρη να συμβάλλουν στην επίλυση του Κυπριακού μειώνει την πιθανότητα επίλυσης του Κυπριακού γιατί εξισώνει την δυνατότητα που έχει η Τουρκία να λύσει το Κυπριακό με την πολύ λιγότερη δυνατότητα που έχει η Ελλάδα, με την πολύ πολύ λιγότερη δυνατότητα που έχουν οι δύο πολιτικοί ηγέτες στην Κύπρο. Άρα το να παραμείνει η φράση ότι καλείται η Τουρκία να συμβάλλει μας δίνει όλους περισσότερη δύναμη προς την κατεύθυνση επίλυσης του Κυπριακού και περισσότερη δύναμη και στην κυρία Φλότ και στον κύριο Βανόρτε η αναφορά που λέει ότι πρέπει να αρθεί η απομόνωση των Τουρκοκυπρίων εμείς πρώτοι οι Ελληνοκύπροι και όλοι οι Κύπροι γιατί εγώ εδώ εκπροσωπώ και τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους η αναφορά αυτή πρώτα απ' όλα εμείς την αποζητούμε γιατί είναι Κύπροι οι συμπολίτες μας αλλά για να αρθεί η απομόνωση των Τουρκοκυπρίων πρέπει να αρθεί η κατοχή και η κατοχή έρεται με την επίλυση του Κυπριακού πρέπει η έννοια μας λοιπόν και η προσήλωσή μας να είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Κλείνω λέγοντας ότι εμείς θέλουμε το ψήφισμα αυτό να συμπεριλάβει αναφορά για τα συμπεράσματα του Δεκέμβρη και να συμπεριλάβει την θέση μας όπως ψηφίστηκε πέρσι για τους αγνοούμενους. δύο λεπτά. ευχαριστώ πολύ. Μερικές παρατηρήσεις ως προς το πρωτόκολλο της Άγκυρας. Θα πρέπει να πούμε ότι έχει προσδοριστεί μια συγκεκριμένη διαδικασία με μια σειρά και με προθεσμίες οι οποίες εξέπνευσαν στα τέλη του 2009. Δεν μπορούμε να αλλάζουμε αυτά τα πράγματα, δεν μπορεί να αλλάξουν αυτά που έχουν συμφωνηθεί. Έχουν προσδοριστεί ρητά και δεν μπορούμε να επανεφευρίσκουμε τίποτα. Υπάρχουν δεσμεύσεις που έχουν αναλυφθεί, έχει έρθει η ώρα να επιτελεστούν και τίποτε άλλο. Για τον κύριο Χόουιτ μια παράκληση δεύτερη, ως δεύτερη παρατήρηση, να ξανασκεφτεί λίγο τη στάση του. Δεν μπορούμε να έχουμε μια στρατηγική ε, διχασμένη, μια στρατηγική κατά την οποία μιλάμε στην Τουρκία με διαφορετικές φωνές, όπου έρχονται διαφορετικά αιτήματα, ε, που λέμε ναι αλλάξτε αυτό, κάντε εκείνο, ή αλλιώς μπορούμε να έχουμε μια γραμμή απλή, σαφή, ξεκάθαρη όπως της κυρία Σόμεν Ρόιτεν, η οποία προχωρεί και βοηθά στην όλη διαδικασία. Και πιστεύω ότι είναι προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κοινοβουλίου και της Τουρκίας να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή πλειοψηφία για την έκθεση χωρίς να διχαστούμε. για να μην δώσουμε την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον το Κοινοβούλιο, είναι διχασμένο, διαλυμένο και δεν έχει μία φωνή για να μιλήσει. Γι' αυτό και επιμένω για την υπαριθμόν 28 παράγραφο να μην επιμείνετε ως προς τις τροπολογίες σας. Είναι αυτή η πιο λογική προσέγγιση, είναι αυτή η οποία αποτεί και φόρο τιμής στην πολύ σοβαρή προσπάθεια της κυρίας Ομενρόιτεν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θέλω να αρχίσω κι εγώ με δίνοντας συγχαρητήρια στην εισηγήτρια για ένα όπως κάθε χρονιά εξαιρετικό και ισορροπημένο κείμενο. Θέλω να πω ότι οι συμβιβαστικές τροπολογίες είναι πολύ καλές και καταφέρνουν να ε, φέρουν κοντά αρκετά διαφορετικές απόψεις. Νομίζω ότι η έκθεση για την Τουρκία έρχεται σε πολύ κρίσιμη στιγμή και η προφορική τροπολογία της εισηγήτριας είναι και αυτή πάρα πάρα πολύ κομβική. Οι τελευταίες αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου για απαγόρευση λειτουργίας του Κουρδικού Κόμματος ΔΤΠ και η ακύρωση του νόμου που προέβλεπε την παραπομπή των στρατιωτικών σε πολιτικά δικαστήρια για ποινικά δικήματα αποδεικνύει ότι δεν έχει ακόμα εδρεωθεί ο έλεγχος της πολιτικής εξουσίας επί των στρατιωτικών. Η θέση της Τουρκίας είναι στην Ευρώπη όμως ο δρόμος που πρέπει να διανυθεί μέχρι την ένταξη είναι ακόμα μακρύς. Παρά τις υποσχέσεις, η Θεολογική Σχολή της Χάλκης παραμένει κλειστή, η χώρα διατηρεί ακέραιο το κάζους μπέλι εναντίον της Ελλάδας και οι παραβιάσεις συνεχίζονται στον ελληνικό εναέριο χώρο. Την ώρα που οι δυο πρωθυπουργοί συζητούν την επανέναρξη του διαλόγου Αθήνα-Άγκυρα, τέτοιε κινήσει στο Αιγαίο είναι απαράδεκτε και ανεπίτρεπτε γιατί σκοπός δεν είναι μόνο να ανοίγουν κεφάλαια ώστε να προχωράει η προσέγγιση Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος πρέπει να είναι η ουσιαστική τήρηση των υποχρεώσεων της Τουρκίας, ο εξευρωπαϊσμός και εκδημοκρατισμός της, που περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανάγκη η ίδια η Τουρκία. Ευχαριστώ. Ο κ. για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστώ και την κυρία Ομενρόιτεν ε, η οποία χρησιμοποιεί την ε, καλύτερη δυνατή επιμέλεια για να συντάξει το κείμενο αυτό. Θα ήθελα τώρα να απαντήσω στο αίτημα που μου έθεσε να, για να αποσύρω τις τροπολογίες ε, μου που αφορούν στην Κύπρο προκειμένου να καταστήσουμε πιο ισόρροπη την, ναι, το ισορροπητό το ψήφισμα. Όσο θυμάμαι, ε, σχετικά με το ψήφισμα του Υπουργείου Κοινοβουλίου πέρυσι στην Τουρκία, μπορέσαμε να καταλήξουμε σε ένα ιδιαίτερα ισορροπημένο κείμενο, το οποίο παρέμεινε και στο αρχικό κείμενο, αλλά με την τροπολογία υπαριθμών 10 που προτείνεται, νομίζω πως ξεφεύγουμε από, αυτό, το, από αυτή την ισορροπία που αρχικά είχε το σχέδιο ψηφίσματο, ειδικά σε ό,τι αφορά το ζήτημα του επικισμού της ε, νήσου ή την κατάσταση στην Αμόχωστο. Αυτό το θέμα αφορά στο πακέτο διαπραγμάτευσης ανάμεσα στις δύο κοινότητες. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να προσθεθούν τώρα στο κείμενο. Επίσης, ε, θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτό που είπε ο κύριος Βαν Όρντεν ότι δηλαδή σε αυτό είναι τη συμβαστική τροπολογία υπαρθμών 10 υπάρχει η προσπάθεια τήρησης ε, της ισορροπίας και να υπάρχει και σύσταση στο Συμβούλιο και στην Κομισιόν σχετικά με τις υποσχέσεις του 2004 και την τήρησή τους προκειμένου να πάψει ε, απομόνωση του βορείου τμήματος της Κύπρου από οικονομική σκοπιάς. Τονίζω λοιπόν ότι για να διατηρήσουμε ακριβώς αυτήν την ισορροπία χρειάζεται να λάβουμε υπόψη και αυτά τα στοιχεία και να δεχτούμε τουλάχιστον μία από τις τροπολογίες που αναφέρεται στην βούληση που πρέπει να εκφράσει το Κοινοβούλιο για την διακοπή της απομόνωσης του βορείου τμήματος της Νήσου. Ευχαριστώ. Η κυρία Κόρμ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Όμαν Ράιτεν για την έκθεση αυτή, γιατί είναι καλή ισορροπία που πέτυχε. Η συζήτηση για την Τουρκία, αντίθετα με τις υπόλοιπες ε, υποψήφιες χώρες, φαίνεται πάντα να μας ε, διαχωρίζει σε υπέρ και κατά. Άκουσα τι είπαν και οι άλλοι βουλευτές. Νομίζω ότι Όλοι συμφωνούμε για την ανάγκη μεταρρυθμίσεων στην Τουρκία και πάντα οι μεταρρυθμίσεις που επιθυμούμε είναι οι ίδιες. Αυτό που μας διχάζει είναι το σκέλος της ε, προοπτικής της προσχώρησης. Οι μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητα απαραίτητε δεν θα γίνουν αν δεν υπάρχει αυτή η προοπτική. Η κυρία Όμεν Ράιτεν είπε ότι εμεί ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να αποστείλουμε ένα σαφέ μήνυμα προ την Τουρκία. Σαφέ και ισχυρό. Νομίζω ότι στο πνεύμα αυτό η ιδεολογική σκέψη Α αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα. Η κυρία Όμεν Ράιτεν επέλεξε να πει ότι η διαδικασία είναι ανοιχτή. Η διαδικασία ποτέ δεν επρόκειτο να είναι ανοιχτή. Πάντα ως σκοπό είχε την προσχώρηση και νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε σαφείς προς την Τουρκία και τον τουρκικό λαό προς το συμφέρον και της Τουρκίας και των μεταρρυθμίσεων αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρία Γιαννάκου, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ την κυρία Όμεν ε, για την έκθεσή της γιατί δεν είναι απλώς μια ισορροπημένη έκθεση, αλλά είναι μια έκθεση αληθινή, είναι κοντά στην πραγματικότητα. Και αυτό είναι σημαντικό. Πέρα από επιθυμίες ή τη στάση που έχει ο καθένας μας για το θέμα της μελλοντική προοπτικής της Τουρκίας. Η Τουρκία είναι υποψήφια χώρα ε, και δεν μπορεί κανείς να της αρνηθεί το δικαίωμα να προσαρμόζεται στα κριτήρια της Κοπενχάγης και επομένως να γίνει κάποτε μέλος της Ένωσης και συμφωνώ και εγώ ότι δεν μπορούμε να περιπέζουμε την Τουρκία, αλλά και εκείνη θα πρέπει εφόσον έχει χαράξει ένα τέτοιο δρόμο, γιατί από αυτή εξαρτάται, να προσαρμοστεί σε όσα προβλέπονται για τις δημοκρατικές χώρες της Ευρώπης. Νομίζω ότι η κυρία Όμεν στην προσπάθειά της και στο αίτημά της να αποσύρουμε τις τροπολογίες προσπαθεί να κρατήσει μια έκθεση που δίνει πράγματι ένα μήνυμα σε μια χώρα η οποία είναι υποψήφια και είναι μια πάρα πολύ μεγάλη χώρα. Δεν είναι μια μικρή χώρα, είναι μια χώρα που θα επηρεάσει τα πράγματα στην Ευρώπη αν γίνει μέλος. Εγώ επίσης θέλω να την ευχαριστήσω γιατί με τη συμβαστική της τροπολογία για την 99 και 102 ε, ε, τροπολογία εκ των οποίων την 99 ε, έχω κάνει εγώ με τον κύριο Κουμουτσάκο αποδέχθηκε να επαναλάβει το ζήτημα που αφορά ε, στα δύο νησιά, στην Ήμβρο και στην Τέννο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κ. Μαυρονικόλα, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την κυρία Νόεν για την προσπάθεια την οποία κατέλαβε ούτως ώστε τουλάχιστον στα μέτρα των υπαρχουσών δυνατοτήτων να έχουμε σχετικά στα χέρια μας τελικά στα χέρια μας ένα σχετικά ισορροπημένο ψήφισμα για την Τουρκία. Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίηση μου για την εμφάνιση της αναφοράς για τον επικισμό για επικισμό μιλούμε και η αναφορά αυτή στο ψήφισμα δίνει τις πραγματικές διαστάσεις ενός τεράστιου και μεγάλου κινδύνου ο οποίος υπάρχει με την δημογραφική αλλαγή που επιχειρείται από την Τουρκία στην Κύπρο. Δεύτερο θέμα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι είναι καλά να λέμε ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να βοηθήσουν στη λύση του Κυπριακού η Τουρκία όμως αποτελεί την κατοχική δύναμη και την στρατιωτική παρουσία που εμποδίζει την επίλυση. Θα έλεγα ότι στις συνομιλίες για το Κυπριακό το μόνο το οποίο έχει συμβάλει η Τουρκία μέχρι αυτή τη στιγμή είναι στο να ζητά ανθρώπινα δικαιώματα για τους Τούρκους πολίτες εντός της Κύπρου και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πράγματα δηλαδή εντελώς απαράδεκτα που οδηγούν σε ομοιροποίηση της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από την προσπάθεια για λύση του κυπριακού προβλήματος. Και τρίτον, όταν μιλάει η Ευρωπαϊκή Ένωση για απομόνωση των τουρκοκυπρίων, ασφαλώς αντιλαμβάνεται ο κύριος λόγος της απομόνωσης είναι η παρουσία του τουρκικού κατοχικού στρατού. Από την πλευρά της δημοκρατίας έχουν γίνει ούκο λίγα. Μέχρι που 20.000 Τουρκοκύπριοι από τις 80.000 πληθυσμών να εργάζονται στα ελεύθερα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Ντάφ για λεπτά. Κύριε, ο κύριος Στέφαν Φούλε Ο κύριος μας είπε ότι θα πρέπει να αξιοπιστήσουμε, ότι πρέπει να, ε, αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία στη διαδικασία διαπραγματεύσεων με την Τουρκία και νομίζω ότι η τροπολογία υπαριθμών 28 ε, υποστηρίζει αυτή την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εγώ θα την υποστηρίξω. Νομίζω ότι καλό είναι να ελέγξουμε και την ατμόσφαιρα στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου για την Κύπρο. Να σας ζητήσω να δείξετε θετική στάση προς την τροπολογίες τροπολογία 164, η οποία αναφέρει την ανάγκη η Τουρκία να αποστείλει ένα κατάλληλο μήνυμα για την υποστήριξη των συνομιλιών Χριστόφια και Ταλάτ. Σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη χρονική στιγμή, ξεκινώντας την απόσυρση κάποιων στρατευμάτων. Σήμερα. Νομίζω ότι επειδή το εμπορικό σκέλος είναι προς το παρόν ε, φραγμένο, η Τουρκία μπορεί να συνδράμει στην επίλυση των προβλημάτων της νήσου. Αυτό δεν θεωρώ ότι αποτυπώνεται επαρκώς στην τροπολογία υπαριθμών, ε, τη συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 10. Ο κύριος Κασουλίδης, δύο λεπτά. Thank you, Chairman. in my turn, would like... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστώ τον κύριο Μανώλη. Και να πω ότι οι τροπολογίες, συμβαστικές τροπολογίες, όπως συμφωνεί, όπως προτάθηκαν, από την εισηγητρία και όπως εγκρίθηκαν από τους κοιόδης εισηγητές προσφέρουν μια πολύ λεπτή ισορροπία για ένα αποτέλεσμα το οποίο θα φέρει πιο κοντά στην ένταξη την Τουρκία. Όταν θα είναι έτοιμη δηλαδή να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα της δώσει μια θετική όθηση. Και αυτό πιστεύω πρέπει να είναι το μήνυμα το οποίο πρέπει να αποστείλει η Επιτροπή μας. Εξίσου σημαντικό είναι στο κυπριακό ζήτημα για το οποίο Ξέρουμε ότι τόσο πολύ εμποδίζει την πρόοδο της Τουρκίας στην ένταξη, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ως προς την διατύπωση και η διατύπωση της κυρίας Σόμεν είναι η καταλληλότερη πιστεύω. Δεν υπάρχει, πιστεύω, δεν γνωρίζω να υπάρχει αλλού τέτοια εξέλιξη ως προς, την κατακεφαλήν, το κατακεφαλήν εισόδημα, το οποίο έχει τριπλασιαστεί το τελευταίο καιρό, όπως έχει τριπλασιαστεί στην ε, Βόρεια Κύπρο ε, και ως εκ τούτου δεν θεωρώ ότι μπορεί να θεωρείται απομονωμένη περιοχή ή εις βάρος της σωτίας και εμπάργο. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να καταλάβει η Τουρκία ότι είναι προς το συμφέρον της και εάν θέλουμε να ανοίξουμε το ζήτημα αυτό προς τους πάντες δεν στέλνουμε θετικό μήνυμα στην Τουρκία. Όσοι λοιπόν υποστηρίξουν την ένταξη της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβουν υπόψη τους και αυτό το δεδομένο. Κυρία Θεοχάρου, δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η προσπάθεια της κυρίας Όμεν είναι εξαιρετική και η πρόταση ψηφίσματος χαρακτηρίστηκε ως πάρα πολύ καλή. Δηλαδή κύριε Πρόεδρε θα έχουμε ακόμη ένα εξαιρετικό ψήφισμα αλλά η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των Κυπρίων πολιτών στην Κύπρο θα εξακολουθήσει να συνεχίζεται αμύωτη και γι' αυτό το λόγο υπεύθυνη θα είναι η Τουρκία. Απόδειξη, το γεγονός ότι οι Ελληνοκύπριοι πρόσφυγες κερδίζουν συνεχώς δίκες εναντίον της Τουρκίας για παραβίαση των δικαιωμάτων του στα ευρωπαϊκά δικαστήρια με πρόσφατη την απόφαση του Βρετανικού εφετείου. Συνεπώς, όλοι όσοι μιλούν για την απομόνωση δήθεν του βορείου τμήματος της Κύπρου πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτό το τμήμα ανήκει στους Ελληνοκύπριους. Το ένα σημείο. Και το δεύτερο είναι αυτό που είπε ο κύριος Μαυρονικόλας, ότι υπεύθυνοι για την οποιαδήποτε απομόνωση, υπεύθυνο είναι ο στρατός κατοχής. Έχω αποσύρει τις δικές μου τροπολογίες για να διευκολύνω την κυρία Όμεν στην προσπάθειά της. Επισημένω όμως δύο σημεία. Ο όρος «settlement of Turkish citizens on the island» πρέπει να ερμηνεύεται οπωσδήποτε ως παράνομος επικισμός, που είναι έγκλημα πολέμου. Και δεύτερον, Όλοι υποστηρίζουμε την διαδικασία των συνομιλιών για την επίλυση του κυπριακού προβλήματο. Και κάποιοι συνάδελφοι ευρωβουλευτέ έχουν χαρακτηρίσει τι πρόσφατε προτάσει τη Τουρκία που υπευλήθησαν μέσω του κυρίου Ταλάτ ω επικοδομητικέ, ακόμη και ω ένα γενναίο βήμα. Όμω πρέπει να γνωρίζετε αυτέ τι προτάσει και περιλαμβάνουν απαράδεκτα στοιχεία όπω τη χωριστή κυριαρχία, δύο πηγέ εξουσία, δύο FIR, δύο κεντρικέ τράπεζε, και επιπλέον περιλαμβάνουν την απέτηση της Τουρκίας για τη μετατροπή των Τούρκων πολιτών σε Ευρωπαίους πολίτες μέσω Κύπρου, μέσω του οποιοδήποτε μορφώματος υπάρξει στην Κύπρο, πριν από την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά, καλής ποιότητας δουλειά σε αυτή την έκθεση. Χαίρομαι ειλικρινά για το επικοδομητικό πνεύμα που έχει υπάρξει, καθώς και για τους συμβιβασμούς που έχουν προταθεί. Γι' αυτό πιστεύω, όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, ότι δεν θα πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο την πολύ εύθραυστη και λεπτή ισορροπία που έχει επιτευχθεί αυτή τη στιγμή στο κείμενο. Δεν σας κρύβω όμως ότι προσωπικά θα επιθυμούσα να είναι πιο ισχυρή, ακόμα πιο καθαρή η αναφορά στην συνεχιζόμενη επικίνδυνη μαζική στρατιωτική δραστηριότητα της Τουρκίας στο Ανατολικό Αιγαίο. Με υπερπτήσεις, δηλαδή με πτήσεις πάνω από έδαφος ελληνικών νησιών, κατοικημένων ελληνικών νησιών, που προξενούν εύλογη ανησυχία, προβληματισμό, φόβο πολλές φορές ότι θα μπορέσει αυτό να οδηγήσει σε ένταση και κρίση στο Αιγαίο. Πρόσφατα, κύριε Πρόεδρε, πολύ πρόσφατα, στον τουρκικό τύπο υπήρξε μια αποκάλυψη ότι την περίοδο 2002 και 2003 το τουρκικό γενικό επιτελείο σχεδίαζε να υπάρξει θερμή κρίση τόσο στο Ανατολικό Αιγαίο όσο και στη Θράκη για εσωτερικούς λόγους εσωτερικής τουρκικής πολιτικής. Αυτά τα δημοσιεύματα δυστυχώς δεν, ε, δεν τα αρνήθηκαν με κατηγορηματικό τρόπο Τούρκοι στρατηγοί. Αυτό τι δείχνει ότι η δραστηριότητα, η συνεχιζόμενη της Τουρκίας στο Ανατολικό Αιγαίο μπορεί πολλές φορές να γίνει εργαλείο για άλλες επιδιώξεις, εργαλείο για να υπάρξει κρίση και ένταση. Κάτι που η Ελλάδα και πιστεύω ότι όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες της περιοχής καθόλου δεν θέλουν. Γι' αυτό θα ήθελα να είναι πιο έντονη αναφορά. Αλλά από εκεί και πέρα πιστεύουμε και θα στηρίξουμε το συμβασμό που έχει επιτευχθεί. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Δόκτωρας Φλιόρη. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επειδή έχω μόνο δύο λεπτά, θα είμαι πάρα πολύ σύντομο για τα συγκεκριμένα θέματα που θίγει η έκθεση της κυρίας Ράιτεν. Καταρχάς, ε, η έκκληση για να γίνει ε, εκταμένη μελέτη για το πρόγραμμα GAP στο Ανατολικά. Όπως είπαμε και πέρσι, θεωρούμε ότι δεν είμαστε σε θέση να διεξάγουμε τέτοια μελέτη. Και οι λόγοι είναι καταρχάς το πεδίο εφαρμογής μιας τέτοιας μελέτης, γιατί το πρόγραμμα GAP περιλαμβάνει θέματα άρδρευσης, παραγωγής, γεωργίας, δοσοκομείας, ε, ε, υγείας, εκπαίδευσης, καλύπτει 9 περιφέρειες, μεγάλη έκτηση, 22 ε, φράγματα, πάρα πολλά προγράμματα και πάρα πολλές, πολύ μεγάλη επιφάνεια. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν όλα αυτά ε, υπερβαίνουν το πεδίο μιας μελέτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ξεπερνάει και τις πόρους αλλά και την εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν έχουμε κοινωνική βάση. Για τη δεύτερη έκκληση, για την αξιολόγηση των προγραμμάτων των πρωτοεξιακών και των σχετικών ε, μέσων. Θα ήθελα να πω ότι προβλέπονται εξπόστε αναλύσεις από το 2011 για όλα τα πρωταξιακά μέσα συμπεριλαμβανομένου του ΦΑΡ και τα αποτελέσματα, τα πορίσματα θα προκύψουν στα τέλη του 2011. Θα διτεθούν και θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τέλος, για το θέμα που θίγεται στην τροπολογία περίθμων 28, ξέρετε ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαστε, υποστηρίζουμε τη γλώσσα της Συμφωνίας ε, Διαπραγματευτικής Πλαισίου θεωρούμε ότι αποτελεί τον καλύτερο συμβιβασμό που υπάρχει στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαδικασία αυτή. Ευχαριστώ. Φιλόρι, Ευχαριστούμε κύριε Φιλόρι. Η κυρία Χόμεν για τα τελικά σχόλια. Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τα λόγια τα επενετικά που απέφθηναν για την ε, έκθεση αλλά και για τους συμβιβασμούς λίγο πολύ. Να ξαναξεκινήσω λέγοντας το εξής. Για το θέμα το Κυπριακό. Αυτό που έκανα για το Κυπριακό και ζήτησα ειδικά από τον Ρίτσαρ Χάουαρτ να το εξετάσει, ζήτησα να πετύχουμε έναν συμβιβασμό ο οποίος θα κάλυπτε όλες τις τροπολογίες για το Κυπριακό. Και αυτό συμφωνήσαμε. Για παράδειγμα, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Δεν θελήσαμε να ψηφίσουμε την 170, την ε, τροπολογία του Σφόμποντα, γιατί πήγαινε πολύ παραπέρα από τη δική, σου, τη δική σας τροπολογία, την 157. Σήμερα λοιπόν τον ερχόμαστε να ψηφίσουμε απόψεις που περιλαμβάνονται, θεωρώ, στο συμβαστική τροπολογία, αυτό θα ήταν κάτι που δεν το επιθυμούσα. Αυτό αφενός. Και αυτό είπα και στον κύριο Φανόρδεν Με ακούτε κύριε Φανόρδεν Κύριε Φανόρδεν δεν σας ε, ικανοποίησε η συμβαστική τροπολογία για το Κυπριακό, αλλά σας καλέσαμε στις συναντήσεις. Δεν σας είδα να έρχεστε ένα το κρατούμενο. Κατά δεύτερον, ασκείται κριτική για κάποιες από τις τροπολογίε, για την αμόχωστο για παράδειγμα. Αλλά ένα από τους συναδέλφους σα μου ζήτησε να τη συμπεριλάβω. Δεν είναι μόνο οι δικοί σα συνάδελφοι από τους Βρετανούς συντηρητικού, αλλά και οι συνάδελφοι σοσιαλιστές και οι συνάδελφοι τη δική μου ομάδα. Δεν τη βρήκα εγώ την τροπολογία. Θέλω όμω να πετύχω ένα συμβιβασμό. Ε, πώς θα γίνει, θα πρέπει να συμπεριλάβω την ε, συνένεση που επικρατεί. Και κύριε Φανόρντεν, δεν μπορώ να συμπεριλάβω τα πάντα, γιατί θα πρέπει να πείσω και τα μέλη της ομάδας μου από την Κύπρο και την Ελλάδα να μην απορρίψουν την τροπολογία αυτή, γιατί για κάποια θέματα πήγαιναν παραπέρα από ό,τι αναφέρεται στο συμβιβασμό. Τι κάνουμε λοιπόν, εξετάζουμε πώς μπορούμε, πώς μπορεί ο κάθε εισηγητής να πετύχει μία ευρεία συνένεση για κάποιες διτυπώσεις, για πολύ δύσκολα θέματα, για το θέμα της Κύπρου για παράδειγμα και ελπίζω και από πλευρά σοσιαλιστών να αποσύρουν την ψηφοφορία των επιπλέον τροπολογίων. Κατά δεύτερον, για την αιτιολογική σκέψη Α. Να πω στη Μαρέικε το, το εξή. Η Μαρέικη Κορνέλη είναι ακόμα στην αίθουσα. Α, έφυγε. Αυτό που θα ήθελα να τη απαντήσω είναι το εξή. Το κείμενο του ιδεολογικής σκέψη Α αποτελεί μια συμφωνία που έγινε πριν από δύο χρόνια για την προσχώρηση. Αυτό επιθυμούσαμε. Κατά δεύτερον, στο κείμενο αυτό μπορούμε, για το κείμενο αυτό μπορούμε να πετύχουμε ευρεία συνένεση στο Κοινοβούλιο. Άρα ξανασκεφτείτε το. Στόχος μας δεν θα πρέπει να είναι να βάλουμε το δικό μας ε, συνέστημα, αλλά το να στείλουμε ένα θετικό και ισχυρό μήνυμα προς την Τουρκία. Αυτός είναι ο δικός μου στόχος και αυτός θα έπρεπε να είναι και δικός σας στόχος για τους σοσιαλιστές, για την προφορική τροπολογία τώρα που έγινε από τη συνάδελφο Φλότρ. Φαίνεται ότι η κυρία Φλότρ δεν ε, ικανοποιήθηκε από τη δική μου προφορική τροπολογία. Τι θέλει λοιπόν. Αυτό που επιθυμεί δεν μου φαίνεται πολύ σκόπιμο, γιατί τι θέλει να πετύχει με την προφορική της τροπολογία, να επανεισάγει η κυβέρνηση την νομοθεσία για τα, δικαστικ... τα στρατιωτικά δικαστήρια στο κοινοβούλιο. Δεν είναι το κοινοβούλιο όμως το πρόβλημα, το συνταγματικό δικαστήριο είναι το πρόβλημα. Αυτό που λέω λοιπόν στην τροπολογία μου ότι δεν έχει νόημα γιατί το κοινοβούλιο υπερψήφισε την απόφαση αυτή. Δεν νομίζω ότι είναι σκόπιμη αυτή η προφορική τροπολογία της ε, κυρίας Φλότρου. Αν γνωρίζει κανείς την κατάσταση πρέπει να ζητήσει συνταγματική εννοθεώρηση και αυτό ζητάω στην τροπολογία. Συνάδελφοι λοιπόν, επαναλαμβάνω, αυτό που προσπάθησα να κάνω είναι να αποτυπώσω στις συμβιβαστικέ το ευρύ φάσμα των απόψεων που επικρατεί στο Κοινοβούλιο. Αν θέλουμε να μην υπάρχουν ασάφειες στο μήνυμα που θα αποστείλουμε, σας παρακαλώ να υποστηρίξουμε τους συμβιβασμού που πετύχαμε και που πετύχαμε και πριν από αρκετό χρόνο με τη βοήθεια των αξιότιμων συναδέλφων. Σκεφτείτε το σήμερα το βράδυ και ξέρετε ότι θα ήθελα να αποσύρετε οτιδήποτε δεν συμπεριλαμβάνεται στο κατάλογο ψηφοφοριών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια. Σε ποιο άρθρο του κανονισμού θέλετε να αναφερθείτε κύριε Χαουίτ. Δεν θέλω να, δεν θέλω να παρατηρήσω τη συζήτηση και να πω ότι ξέρω ότι ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Σας δω εσάς πρόεδρε να κοιτάξετε την γραπτή έκθεση που έχουμε μετά από μία συνάντηση συμβιβαστική να ελέγξετε ότι η 170 του Χανεσφόποντα συμπεριλήφθηκε στις τροπολογίες αυτές και η 152 και η 22 και 23 δεν συμπεριλήφθησαν. Δεν είναι το θέμα πιανού η άποψη θα συμπεριληφθεί, αλλά θα ήθελα να το επιβεβαιώσει αυτό η γραμματεία και να το επιβεβαιώσετε κι εσείς, γιατί ε, φαίνεται ξεκάθαρα από το γραπτό κείμενο της ημέρας εκείνης. Φάτελο però bilateralmente perché non può essere una... Ε, εντάξει, θα το επαληθεύσουμε. Θα το ελέγξει η γραμματεία. Ωραία. Μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διατάξεως, Βανόρντεν. Διαδικαστικό. Επί Του κανονισμού, ε, διαδικαστικό, Πρόεδρε για τον τρόπο με τον οποίο ε, χειριζόμαστε τις συμβαστικές τροπολογίες. Δεν ε, μπορεί η Επιτροπή μας να διατηρήσει να χρησιμοποιεί ένα σύστημα όπου μια συμβαστική τροπολογία ισχυρίζεται ότι έχει καλύψει και απορροφήσει τροπολογίες των βουλευτών και ως εκ τούτου τις θέτει εκτός καταλόγου, τις διαγράφει από τον κατάλογο ψηφοφοριών. Γιατί αυτό συμβαίνει. Εάν δεν λαμβάνετε υπόψη μια συγκεκριμένη τροπολογία, δεν μπορείτε να ισχυριστείτε ότι την έχετε συμπεριλάβει στην συμβαστική πρόταση. Και πρέπει να γίνει χωριστά η ψηφοφορία αυτών των τροπολογιών που δεν καλύπτονται από το συμβασμό. Ξέρω ότι και άλλοι συνάδελφοι έχουν θέσει το ζήτημα αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει για μένα τον ίδιο μιλάω μόνο. Οι 140, οι 169 και οι 175 τροπολογίες μου δεν έχουν καλυφθεί από τη συμβαστική και θα πρέπει να ψηφιστούν χωριστά. Και κατά τη διάρκεια της συζητήσεως άκουσα και άλλους συναδέλφους να αναφέρουν τις δικές τους τροπολογίες σε αντιστοιχή κατάσταση. Εντάξει. Καταλαβαίνω το ότι το ζήτημα είναι ευαίσθητο και θα το σκεφτούμε. Τώρα, συμβαστικές τροπολογίες οδηγούν στο να καταπέσουν οι τροπολογίες οι οποίες συμπεριλαμβάνονται. Τώρα, αν εσείς αμφισβητείτε το ότι η συμβαστική τροπολογία δεν συμπεριλαμβάνει, δεν εμπεριέχει τις θέσεις σας. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να αποφασίσει ο Προεδρείο σε συνεργασία με τον ε, συγγητή. Όλα καλά, αλλά ξέρετε πως ε, κάποιος πρέπει το τέλος να αποφασίσει. Κύριε Μενρόιτεν, Ρόιτεν, κύριε Πρόεδρε, είμαι πολλά χρόνια σε αυτό το σώμα και μια συμβαστική τροπολογία καλύπτει μια συγκεκριμένη πολιτική. Και αν υπάρχει συμφωνία αναφορικά με το περιεχόμενο του κειμένου, τότε οι τροπολογίες οι υπόλοιπες καταπίπτουν. Τελεία και παύλα. Διότι το περιεχόμενο Ε, του κειμένου από το οποίο έχουμε συμφωνήσει ενδεχομένως να διαφέρει από το αρχικό κείμενο από την τροπολογία και σίγουρα διαφέρει διότι πολύ από τους συναδέλφους σας έχουν εντελώς διαφορετικά κείμενα για την Κύπρο. Μιλάω για τους συντηρητικούς συναδέλφους σας. Τώρα, αν αυτό το συμβαστικό κείμενο γίνει δεκτό, τότε αυτομάτως ό,τι αντιβαίνει στο συμβασμό καταπίπτει. Δεν χρειάζεται να δοθούν περαιτέρω εξηγήσει, Πρόεδρε. Και στο κείμενο αναφέρεται ότι ψηφίζεται μόνο εάν καταπέσει η συμβαστική τροπολογία, κύριε Βανόρδεν. Τι το κακό, τι το στραβό υπάρχει εδώ. Δεν έχει νόημα αυτό που λέτε. Πρόεδρε, μου ετέθη ένα ερώτημα, μπορώ να απαντήσω. Φυσικά θα μπορούσαμε πάντα να λέμε τυχαία ή ε, όποια τυχαία τροπολογία ότι έχει καλυφθεί από μια συμβαστική και από αυτόν τον τρόπο αντιβγάζουμε από τη συμφορία. Ο κάθε βουλευτή έχει το δικαίωμα να υποβάλει τροπολογία και ο ίδιο θα πρέπει να αποφασίζει αν θεωρεί ότι καλύπτεται από τη συμβαστική η τροπολογία του ή όχι. Και αν θεωρεί ότι δεν καλύπτεται, δεν μπορείτε εσεί να ισχυρίζεστε ότι καταπίπτει λόγο ή χάρη τη συμβαστική. Ο πρόεδρος ναι, μπορούμε να πούμε πως καταπίπτει μια τροπολογία ε, που δεν καλύπτεται εφόσον δεν είναι συμβάτη. Εν αυτή η ζήτηση ενδιαφέρουσα μεν, αλλά εκτός τόπου και χρόνου δε. Πρέπει να περάσουμε στο επόμενο σημείο της διατάξεως. Τώρα, εάν υπάρχουν κάποιες ε, διαφορές, εκκρεμότητες αναφορικά με τη συμβατότητα ή την ε, συμπερίληψη τροπολογιών στην ε, συνδυαστική τροπολογία, αυτό θα πρέπει να το αποφασίσουμε σε υπευθυνότητα του εισηγητή και του, και του Προεδρείου. Λοιπόν, περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο, ασφάλεια του εφοδιασμού σε φυσικό αέριο. Το λόγο έχει ο εισηγητής κύριος Σάιρους Βόλσκι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να επιστήσω την προσοχή σας στην γνωμοδότηση για την ασφάλεια της ε, προμήθειας αερίου, του υποδιασμού σε φυσικό αέριο. Είναι γνωμοδότηση για την Επιτροπή Ήτρε 22 Τροπολογίε υπέβαλε η, ε, η Επιτροπή ΑΦΕΤ και εγώ υπέβαλα κάποιες και προσπάθησα να συμπεριλάβω την προτάση των συναδέλφων. Να πω ότι ο κανονισμό αυτός για τον εφοδιασμό σε φυσικό αερίο είναι κρίσιμος για τι πρακτικές εφαρμογές και για το άρθρο 176α της Συνδίκης Λισαβόνας σε ό,τι αφορά την αλληλεγγύη σε καταστάσεις ενεργειακής κρίσης. Η γνωμοδότηση αυτή έχει καταρτιστεί βάσει της έκθεσής μου του 2007 για την πολιτική εξωτερικής πολιτικής, την, οποία και υποστήριξε πλειοψηφικά το Κοινοβούλιο και καμία... Συγγνώμη κύριε Σάρους Βόλσκι, παρακαλώ συνάδελφοι, αν έχετε να πείτε το οτιδήποτε, εκτός εθούς παρακαλώ. Η συνεδρία συνεχίζεται. Παρακαλώ, μπορώ να έχω την προσοχή σας. Εξέλθετε τις αιθούσεις και αφήστε μας να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Αλλά δεν με ακούτε. Παρακαλώ, αν υπάρχει κάποιος κλητήρας ε, μπορεί να επέμβει και να απομακρύνει τους συναδέλφους. Παρακαλώ, εγκαταλείψτε την αίθουσα. Να πω λοιπόν ότι η γνωμοδότηση αυτή συνάδει με την έκθεση του 2007 του Κοινοβουλίου μας. Οι πιο πολλές τροπολογίες που έχουν υποβληθεί ήταν επικοδομητικές και σας ευχαριστώ και αποτελούν ε, ένα σημαντικό συμπλήρωμα στο σχέδιο το παρόν. Ιδιαίτερα οι προτάσει του κυρίου Μπρόκ που περιλαμβάνονται στι συμβαστικέ 3 και 11, τη κυρία Βασέσκου για το άρθρο 1, του κυρίου Σβόμποντα για την παράγραφο που προσθέτω στην ε, συμβιβαστική 2 και 11 για τις κυρίες Ομονράιτεν, του κυρίου Λαντσμπέργκης, του κυρίου Κοβάτσεφ, που διευκρινίζουν τις τροπολογίες 9 και 21. Όλα αυτά συμπεριλήφθησαν στις 11 συμβιβαστικές τροπολογίες στην πρώτη συμβαστική τροπολογία συμπεριέλαβα τι προτάσει τη κυρία κυρίας Μπασέσκου, στην δεύτερη τη κυρία Όμον Ράιτον και του κυρίου Σβόμποντα, στην τρία τι προτάσει του κυρίου Μπρόκ, στην τέσσερα του κυρίου Κόβατσεφ, στην πέντε τη κυρία Μπασέσκου, στην έξι του κυρίου Μπρόκ, στην επτά του κυρίου Κόβατσεφ. στην οκτώ του κυρίου Πρέντα, στη συμβαστική παριθμόν εννέα της κυρίας Ρίρα στην 10 του κυρίου Λαντσπέρκης και στην 11 του κυρίου Σβόποτα, Λαντσπέρκης και Σβόποτα. Οι προτάσεις λοιπόν αυτές ήταν πολύ πολύτιμες. Προσπάθησα να τις συμπεριλάβω για να ενισχύσω το κείμενο και μία σειρά τροπολογιών η οποία κατέφθασα σε χτες, Δευτέρα. Πολύ καθυστερημένα και δεν μπόρεσα να τις λάβω υπόψη. Την ευχαριστώ βέβαια. Αλλά θεωρώ ότι περιορίζουν τις φιλοδοξίες της γνωμοδότησης αυτής. Και επικαλούνται χωρίς λόγο ήδη ισχύουσες ε, νομοθεσίες και θα ήθελα να παραμείνουμε στο κείμενο ως έχει που αντικατοπτρίζει την έκθεση του 2007 που υπερψηφίστηκε. Αυτά είχα να σας παρουσιάσω, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βαν Μπάλεν έχει το λόγο. Με δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όλοι θυμούνται τη μεγάλη κρίση του φυσικού αερίου που έπληξε την Ανατολική Ευρώπη, επηρέασε τη σταθερότητα των ανατολικών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ολόκληρη της Ένωσης και είναι απαραίτητο να ε, αποτρέψουμε για το μέλλον τέτοιο ενδεχόμενο. Αν δείτε λοιπόν και την πρόταση και τη γνωμοδότηση, όπως και τις συμβαστικές λύσεις που έχουν εξασφαλιστεί, έχουμε σαν σύνολο ένα πολύ, δυνατό, ένα πολύ ισχυρό συνδυασμό των εθνικών ευθυνών και των ευθυνών και υποχρεώσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς λοιπόν ως Άλντε θα υπερψηφίσουμε χρησιμοποιήσουμε ε, τις συμβαστικές τροπολογίες που εξασφαλίζουν μια πολύ ισχυρή τοποθέτηση. Σημάνς και δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, ο Σιώδης ηγητής θα ήθελα να πω πως ε, η υπάρχουσα γνωμοδότηση έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πρέπει να την ε, υιοθετήσουμε, πρέπει να υιοθετήσουμε αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης. δεν πρέπει να λησμονούμε ότι προκύπτει ε, ως αποτέλεσμα μιας πολύ δύσκολης κατάστασης η έκθεση αυτή. Ο ύπατος εκπρόσωπος και η Επιτροπή ε, πρέπει να έχουν έναν σαφή ρόλο σε περιπτώσεις τέτοιων κρίσεων και χρειαζόμαστε και σαφείς ρήτρε που να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κατάσταση στα, στις σχέσεις μας, τα ενεργειακά θέματα στις σχέσεις μας με τα τρίτα κράτη. Χωρίς διευκρίνηση αυτών των στοιχείων θα είναι πολύ ισχνός αυτός ο κανονισμός δεν θα ε, αρθεί στο ύψο των προσδοκιών και των απαιτήσεων σε τελευταία ανάλυση και της συνθήκης Λισαβόνας. Γι' αυτό θα ήθελα να υποστηρίξω την πρόταση του κ. Σάριου Βόλσκη. La parola alla collega Riera Madurei. Η κυρία Ριέρα Μαντουρέ έχει το λόγο. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να επενθυμίσω πως είναι η πρώτη φορά που μιλάμε για την έκθεση αυτή στην Επιτροπή. Θα ήθελα να πω λοιπόν κάποια πράγματα παραπάνω και να εξηγήσω την θέση της ομάδας μου. Εν πάση δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες, οι οποίες είναι πολλές και συμφωνούμε με τον εισηγητή. Θα ανασχοληθώ με τα θέματα με τα οποία διαφωνεί η ομάδα μου σε σχέση με τον εισηγητή. Είναι δύο πρώτα απ' όλα ο ρόλος του συντονισμού που θα έχει ο ύπαρος εκπρόσωπος και το ζήτημα της ρήτρας της τρίτης χώρας. Ε, γιατί λέμε ότι δεν συμφωνούμε με τον συντονιστικό ρόλο που ανατίθεται στον ύπατο ε, εκπρόσωπο. Πρώτα απ' όλα, διότι ο στόχος μας είναι να υπάρξει μια εσωτερική αγορά και η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, μιλάει με μια φωνή. Δεν έχει νόημα λοιπόν να υπάρχει ο Επίτροπος που θα είναι υπεύθυνο για το ιστορικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει εκπρόσωπο για το εξωτερικό. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν μια ενεργειακή πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να παραμείνουν εντό του κοινοτικού πλαισίου όλα αυτά. Επίση, η συνθήκη τη Αβώνα δεν δίνει αρμοδιότητε ε, στην ύπατο εκπρόσωπο για αυτά τα ζητήματα. Και να υπενθυμίζω πω ε, όταν είχαμε τελευταία κρίση μεταξύ Ρουσία και Ουκρανία, η επίλυση σε αυτήν την κατεπίγουσα κατάσταση πέρασε όπω και περνά πάντα από τη λήψη δημοκρατι... διπλωματικών μέτρων αλλά και την ε, επίλυση των διαφωνιών αυτών ανάμεσα στις ενδιαφερόμενες χώρες. Για τέλος να αναφερθώ στην ε, ρήτρα της τρίτης χώρας. Το Κοινοβούλιο υποστήριξε την ρήτρα της τρίτης χώρας, καρδιά και των διαπραγματεύσεων του τρίτου πακέτου στην ιστορική αγορά, βασικά ως ένα μέσο το οποίο οδηγούσε στην προστασία των ε, κοινωτικών ε, συμφερόντων. Θα ήθελα να υπενθυμίσω πως ε, τα κράτη που εξαρτώνται από το ρωσικό αέριο ε, είναι τα άμεσα εμπλεκόμενα και θα πρέπει να ξεχνάμε ότι μερικές φορές μετατράπει η στάση μας, η στάση ορισμένων κρατών ως επίδεση απέναντι στην Ρωσία. Χρειάζεται λοιπόν οι επιχειρήσεις που λειτουργούν και προμηθεύουν αυτό το αέριο να τηρούν μια ενιαία στάση Προστατεύοντα προστατεύοντας τα συμφέροντα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου λοιπόν καταλαβαίνετε πως ε, αιτιολόγησα ήδη το θέμα. Παρακαλώ, λέει ο Πρόεδρος, ε, έχετε εξαντλήσει κατά πολύ το χρόνο μιλία σας. Μισό δευτερόλεπτο Πρόεδρε, να αναφερθώ στην ε, τροπολογία μου που έλαβε χθε ο εισηγητή, όπω δήλωσε. Δεν πρόκειται για μια καινούργια τροπολογία, είναι απλά μια σύνθεση κάποιων τροπολογιών και προτείναμε να ε, ληφθεί υπόψη ω συμβαστική τροπολογία. Εμεί όμω θα καταψηφίσουμε την πρότασή του σε αυτό το ζήτημα. κύριο Μπρόκ για δύο λεπτά. Πρόεδρε, θα είμαι σύντομο. Θα ήθελα εξ του ΕΛΚ να πω ότι Υποστηρίζουμε την έκθεση του Σαρισβόλσκη και τις συμβαστικές τροπολογίες και νομίζω ότι είναι ισορροπημένο το αποτέλεσμα. Βλέπουμε ότι αναφέρεται για παράδειγμα το Συμβούλιο της Ενέργειας όπου η κυρία Κλίντον είναι υπεύθυνη ε, από αμερικανικής πλευράς και από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. Νομίζω ότι υπάρχει εδώ μία αντίθεση προς την κινητική μέθοδο την οποία σαφώς υποστηρίζουμε και θα πρέπει να ενισχυθεί όπως είπε και η προηγούμενη ομιλήτρια. Γιατί θα πρέπει να ενισχυθεί η αρχή της πλειοψηφίας. Bene. La parola conclusiva al το λόγο έχει ο συγητής Άιρος Βόλτ για τα τελικά σχόλια. Ευχαριστώ. Ε, σύμφωνα με τα όσα άκουσα από τις ομάδες, ε, κατάλαβα ότι υπάρχει μια γενικευμένη υποστήριξη και νομοδότησης ε, με μια εξαίρεση τροπολογία 63 από πλευρά σοσιαλιστών. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω για αυτή την υποστήριξή σας, να πω κάτι για την 63 να τη σχολιάσω το μήνυμα ειδικά με το ποιος ε, θα είναι υπεύθυνο για το να μιλάει η Ευρώπη με μία φωνή. Είμαι αντιπρόεδρος της ε, Κομισιόν, κάθετος, ύπατος εκπρόσωπος, ε, σε στενή συνεργασία με τους κατέχοντες τα αντίστοιχα χαρτοφυλάκια. Λοιπόν, αυτό ακριβώς αναφέρεται και σε έκθεση η οποία έγινε δεκτή το 2007. Και μιλάει για την κοινοτικοποίηση της πολιτικής και ήταν ε, πεποίθηση της Επιτρεπής μας ότι ήταν ένα ζήτημα εξωτερικής πολιτικής και όχι ε, θέμα ενεργειακό μόνο. Αυτό έγινε αποδεκτό από το Σώμα συμπεριλαμβανομένης και της Επιτροπής Ήτρε. Και σε ό,τι αφορά την ε, ρήτρα τρίτης χώρας, αυτό δεν ε, περιέχεται στην σχετική οδηγία, αλλά υπάρχει το θέμα της ροής των χρηματοδοτήσεων και πόσο αυτό είναι ε, σύμφωνο με την κοινωτική νομοθεσία. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο θα πρέπει να διαφωνήσουμε. Παραμένει η διαφωνία μας επί της τροπολογίας 63, αλλά θα περάσουμε αύριο στις ψηφοφορίες. Ολοκληρώσαμε την ημέρα διάταξη. Διακόπτουμε τη συνεδρίαση. Θα συνεχίσουμε τώρα με το διευρυμένο Προεδρείο της Επιτροπής μας. Παρακαλώ